Καλησπέρα σας. Συνεχίζεται λοιπόν η συνεδρίασή μα και με πάρα πολύ μεγάλη χαρά καλωσορίζω στην ε, Επιτροπή μας, την Επιτροπή Αλίας, ε, τον ε, Κύπριο Υπουργό Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, κύριο Σοφοκλή Αλετράρη, ασκούντα την Προεδρία του Συμβουλίου. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που συναντιόμαστε. Άλλε δύο φορέ ε, και σήμερα γευματίσαμε μαζί, αλλά και στο Στρασβούργο είχαμε συνεδριάσει. Άρα δεν είναι η πρώτη φορά που γνωριζόμαστε, που τον βλέπω. Αλλά η επίσκεψη αυτή πραγματικά εντάσσεται σε μια παράδοση που έχουμε, όπου κάθε Προεδρία ε, παρουσιάσει τις προτεραιότητες για το εξάμεινό της επιτροπές. Αλλά είναι και κάτι περισσότερο είναι η δυνατότητα που έχουμε να ανταλλάξουμε απόψεις. Είναι ένα σημείο συνάντησης, στην προκειμένη περίπτωση με την Κυπριακή Προεδρία, Μπορούμε λοιπόν ε, να σχολιάσουμε διάφορα πράγματα και κάποιες φορές ε, ξέρουμε ότι το Κοινοβούλιο δεν αντιμετωπίζεται από το Συμβούλιο ακριβώς όπως θα έπρεπε δυνάμει των συνθήκων. Πάντως πρέπει να γνωρίζετε ότι το Κοινοβούλιο έχει διάθεση να συνεργαστεί με το Συμβούλιο. Η Κύπρος είναι μια μικρή μεν χώρα αλλά και πολύ μεγάλη. Έχει έξι μήνες μπροστά της η Κύπρος, έχει καθήκοντα να δεκπεραιώσει που μπορούν να είναι σημαντικά. Είναι πολλά τα θέματα που εκκρεμούν, ο Υπουργός το γνωρίζει άλλωστε, δεν θα τα επαναλάβω. Θα προτιμούσα ο ίδιος να μας ε, αναφέρει τις προτεραιότητές του και έπειτα οι συντονιστές και οι λοιποί βουλευτές της Επιτροπής μας θα μπορούσαν να, να εκφράσουν τις δικές τους απόψεις που φαντάζομαι είναι γνωστές και στον Υπουργό. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι είναι μια πολύ σημαντική χρονική στιγμή για το Κοινοβούλιο αλλά και για το Συμβούλιο, διότι έχουμε επιτάπητος ε, το θέμα της μεταρρύθμισης. Πολλά ζητήματα είναι ανοιχτά που πρέπει να τα ρυθμίσουμε. Υπάρχει μια μακρά διαμάχη ό,τι αφορά τα σχέδια διαχείρισης η θέση του Συμβουλίου ε, είναι ε, σημαντικά αποκλίνουσα σε σχέση με τη θέση του Κοινοβουλίου και η Κυπριακή Προεδρία και ο αρμόδιος υπουργός στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να βοηθήσει να απεμπλακούν τα πράγματα, αν αυτό είναι δυνατό, μεταξύ άλλων διότι το έχουμε πει επανειλημμένως και φυσικά δεν καμία συνιστά απειλή αυτό, αλλά ε, προειδοποίηση ίσως ναι. Υπό την έννοια ότι εάν δεν απεμπλακούν τα πράγματα ε, σε ό,τι αφορά τα σχέδια διαχείρισης, όλοι μας, και επαναλαμβάνω όλοι μας, ε, διατρέχουμε τον κίνδυνο να παραμείνει στα λόγια η όλη η μεταρρύθμιση, να στερείται ουδήποτε νοήματος. Εάν έχουν εμπλοκή με τα σχέδια διαχείρισης, δεν έχει και νόημα να συνεχιστεί η μεταρρύθμιση. Εγώ ελπίζω να μην ε, επιβεβαιωθώ. Ε, ελπίζω πραγματικά να μπορέσουμε να δώσουμε σάρκα και οστά, να μην μείνει κενό γράμμα. Και νομίζω είμαστε ομόφωνοι όλοι στο Κοινοβούλιο. Αυτό που περιμένουμε από το Συμβούλιο είναι να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και όχι να κοιτάζει από την άλλη πλευρά και να παραμείνουν τα πράγματα ως έχουν, να παραμείνει αυτό το αδιέξοδο. Υπάρχουν και πολλά άλλα θέματα όμως. Έχουμε τις συμφωνίες που αποτελούν και αυτές ένα σημαντικό κομμάτι των εξωτερικών πτυχών της κοινή αλληλευτικής πολιτικής και έχουμε και πολλά άλλα ζητήματα που φαντάζομαι ότι θα ανακύψουν και σήμερα στη διάρκεια των παρεμβάσεων. Εδώ όμως ε, θα σταματήσω να μιλώ εγώ και θα δώσω το λόγο στον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, τον κύριο Υπουργό, επαναλαμβάνοντας πόσο χαιρόμαστε που τον έχουμε σήμερα μαζί μας και εγώ προσωπικά Χαίρομαι γιατί υπάρχει βούληση, ε, την ε, αποδεικνύει ο Υπουργό, ε, να έρχεται σε επαφή με το Κοινοβούλιο. Γι' αυτό και είμαι πεπισμένο ότι θα είναι άκρο αποδοτική οι έξι αυτοί μήνε. Ιδίω ό,τι αφορά τι σχέσει γενικότερα των δύο οργάνων, αλλά και ό,τι αφορά τι διαπροσωπικέ μα επαφέ. Κύριε Υπουργέ, σα δίνω το λόγο, αλλά προτού σα δώσω το λόγο να πω ότι θα γίνει ως εξή η διαδικασία. Θα μιλήσει ο κύριος Υπουργός, έχει στη διάθεσή του όσο χρόνο θέλει, ε, μία μέρα, δύο μέρες, έξι μήνες έχουμε στη θέση μα. Αλλά βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, είναι περιορισμένος ο χρόνο ε, τη ε, Επιτροπής μας Άρα μπορείτε να μιλήσετε εσείς κύριε Υπουργέ, για 20-25 λεπτά. Εν συνεχεία θα δώσω το λόγο στους συντονιστέ και εν συνεχεία σε οποιονδήποτε άλλο βουλευτή θελήσει το λόγο. Και στο τέλο θα απαντήσει ο κύριο Υπουργό στα ερωτήματα, σχόλια. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ σήμερα για να παρουσιάσω στην Επιτροπή σας το πρόγραμμα εργασίας μας με την ευκαιρία που η Κυπριακή Δημοκρατία αλλά αναβάνει για πρώτη φορά στην ιστορία της την Προεδρία του Συμβουλίου. Η ανάληψη της ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χώρα μου είναι μια ιστορική στιγμή την οποία προσμέναμε καθώς και μεγάλη πρόκληση και τεράστια ευθύνη που αναλαμβάνουμε με προθυμία αλλά και σοβαρότητα. Μέρος αυτής της πρόκλησης για εμένα ως Προέδρου του Συμβουλίου είναι η συνεργασία μαζί σας ως συνομοθετικό όργανο και πάντοτε μέσα στο πνεύμα της συνθήκης της Λισαβόνας προκειμένου να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στον τομέα της αλληλείας για τους πολίτες μας. Οι Ευρωπαίοι πολίτες περιμένουν από εμάς να ηγηθούμε, να καθοδηγήσουμε και να συνδιαμορφώσουμε σημαντικές πολιτικές όπως η μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής αλλά και πιο βραχυπρόθεσμα σχετικά ζητήματα που αφορούν την διαβίωση των συνανθρώπων μας και ασχολούνται στον τομέα της αλίας. Προσδοκώ σε μια πολύ συνεργασία, στενή συνεργασία μαζί σας, καθώς έχουμε μπροστά μας ένα βαρύ και σημαντικό νομοθετικό πρόγραμμα. Η ίδια συνεργασία θα υπάρχει και σε επίπεδο τεχνοκρατών. Πριν περάσουμε στις λεπτομέρειες του προγράμματος της Προεδρίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την προκάτοχό μου κυρία Μέτε Κέσκοφ, Υπουργό Τροφίμων Γεωργίας και Αλίας της Δανίας, για την εξαιρετική δουλειά της και την επιτυχία της να καταλήξει σε μια γενική προσέγγιση σχετικά με το βασικό κανονισμό της κοινή αλευτικής πολιτικής και την κοινή οργάνωση αγοράς. Τα παραπάνω υπήρξαν αρκετά σημαντικά επιτεύγματα, ενώ ταυτόχρονα κατάφερε κατά την Προεδρία της να πετύχει συμφωνία μαζί σας στα ζητήματα σχετικά με τα μέτρα εμπορικών κυρώσεων και της τροποποίησης του σχεδίου αποκατάστασης του ερυθρού τόνου. Τώρα όσο αφορά τις προτεραιότητες, έχουμε χωρίσει τις προτεραιότητές μας σε δύο σκέλη. Το πρώτο αφορά την επίτευξη πρόοδου στη δέσμη μεταρρυθμίσεων της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Το δεύτερο, δεδομένου ότι βρισκόμαστε στο δεύτερο εξάμεινο, αφορά την έγκριση 10 προτάσεων ως το τέλος του έτους, μεταξύ των οποίων η πρόταση για τα τεχνικά μέτρα και πρόταση για το καθεστώς πρόσβασης των 12 ναυτικών μιλίων. Όσον αφορά τη δέσμη μεταρρύθμισης της κοινή αλληλευτικής πολιτικής, ως κύρια προτεραιότητά μας έχουμε θέσει την επίτευξη μιας μερικής γενικής προσέγγισης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας στο Συμβούλιο του Οκτωβρίου. Σε γενικές γραμμές, οι Υπουργοί είναι αρκετά ικανοποιημένοι από το προτινόμενο γενικό επίπεδο χρηματοδότησης, παρόλο που ορισμένοι θα προτιμούσαν περισσότερη ελαστικότητα όσον αφορά τις μεταφορές μεταξύ των κεφαλαίων του προϋπολογισμού. Ορισμένοι επίσης θα ήθελαν να δουν αύξηση των πόρων για τα μέτρα ελέγχου και εφαρμογής και για τη συλλογή δεδομένων. Από τις ως σήμερα συζητήσεις των Υπουργών εξάγεται το συμπέρασμα ότι επιθυμούν ένα πιο ενεργό ρόλο για το Ταμείο. Πιο συγκεκριμένα θα επιθυμούσαν να δουν τη συνέχιση και επαναφορά ορισμένων μέτρων για την αναδιάρθρωση του στόλου ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην υδατοκαλλιέργεια, τη θέσπιση περισσότερων μέτρων για τη μεταποίηση και εμπορία, τη μεταφορά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την αλία και απορρέουν από το πρόγραμμα Φύση 2000 και την οδηγία πλαίσιο σχετικά με τη στρατηγική για τη θάλασσα την απλούστευση των διοικητικών κανόνων και διαδικασιών. Σας διαβεβαιώνω ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια με ένα πνεύμα συναντήληψης ώστε να υπάρχει σύγκληση απόψεων σε όλα τα εκκρεμή θέματα. Εφόσον οι Υπουργοί κρίνουν ότι υπάρχει ανάγκη περαιτέρω συζήτησης προς ανατολισμού, αυτή θα διεξαχθεί το Σεπτέμβριο. Όσον αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία της μεταρρύθμισης, είμαστε πρόθυμοι να πραγματοποιήσουμε μαζί σας άτυπες προκατακτικές επαφές σχετικά με τον βασικό κανονισμό τόσο πριν όσο και μετά τη ψηφοφορία στην Επιτροπή σας. Όπως μας έχετε ενημερώσει, και το σεβόμαστε πλήρως κύριε Πρόεδρε η πρακτική είναι τέτοια ώστε δεν αναμένεται να επιτευχθεί συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Ωστόσο, θεωρούμε ότι ο συνεχιζόμενος διάλογος μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων της νομοθετικής εξουσίας δεν μπορεί παρά να οδηγήσει μεσοπρόθεσμα στην εξέβρεση λύσης. Όσον αφορά την κοινή οργάνωση αγοράς, προσδοκούμε την έναρξη άτυπων επαφών μαζί σας εντός του τρέχοντος μηνός, εφόσον έχετε ήδη υιοθετήσει τη θέση σας εντός της Επιτροπής. Ήδη φαίνεται ότι υπάρχουν συγκλήσεις σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων των οργανώσεων των παραγωγών στην, πρόθεση της βιώσιμης διαχείρισης περιλαμβανομένης της επιλεξιμότητας των εργαλείων και του χειρισμού των ανεπιθύμητων αλλιευμάτων που πρέπει να εκφορτωθούν μετά την έναρξη ισχύω της απαγόρευσης των απορρίψεων και την πρόσκληση προς την Επιτροπή για υποβολή πρότασης θέσπισης ελάχιστων προτύπων για την οικολογική επισήμανση αλλιευτικών προϊόντων συμπεριλαμβανομένων και των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. Με ενθαρρύνει το γεγονός ότι η πολιτική μας γραμμή συγκλίνει στο ότι τα αλλιεύματα που δεν καλύπτουν τις προδιαγραφές εμπορίας πρέπει σε κάθε περίπτωση να εκφορτώνονται για παραγωγή ηχθιαλεύρων και ηχθιελαίων και όχι για ανθρώπινη κατανάλωση. Δεν κρίνονται σκόπιμες σημαντικές αλλαγές στην πρόταση της Επιτροπής για την απλούστευση των παρεμβάσεων. Ασφαλώς, κύριε Πρόεδρε, δεν συμφωνούμε σε όλα. Για παράδειγμα, εσείς προκρίνετε την πρόβλεψη περισσότερων υποχρεωτικών πληροφοριών για τους καταναλωτές από ό,τι εμείς. Αυτά τα ζητήματα μπορούμε να τα εξετάσουμε περαιτέρω προκειμένου το κάθε μέρος να κατανοήσει καλύτερα τη θέση του άλλου. Τώρα αναφορικά με τις προτάσεις για τις οποίες πρέπει κύριε Πρόεδρε να επιτευχθεί συμφωνία ως το τέλος του έτους. Όπως καλά γνωρίζετε, το Συμβούλιο αφιερώνει μεγάλο μέρος του χρόνου του το δεύτερο εξάμεινο στην προετοιμασία και λήψη απόφασης σχετικά με τα συνολικά επιτρεπόμενα αλλιεύματα, τα tax, και τις ποσοστώσεις για το επόμενο έτος. Αυτή τη χρονιά πρέπει να λάβουμε έξι τέτοιες αποφάσεις. Ως πρώτο βήμα την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί στο Συμβούλιο ανταλλαγή απόψεων επί της ανακοίνωσης της Επιτροπής διαβούλευση για τις αλλιευτικές δυνατότητες κατά το 2013. Ένα από τα σημαντικά ζητήματα για το οποίο θα κληθούμε να λάβουμε απόφαση το προσεχή φθινόπωρο είναι τα τάξη για τα οποία υπάρχει ενδεικτική επιστημονική γνωμοδότηση που βασίζεται σε ολοκληρωμένα στοιχεία. Πρόκειται για μια νέα και ευπρόσδεκτη εξέλιξη σε σχέση με πέρσι και ως εκ τούτου ανυπομονώ να ακούσω τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών και το πώς οι Υπουργοί αντιμετωπίζουν το θέμα αυτό. Στην ανακοίνωση βρίσκονται ορισμένα καλά νέα. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πλέον ποια είναι η μέγιστη βιώσιμη απόδοση MSY σε όρους θνησιμότητας λόγω αλίας για το 80% των αλλιευμάτων που αφορούν 38 αποθέματα για περισσότερα από τα μισά των συγκεκριμένων αποθεμάτων αλλιεύομαι σε επίπεδα μέγιστης βιώσιμης απόδοσης από τώρα, δηλαδή τρία χρόνια νωρίτερα από τον στόχο που τέθηκε στο Johannesburg. Σκοπεύω να στηριχτώ στην ενθαρρυντική αυτή πορεία και στη σκληρή προσπάθεια που κατέβαλαν οι προκατόχοι μου για να υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα οι τέσσερις βασικές αρχές που καθορίζουν τις επιλογές μας σχετικά με τα ΤΑΚ είναι ακόλουθες. Η πρώτη αρχή αφορά τη συνέχιση των μακροπρόθεσμων διαχειριστικών σχεδίων όπου αυτά υφίστανται. Δεύτερη αρχή είναι ότι τασόμαστε υπέρ της βιώσιμης αλίας και της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης και ως εκ τούτου επιθυμούμε όσο το δυνατό μεγαλύτερη πρόοδο σε αυτά τα ζητήματα. Για αυτό το σκοπό επιδιώκουμε να φτάσουμε κατευθείαν στην MSY, όπου αυτό συνεπάγεται αύξηση των ΤΑΚ. Αρχή μας, κύριε Πρόεδρε, έντιμα μέλη της Επιτροπής, είναι το επάγγελμα του Ευρωπαίου Αλιέα πρέπει να είναι βιώσιμο και αξιοπρεπές. Επομένως, είμαστε ευαίσθητοι σε κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα. Η τελευταία αρχή είναι να είμαστε ουσιαστικοί και παραγωγικοί κατά τη διαδικασία καθορισμού των ΤΑΚ. Σε αυτούς τους δύσκολους οικονομικά καιρούς είναι δύσκολο να δικαιολογήσουμε την δαπάνη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ προκειμένου εμείς να ψάχνουμε επί δύο ολόκληρες μέρες και νύχτες λύση για τα ταχ του Δεκεμβρίου. Ακόμα και αν η σύνοδος του Δεκεμβρίου έχει καταλήξει παραδοσιακά να είναι μαραθώνια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης ή ότι δεν θα καταβάλουμε όσο το δυνατό μεγαλύτερη προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τα ΤΑΚ. Τον Ιούλιο, το Γάβρο, μετά την αυριανή έκδοση της επιστημονικής γνωμοδότησης. Τον Οκτώβριο, ΤΑΚ Βαλτικής και Ειδών Βαθαίων Υδάτων. Τον Νοέμβριο, ΤΑΚ της Μαύρης Θάλασσας και το Δεκέμβριο εσωτερικά και εξωτερικά ΤΑΚ. Ως το τέλος του έτους πρέπει να υιοθετήσουμε άλλες δύο νομοθετικές πράξεις και προς τούτο υπολογίζουμε στη δική σας στενή συνεργασία. Η πρώτη αφορά την παράταση του καθεστώτος πρόσβασης στα 12 ναυτικά μίλια για άλλα δύο έτη ως το τέλος του 2014. Αυτό θα μας δώσει χρόνο να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις για τη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Το Συμβούλιο μπορεί να συμφωνήσει με αυτή την πρόταση και ελπίζω ότι το ίδιο μπορείτε να κάνετε και εσείς. Αναμένω με την ψηφοφορία σας επί του θέματος στη σύνοδο της Επιτροπής σας τον Οκτώβριο. Η δεύτερη αφορά μετατροπή σε μόνιμα μια σειράς μεταβατικών τεχνικών μέτρων τα οποία ισχύουν από την περίοδο της Σουηδικής Προεδρίας στα τέλη του 2009. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση χρόνου στους ώμους των συνομοθετών. Ακόμα δεν έχουμε πάρει θέση σχετικά με την πρόταση αφού μόλις τη λάβαμε. Ωστόσο, η Προεδρία γνωρίζοντας τις ευθύνες της θέτει ως στόχο την έγκριση και έκδοση της πρότασης ως το τέλος του έτους το υπολογίζουμε στη στήριξή σας. Αναφορικά με τις άλλες προτάσεις και συγκεκριμένα με τα μακροπρόθεσμα σχέδια διαχείρισης θεωρούμε ότι είναι ένα από τα δυσκολότερα πεδία της συνεργασίας μας μου προκαλεί πραγματικά λύπη κύριε Πρόεδρε έντιμα μέλη της Επιτροπής να βλέπω το πιο επιτυχημένο μέσο της κοινή αλληλευτικής πολιτικής να πλήττεται λόγω διαφορετικών προσεγγίσεων στο θέμα των κανόνων ελέγχου της αλίευσης μετά την έναρξη ισχύω της συνθήκης της Λισαβόνας. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να σημειωθεί πρόοδος για τους φακέλους που εκκρεμούν. Θα μελετήσουμε τη θέση σας για το σχέδιο διαχείρισης του Σολομού της Βαλτικής θάλασσας, το οποίο τέθηκε προς ψηφοφορία στην τρέχουσα σύνοδο της Επιτροπής σας. Πρόκειται για ένα σημαντικό σχέδιο για τη Βαλτική, ιδίως αν λάβουμε υπόψη την δύσκολη κατάσταση του αποθέματος. Όσον αφορά το Σαφρίδι, χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία σας να πραγματοποιήσετε σχετική ακρόαση τον προηγούμενο μήνα. Αυτή επέτρεψε στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους ενδιαφερόμενους φορείς να εκφράσουν τις θέσεις τους και να διεξαχθεί μια παραγωγική συζήτηση για το θέμα αυτό. Σχετικά με το συγκεκριμένο σχέδιο, οι θέσεις του Συμβουλίου είναι γνωστές, καθώς έχουν εκφραστεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Όπως έχω δηλώσει, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, θα επιδιώξουμε να συνεργαστούμε μαζί σας για να σημειώσουμε πρόοδο πάνω στο θέμα. Το ίδιο ισχύει όσον αφορά την ευθυγράμμιση των προτάσεων στο πλαίσιο και στο πνεύμα της συνθήκης της Λισαβόνας. Με αυτό το δεδομένο μελετούμε τη θέση σας επί της πρότασης ευθυγράμμισης των τεχνικών μέτρων στη Μεσόγειο. Η μελέτη βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο. Απομένει να δούμε εάν οι αντίστοιχες θέσεις μας επί των άρθρων μπορούν να ευθυγραμμιστούν με τις δικές σας. Είμαστε πρόθυμοι να εξετάσουμε μαζί τρόπους επίτευξης συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση εάν αυτό είναι δυνατό. Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε καλό παράδειγμα της μεταξύ μας συνεργασίας και θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για μια μεσογειακή χώρα όπως είναι η δική μου. Όσον αφορά την αλλιευτική προσπάθεια στην ανοιχτή θάλασσα και την αλλιευτική προσπάθεια για τον μπακαλιάρο και αφαίρεση των θεριγίων των καρχαριών, υπάρχουν αυτές οι τρεις προτάσεις σχετικά με τις οποίες θα θέλαμε να σημειώσουμε πρόοδο. Η πρώτη αφορά την αλλιευτική προσπάθεια στην ανοιχτή θάλασσα. Η πρόταση αναμένεται να παρουσιαστεί στη Σύνοδο του Συμβουλίου το Σεπτέμβριο και οι Υπουργοί θα έχουν την δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά. Το ζήτημα αυτό σχετίζεται με την φιλοσοφία των ΤΑΚ, επομένως η ανταλλαγή απόψεων θα παίξει σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων για τα ΤΑΚ των ειδών βαθαίων υδάτων τον Οκτώβριο. Ανυπομονούμε να ακούσουμε τις απόψεις σας επί του θέματος, αν και το πιθανότερο είναι ότι το ζήτημα θα απασχολήσει περισσότερο την Ιρλανδική Προεδρία. Το ίδιο ισχύει και για την αναθεώρηση του καθεστώτος αλληλευτικής προσπάθειας στο σχέδιο του Μπακχαλιάρου, για το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να υποβάλει τροποποίηση στις αρχές του φθινοπόρου. Δεν μπορώ να προβώ σε σχόλια πριν δω την πρόταση, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Συνεπώς, θα προβούμε σε ανταλλαγή απόψεων κατά το Συμβούλιο του Νοεμβρίου. Η αλλιευτική προσπάθεια για τον Πακαλιάρο αναμένεται να βρίσκεται στο επίκεντρο του Συμβουλίου για τα ΤΑΚ και τις ποσοστώσεις το Δεκέμβριο, όπως ακριβώς και πέρσι. Η τρίτη πρόταση επί της οποίας αναμένουμε τις απόψεις σας με μεγάλο ενδιαφέρον αφορά την αφαίρεση των πτενιγίων των καρχαριών. Όπως γνωρίζετε, το Συμβούλιο στη γενική προσέγγιση του στήριξε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο ελκύει την προσοχή της κοινή γνώμης. Ο κόσμος προδεύει, εικόνες καρχαριών με πτυρίχια που κόβονται και η απάνθρωπη απόρριψη των σφαγίων προκαλούν έντονες αντιδράσεις ακόμα και κατακραυγή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να φαίνεται ότι στηρίζει ή συμμερίζεται με κανένα τρόπο τέτοιες πρακτικές. Αναμένουμε τις απόψεις σας και ελπίζουμε ότι μπορούμε να υπολογίζουμε στη συνεργασία σας ώστε η πρόταση να υιοθετηθεί ως το τέλος του έτους. Αναφορικά με τα εξωτερικά ζητήματα, είναι γνωστό ότι το φθινόπωρο είναι η εποχή που οι αξιωματούχοι μας γυρίζουν όλη την Ευρώπη και τον κόσμο επιδιώκοντας συμφωνίες για τα αποθέματα που δεν έχουν διαβατήριο και ταξιδεύουν στις θάλασσες έτσι όπως ορίζει η φύση. Πρώτον, έχουμε το διαμάντι του στέματος, της Μάρε Νόστρουμ, τον ερυθρό τόνο πρέπει να αποφασίσουμε σχετικά με τη νέα εντολή εν ώψη της φετινής συνόδου της ICAT. Ευελπιστώ ότι η διαδικασία θα είναι λιγότερο αγχωτική από ό,τι πριν από δύο χρόνια, αν και κανείς δεν μπορεί να είναι ποτέ σίγουρος. Για το σκοπό αυτό, στο Συμβούλιο του Οκτωβρίου, οι Υπουργοί θα προβούν σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη σύνοδο της ICAT. Στο μενού του Οκτωβρίου περιλαμβάνεται επίσης ρέγκα χωρίς βίζα, παπαλίνα Σέγγεν και αρτικό μπακαλιάρο στα πλαίσια της ετήσιας διαβούλευσής μας με την Ορβηγία, όπου θα ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με τα αποθέματα που τελούν υποκοινή διαχείριση στη Βόρεια Θάλασσα και την ετήσια ανταλλαγή αλλιευτικών δυνατοτήτων. Όσον αφορά τις συμφωνίες αλλιευτικής σύμπραξης, αναμένουμε τη συγκατάθεσή σας για το νέο πρωτόκολλο με τη Γρυλανδία, για το οποίο θα σας αποστείλουμε έτοιμα εντός του ερχόμενου μήνα, μετά την υπογραφή του νέου πρωτοκόλλου. Σχετικά με την Μαυριτανία, παρά τις εντατικές διαβουλεύσεις και ενώ βρισκόμαστε λιγότερο από ένα μήνα πρώτης λήξη του πρωτοκόλλου, δυστυχώς δεν φαίνεται να υπάρχει καλή προοπτική για συμφωνία. Σας διαβεβαιώνω ότι θα αφιερώσουμε όσο χρόνο και προσπάθεια χρειάζεται για εξάντληση όλων των περιθωρίων για κατάληξη στο θέμα. Σχετικά με το Μαρόκο, είναι ακόμα πολύ νωρίς, επομένως πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σχετικά με την Ουινέα Μπισάου πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πολιτική κατάσταση. Κύριε Πρόεδρε, η χώρα μου είναι μια δημοκρατία με μακρά ιστορία και αρχαίο πολιτισμό βαθιά ριζωμένο στη Μεσόγειο. Η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου αποτελεί μια νέα πρόκληση για μας, ιδίως όταν τίθονται τόσα πολλά ζητήματα επιτάπητος και οι προσδοκίες για πραγματική αλλαγή στην κοινή αλλιευτική πολιτική όλων μας είναι τόσο μεγάλες. Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας στα πλαίσια μιας εταιρικής σχέσης προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να παραδώσουμε ένα καλύτερο μέλος στους αλληλείς μας, στις αλληλευτικές μας κοινότητες, στους καταναλωτές και στις θάλασσές μας. Θα καταλήξω, κύριε Πρόεδρε, έντιμα μέλη της Επιτροπής, λέγοντας το εξής. Για μένα δεν υπάρχουν προεδρίες για μικρές και μεγάλες χώρες. Υπάρχουν προεδρίες επιτυχημένες και μη. Και θα κάνουμε το παν δυνατό ώστε η δική μας προεδρία να είναι επιτυχημένη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και θα χαρώ να δεχτώ τις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν τον πρώτο γύρο των ερωταπαντήσεων με τους συντονιστές που έως παρακαλώ να διατυπώσουν μία ερώτηση. Ο κύριος Αντινόρο είναι ο πρώτος ομιλητής από το ΕΛΚ, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να σας καλωσορίσουμε κύριε Υπουργέ να σας ε, καλωσορίσουμε και να συγχαρούμε ιδίω για τα καθήκοντα να λαμβάνετε αυτό το εξάμεινο. Ε, να ξεκινήσω από το τελευταίο. Είπατε δεν υπάρχουν μικρές και μεγάλες χώρες. Υπάρχουν προεδρίες που τα καταφέρνουν, που έχουν επιτυχία και άλλες που τα καταφέρνουν. Ε, μάλιστα, είχατε πει λίγο νωρίτερα κάτι άλλο. Είπατε ότι η Κύπρος είναι μια μικρή χώρα, αλλά μπορεί να ασκήσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Συμφωνώ. Σε ό,τι μας αφορά, Θέλω να πω ότι περιμένουμε πολλά από την Προεδρία σας. Είπατε ε, πολλές φορές, ε, αναφερθήκατε στην Μεσόγειο, στο Μάρε Νόστρομ, ξέρετε, εγώ ως Ιταλός, Σικελός, με ικανοποιεί ιδιαίτερα αυτή η αναφορά και ως εκπροσωπός του ΕΛΚ. Στον μακρύ κατάλογο που μας παρουσιάσατε, και μας καταστήσετε κοινωνού σχετικά με όλα σας τα σημαντικά ραντεβού και όλα τα σημαντικά θέματα που θα έχετε να αντιμετωπίσετε στο Συμβούλιο. Θα ήθελα να προσθέσω, αν επιτρέπετε, ε, κάτι παραπάνω. Αν μπορώ να σας προτείνω κάτι. Βεβαίως φαντάζομαι ότι ήδη η ατζέντα σας είναι γεμάτη από υποχρεώσεις και οι έξι μήνες δεν αρκούν. Όμως, ξέρετε, μιλήστε για τη Μεσόγειο. Εμείς ξέρουμε ότι έχουμε σε εφαρμογή την ακρονισμό του 2010 που θεωρητικά μπορεί να αναθεωρηθεί μετά την έγκριση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Όμως και θεωρητικά και πρακτικά ο κείμενος κανονισμός προβλέπει ότι μετά από δύο χρόνια θέσεως σε ισχύ υπάρχει ανάγκη για monitoring, για παρακολούθηση, για να δούμε πρακτικά αν λειτουργεί ή όχι. Λοιπόν, λέω ότι πέρασαν αυτά τα δύο έτη μόλις τώρα και ε, φρονώ ότι η επανεξέταση αυτού του κανονισμού είναι προς το συμφέρον όλων αν περιμένουμε να μπει σε ισχύ η νέα κοινή αλληλευτική πολιτική και η περιφερειοποίηση ε, που θα συμπεριλαμβάνεται λοιπόν στην κοινή αλληλευτική πολιτική, αυτός ο κανονισμός για τη Μεσόγειο καλό θα ήταν ταυτόχρονα να αρχίσει να εξετάσετε. Αν μου επιτρέπετε λοιπόν αυτή την πρόταση. Κάτι άλλο τώρα που μας και με αφορά Θυμάμαι ότι όλοι οι προεδρεύοντες του Συμβουλίου τα τελευταία χρόνια ε, αντιμετωπίζουν το ζήτημα των χωρικών υδάτων. Ξέρετε, εμεί στην Ιταλία, φαντάζομαι και εσείς στη δική σα χώρα, στη δική σας χώρα, ίσω πιο πολύ από άλλε χώρε, το θέμα των ε, χωρικών υδάτων είναι σημαντικό. Εμεί δεν έχουμε καθορίσει ε, πολυμερό ε, τα χωρικά υδάτα, τουλάχιστον μονομερό τα έχουμε ορίσει. Πρέπει να υπάρξει όμω ένα κοινό κανόνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θεωρώ ότι η Λέδη Άστον που μα εκπροσωπεί σε εξωτερικέ υποθέσει. Πιστεύω ότι δεν θα κάνει κάτι αν δεν κινητοποιηθεί από εσά το Συμβούλιο. Πιστεύω ότι κάποιο πρέπει να κάνει μια απαρχή για να βρει μια λύση. Σήμερα μόνο προβλήματα έχουμε εμεί ω Ιταλοί, εγώ ω Σικελό, βλέπω ότι συνεχώ μα παραβιάζουν τα χωρικά ύδατα. Ε, έχουμε συνεχώ ε, ε, ε, σκαφών που εισέρχονται παρανόμω στα χωρικά ύδατα. Και θέλω ότι αυτό το πρόβλημα δεν είναι μόνο ιταλικό, Θέλω να πω λοιπόν ότι αν θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι μόνο η οικονομική ένωση αλλά και πολιτική, αν μου επιτρέπετε να σα προτείνω κάτι, μήπω θα θέλετε να θέσετε και αυτό το θέμα στο τραπέζι που θα απασχολεί θα του προετοιμασμού. Σα ευχαριστώ. Καλή δουλειά και καλώ ήρθατε στι Βρυξέλλε. Σίγουρα πιστεύω ότι θα έχουμε μια αγαστή συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε πολύ κυρία Αντινόρα. Κυρία Ρόντουστ. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, Χαίρομαι ιδιαίτερος που σας βλέπω σήμερα εδώ. Είχαμε και άλλες ε, ευκαιρίες για συνομιλία μαζί σας. Θα πρέπει να εκφράσω το σεβασμό μου προς το πρόσωπό σας, διότι έχω την ε, αίσθηση ότι πράγματι καταβάλατε μεγάλη προσπάθεια για να είστε παρόν εδώ στο Κοινοβούλιο. Είχατε έρθει μάλιστα και πολύ πριν να ξεκινήσει η Κυπριακή Προεδρία. Με εντυπωσίασε λοιπόν η διάθεση σας για συνεργασία και ότι είμαι πολύ αισιόδοξη την περαιτέρω συνεργασία μας και τους καρπούς της. Θα ήθελα λοιπόν πολύ σύντομα να αναφερθώ στα σημαντικά κατεμέ ζητήματα του βασικού κανονισμού και θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας γιατί αυτά που μέχρι στιγμής έχω ακούσει από πλευράς του Συμβουλίου δεν με πείθουν. Το MSY λοιπόν, η μεγίστη βιώσιμη απόδοση που συμφωνήθηκε το 2002 στο Johannesburg με την συμπλήρωση όπου δυνατόν. Νομίζω ότι τα κράτη, οι χώρε είχαν αρκετό χρόνο στη θέση του για να κάνουν τι σχετικέ προσαρμογέ. Και αν λένε ότι το 2012 είναι ακόμα δύσκολο, να, αν λένε το 2012 ότι είναι ακόμα δύσκολο να ε, περιοριστούν ε, στο MSY, νομίζω ότι δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι. Ερωτώ λοιπόν τι είδου δεδομένα έχετε και μπορείτε να μας διαθέσετε τα στατιστικά δεδομένα γιατί δεν ε, βλέπουμε καλή, ε, καλές επιδόσεις από το Συμβούλιο για, το, για τα ΤΑΚ. Νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε ότι επί έξι χρόνια έχουμε πει στους αλείς ότι έχουν στη διαθεσή τους την ε, δυνατότητα με τα να πάνε στην τράπεζα να βρούνε τα δάνεια που χρειάζονται και να οργανωθούν όπως πρέπει. Μπορείτε λοιπόν, ότι, μπορείτε, λοιπόν να μας πείτε ε, τη γνώμη σας για το θέμα αυτό, για την απαγόρευση της, ε, των απορρίψεων Εμείς ως ομάδα θεωρούμε ότι πρέπει να ισχύσει και πρέπει να δοθούν αρκετά κονδύλια στους αλληλείς ώστε να μπορέσουν να κάνουν τις τροποποιήσεις στους μηχανισμούς ε, των σκαφών τους έτσι ώστε να λειτουργήσει το σύστημα της απαγόρευσης ε, των απορρίψεων αποτελεσματικά. Και επίσης θέλω να ρωτήσω για την ε, περί για την υπερβολική δυνατότητα, capacity, τι έχετε υπόψη σας, τι συζητήσεις ε, μπορείτε να περιμένετε ότι θα αναπτυχθούν για τον περιορισμό αυτής της ε, ε, υπερβολικής δυνατότητας αλίευσης. Ερωτώ λοιπόν καθώς και από ενώσεις των αλλιέων και από τα συνδικάτα βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη αδημονία για πρόοδο στην υπόθεση αυτή και θα ήθελα να μας πείτε τις ε, δικές σας θέσεις. Αυτά λοιπόν επιγραμματικά, αλλά πιστεύω ότι αν μπορέσουμε τα πέντε αυτά σημεία, τα πέντε αυτά θέματα να τα επεξεργαστούμε και να προχωρήσουμε αποτελεσματικά θα έχουμε επιτύχει πάρα πολλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Ρόντιστο, κύριος Γκάλαχερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ, όπως οι συνάδελφοι, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, να ε, καλωσορίσω τον Προεδρεύοντα, τον ε, Υπουργό, στην Επιτροπή μας. Είχα την ευκαιρία, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά, όπως είπα, να συναντηθούμε μαζί του και στο Στρασβούργο. Είχα μάλιστα και εγώ μια σύντομη συζήτηση μαζί του. Έχει μακροσκελέστατο πρόγραμμα, πληρέστατο πρόγραμμα που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 2012, πριν το τέλος του έτους δηλαδή. Και εμείς βεβαίως θέλουμε να βοηθήσουμε, να συμπράξουμε στο βαθμό που μπορούμε για επιτυχή ε, υλοποίηση αυτού του προγράμματος, αυτού του θεματολογίου, διότι ξέρετε ότι αν δεν ολοκληρωθούν ορισμένα από τα μέτρα μέχρι τα τέλη του Δεκεμβρίου του 2012, μπορεί να έχουμε σημαντικές επιπτώσεις σε ορισμένα θέματα. Και δεν θέλω να πω κύριε Πρόεδρε ότι το θέμα δεν είναι να έρθει η Επιτροπή εδώ και να περιμένει να ε, παραδοθούμε ανεφόρων για δεύτερη φορά, γιατί ήδη μας είχαν προβλέψει κάποιες εξελίξεις ήδη από το Σεπτέμβριο πέρυσι και φαίνεται ότι μέχρι το 2013 ε, περιμένουν ότι θα έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές, αλλά πρέπει αρχές αυτές να αρχίσουν να υλοποιούνται, πρέπει να είναι αλλαγές ρεαλιστικές, πρέπει να είναι αλλαγές σε επαφή με την πραγματικότητα και όχι Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να συνεργαστούμε και σας διαβεβαιώ ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να σας βοηθήσουμε μέχρι το τέλος του χρόνου να μην βρεθείτε σε ε, δύσκολη θέση. Για το θέμα του ορίου των 12 μιλίων ξέρουμε βεβαίως ότι ίσως να μην αποφασίσει το Κοινοβούλιο να το εφαρμόσει αυτό, να μην το υλοποιήσει, αλλά είναι μια άλλη ιστορία. Για, τον, ε, για το μακροπρόθεσμο προγραμματισμό. Ποιο μπορεί τώρα, ειδικά τώρα αυτή την εποχή, να απευθυνθεί σε μια τράπεζα μέσα σε αυτή τη μεγάλη οικονομική κρίση και να εξασφαλίσει, να προσπαθήσει να εξασφαλίσει χρηματοδότηση ε, με ένα προγραμματισμό ή μια πρόβλεψη ετήσια, ενιάυσια. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα πλέον. Πρέπει να έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να προσφέρουμε πολυετή προγραμματισμό, αλλά όχι μόνο για αυτόν τον λόγο, όχι μόνο για τη χρηματοδότηση, αλλά και για να υπηρετήσουμε το στόχο της βιώσιμης αλίας. Και σε άλλες συζητήσεις λοιπόν ε, με εκπροσώπου Συμβουλίου στο παρελθόν το έχουμε τονίσει αυτό, αλλά ελπίζω ότι εσείς με την ιδιότητα σας τώρα ω Προεδρεύοντα ε, θα μπορέσετε να το προωθήσετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί και εσείς και εμείς ε, εδώ από το Κοινοβούλιο έχουμε σημαντική εντολή να προωθήσουμε αυτά τα θέματα της μακροχρόνιας προγραμματικής περίοδου η διαχείρισης ε, και αν δεν το καταφέρουμε φέτος, νομίζω θα έχουμε ουσιαστικά, εγώ τουλάχιστον για τον εαυτό μου θεωρώ ότι θα έχω αποτύχει στο έργο μου. Από το Δεκέμβριο του 2009 στη θητεία μας ήταν η πρώτη έκθεση που ε, ξεκίνησε αυτή η υπόθεση. Δεν μπορέσαμε να την προωθήσουμε. Τελικά είχαμε πει ότι μπορούμε να συμφωνούμε πως διαφωνούμε και αφήνουμε τα πράγματα έτσι. Το Συμβούλιο θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο έχει λάθος. Το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι το Συμβούλιο απατάται. Εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι θα πρέπει και μπορούμε πολλές φορές να διατυπώνουμε σαφείς επικρίσεις στις βάρος του Συμβουλίου ε, σε ορισμένα θέματα, αλλά εγώ πρέπει να πω ότι από τον τριμερή διάλογο που είδα να βιώνει να αναβιώνει πριν από μερικές εβδομάδες, μπορούμε να έχουμε κάποιες ελπίδες με, με επίσημες αλλά και με άτυπες συνεδριάσεις, μπορούμε να προχωρήσουμε πιστεύω βήμα το βήμα σε ένα καλό και θετικό αποτέλεσμα. Σήμερα αποδείξατε και εσείς πιστεύω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα ζητήματα των κυρώσεων πρέπει να τα εξετάσουμε διαφορετικά και ότι Μπορεί ίσως το θέμα αυτό να προχωρήσει στο Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια στοιχεία από τις ε, υπηρεσίες σας για το πότε μπορεί να μπει στο πρόγραμμα του Συμβουλίου. Ε, ίσως μετά την έγκριση του Κοινοβουλίου. Εμείς ξεκινάμε στις 12 Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρω εσείς πότε έχετε υπόψη τη συζήτηση και την απόφαση το θέμα αυτό και αν μου επιτρέπετε, χωρίς να έχω καμία διεκδίκηση ε, ότι μπορώ να σας δώσω συμβουλέ κύριε Υπουργέ, αλλά, αλλά σε ένα Υπουργικό Συμβούλιο, νομίζω πριν από κανένα μήνα περίπου, ε, έδινε, δόθηκε η εντύπωση από τη συνάντηση αυτών Υπουργών, στην ευρύτερη κοινή γνώμη, ότι οι Υπουργοί είναι εκείνοι, το Συμβούλιο δηλαδή είναι εκείνο το οποίο λαμβάνει τις αποφάσεις. Ε, αυτό τουλάχιστον βγήκε προ την κοινή γνώμη από του υπουργού. Παρακαλώ λοιπόν να υπενθυμίσετε στου ε, συναδέλφου υπουργού των κρατών μελών ότι δεν μπορεί το Σύμβουλο να λαμβάνει τι αποφάσει αυτέ. Η τελική απόφαση, μόνο μια ε, κρίση, μια σύσταση μπορεί να πάρει το Συμβούλιο αυτόνομα. Η τελική απόφαση και αυτό εδώ μπορεί να ισχύει για την Αλία, αλλά μπορεί να ισχύει και για οτιδήποτε άλλο. Θα γίνει μόνο, γιατί ισχύει, ξέρετε, η συνθήκη τη Λισαβόνα και ισχύει για όλου μα. Θα γίνει αναγκαστικά λοιπόν η απόφαση, θα περάσει μέσα από τη διαδικασία τη συναπόφαση, δηλαδή σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Αυτό το επισημαίνω, κύριε Πρόεδρε, χωρί όμω να θέλω να ε, παρέμβω κατά τρόπο στι εργασίες του ε, Συμβουλίου. Και πρέπει να πω ότι υπάρχουν ε, αποφάσεις οι οποίες μπορούν να λαμβάνονται χωρίς πρόβλημα όπως οι παραδείγματι τα τάκ και οι ποσοστώσεις ε, νομίζω ότι εκεί πέρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει καλό θα ήταν να το έχουν αυτό υπόψη οι συναδέλφοι σας στο Συμβούλιο. Η περιφερειοποίηση επίση για να ολοκληρώσω είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα πρέπει και η Επίτροπος και το Συμβούλιο να διακατέχονται από το πνεύμα της ε, Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να το τηρούν. Ξέρουμε ότι υπάρχουν περιπτώσει θεμάτων που δεν ενδιαφέρουν ορισμένα κράτη-μέλη γιατί ε, δεν έχουν γενική εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκείνοι λοιπόν, οι οποίοι, λοιπόν τα θέματα που θα πρέπει σε περιφερειακό επίπεδο να συζητηθούν και να κυρωθούν ε, μπορούν να περνάνε είτε από την Επιτροπή είτε από την Ολομέλεια. Ξέρω βεβαίω, κύριε Υπουργέ, ότι εσεί έχετε πολύ σκληρό έργο μπροστά σα, εσεί και η Επίτροπο βεβαίω. Πάντω, σα διαβεβαιώ ότι εμεί θα είμαστε και λογικοί και ρεαλιστές στην συζήτηση μαζί σας. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκάλερ, παρακαλώντα όλου όσου λάβουν το λόγο από εδώ και πέρα να είναι πολύ πιο σύντομοι, διότι δεν θα έχουν χρόνο όλοι για τι ερωτήσει. Ε, και ούτε ο κύριο Υπουργό να απαντήσει. Κυρία Λέβιν έχει τώρα μάλλον το λόγο. Να καλωσορίσω τον ε, κύριο Υπουργό στην ε, συνεδρία τη Επιτροπή μα. Να πω ότι άκουσα πολύ προσεκτικά αυτά τα οποία μας εξηγήσατε και για το φόρτο εργασία, Κάτι το οποίο έτσι συγκράτησα και ίσως είναι και ένα από τα σημαντικότερα είναι ότι θα καθοδηγήσετε το Συμβούλιο προς μια κοινή προσέγγιση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ανήκω στην ομάδα των Πρασίνων και από ό,τι γνωρίζετε, πολλοί βουλευτές της Επιτροπής μας δεν είναι ικανοποιημένοι σε σχέση με την προσέγγιση της, του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά το βασικό κανονισμό ε, και φοβούμε ακούγοντας ότι πολλές χώρες θέλουν ε, περισσότερη ευελιξία σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση. Δηλαδή θέλουν ε, χρήματα για την ε, ε, ναυπηγήση νέων πλοίων, τον εξυγχρονισμό κτλ. κτλ. Εγώ πραγματικά σας απευθύνω έκκληση να μην ξανακολουθήσετε αυτό το μονοπάτι, διότι ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στην τελευταία μεταρρυθμίση του 2004 αυτό σταμάτησε να κάνει σε ό,τι αφορά δηλαδή τη χρηματοδότηση για την ανανέωση του ε, στόλου, τον παροπλισμό του, στη διάλυση δηλαδή των ε, πλοίων και την ναυπήγηση νέων και αυτό οδήγησε σε υπεραλίευση. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να προστατεύσουμε τα λεύματα. Υπάρχουν πολλές μελέτες που δείχνουν ότι ε, αν καταφέρουμε να αποκαταστήσουμε τα μεγάλα ε, 132 τον αριθμό αλλιεύματα, τα οποία αλλιεύονται σε επίπεδα άνω ε, αυτών που επιτρέπουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν και θα διπλασιάσουμε τα αλλιεύματα και θα διπλασιάσουμε το εισόδημα ε, και θα μπορεί ο αλλιέας να έχει χρήματα για να μπορέσει να εξυγχρονίσει το στόλο του από μόνο του. Αυτό χρειάζονται οι φορολογούμενοι σήμερα. Είμαστε σε καιρό οικονομική κρίση. Και νομίζω ότι ο πολίτη δικαιούται να μας το ζητά αυτό σήμερα όχι να βάζουμε και πάλι κατά μέρο χρήματα για την υπεραλίευση, για υπερβολικέ αλληλευτικέ προσπάθειε. Δεν θα πρέπει να πάνε εκεί τα χρήματα. Τα χρήματα πρέπει να πάνε στην έρευνα, στον έλεγχο ε, και την αποκατάσταση των αλλημάτων, στα επιλεκτικά αλληλευτικά εργαλεία και σε όλα αυτά τα σχετικά. Εκεί πρέπει να ε, χρησιμοποιηθούν τα χρήματα των φορολογουμένων. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω πραγματικά ποια είναι η άποψη τη Κυπριακή Προεδρία για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας, πού θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ε, οι πόροι και πώς ε, προτίθεστε να καθοδηγήσετε το Συμβούλιο και σε ό,τι αφορά την κοινή προσέγγιση. Ευχαριστώ πολύ. Το έχει το λόγο η κυρία Ντότζ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως ε, και προλαλήσαντες, να σας καλωσορίσω και εγώ κύριε Υπουργέ στην Επιτροπή μας. Ελπίζω και πιστεύω ότι θα σταθεί με επιτυχία αυτό το καθήκον που λαμβάνετε. Και είναι σίγουρο ότι αναλαμβάνετε αυτά τα καθήκοντα μία πολύ σημαντική στιγμή για την αναθεώρηση τη κοινή ελληνική πολιτική, αλλά και για μια σειρά άλλων πραγμάτων. Πολλοί ήδη συνάδελφοι έθιξαν τα θέματα που απασχολούν την Επιτροπή μας. Εγώ θέλω να εστιάσω την παρέμβασή μου σε τρία ζητήματα που θεωρώ πολύ σημαντικά. Το θέμα είναι το ζήτημα της περιφερειοποίησης. Είμαι της γνώμης ότι η μεταρρύθμιση της κοινή αγροτική πολιτικής θα πρέπει να μας οδηγήσει σε πραγματική περιφερειοποίηση. Πολλοί αλλοί, τους οποίους εκπροσωπώ, πραγματικά έχουν φτάσει στα όρια τη αγανάκτηση από τον έλεγχο που ασκείται από Βεξέλλε, από την καθημερινή διαχείριση. Και πιστεύω ότι η καθημερινή διαχείριση θα πιο αποτελεσματικά από αυτού που ζουν εκεί επιτοπίως, που εργάζονται και γνωρίζουν πολύ καλύτερα τον τόπο τους και τη θάλασσά τους. Σίγουρα στην Ευρώπη εδώ χαράσουμε γενικέ πολιτικές, αλλά θα πρέπει να επιτύχουμε την περιφερειοποίηση αυτά και αποτελεσματικά. Θα ήθελα επίσης να πω ότι εξ όσων γνωρίζω, στο Συμβούλιο αυτή την εβδομάδα, ένα από τα θέματα που θα ανακύψουν εκ νέου είναι το θέμα του σκουμπριού και η υπεραλίευσή του από τους Ισλανδούς ε, και από τις αλληλείς από τις Φερόες νήσους. Είναι ένα θέμα το οποίο έρχεται και επανέρχεται εδώ και καιρό. Και πιστεύω ότι η Επιτροπή μας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σας δίνουν τα κατάλληλα εργαλεία για να μπορέσετε να συμφωνήσετε τελικά σε κάποιες κυρώσεις. Επιτέλους πρέπει και η Επιτροπή και το Συμβούλιο να αρχίσει να δουλεύει το του θέματος. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε ένα νέο γύρο διαπραγματεύσεων το Σεπτέμβρη όταν παραμένουμε αγκυλωμένοι στην ίδια κατάσταση η Ισλανδία και οι Φερές Νήσοι μονομερός να δηλώνουν αύξηση στα αποθέματα και στα αλληλευτικά τους δικαιώματα. Ενώ ταυτόχρονα τα αποθέματα έχουν, τα δικά τους αλληλευτικά αποθέματα έχουν χάσει τη διαπίστευση και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για αυτά τα αποθέματα. Εδώ και δύο χρόνια το λέμε εδώ στην Επιτροπή μας αλλά δεν έχουμε επιτύχει τίποτα σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα. Επιτέλους, επιτέλους πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις διαπραγματεύσεις του Σεπτέμβρη για να καταλήξετε κάπου, όπως και κυρώσεις να επιβάλλετε, καθώς πλέον υπάρχει συμφωνία από αυτόν. Το τελευταίο μου σχόλιο αφορά τα προγράμματα μακροχρόνιας διαχείρισης. Σας άκουσα μεγάλη προσοχή. Συμφωνούμε πιστεύω, στο εξή. Ένα από τα πλέον επιτυχή στοιχεία τα οποία αναπτύσσουμε είναι αυτή η ιδέα των μακρόπνων προγραμμάτων διαχείρισης. Δεν είναι δυνατόν κάθε χρόνο, ουσιαστικά στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, να υπάρχει αυτός ο αγώνας και η μάχη ανάμεσα στις κυβερνήσεις στην Κομισιόν για να αποφασίζουν τα τάκ και τις ποσοστώσεις. Ε, δεν είναι αυτός ο τρόπος για να βελτιώσουμε τα λευτικά αποθέματα, ούτε είναι ένας τρόπος για να βοηθήσουμε ε, τις αλληλευτικές κοινότητες και την αλληλευτική οικονομία. Πιστεύω ότι ο μόνος τρόπος για να βρούμε αποτελεσματικές λύσεις είναι τα μακροχρόνια σχέδια διαχείρισης. Το πρόβλημα όμως είναι το αδιέξοδο στο οποίο έχουμε περιέλθει. Αυτό το αδιέξοδο προέρχεται λόγω της ανάγκης ευθυγράμμισης με τις συνθήκες Λισαβόνας. Πρέπει λοιπόν να ευθυγραμμιστούν αυτά τα μακρόπνοα προγράμματα διαχείρισης με τις συνθήκες Λισαβόνας. Εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε τη βούληση, έχουμε την επιθυμία να συνεργαστούμε μαζί σας για να μπορέσουμε να φέρουμε αυτό το θέμα σε πέρα. Πρέπει να βρεθεί μια λύση γι' αυτό. Θα ήθελα πραγματικά να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή εσείς και η Προεδρία σας σε αυτό το ζήτημα και σε συνεργασία ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να καταλήξουμε σε μια λύση ώστε ομοιόμορφα να επιλύσουμε το πρόβλημα και να γίνει η ευθυγράμμιση με τη συνθήκη της Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Πατράου. Ευχαριστώ πολύ. Να σας καλωσορίσω και εγώ, κύριε Υπουργέ, και να ευχηθώ ότι καλύτερο για την Προεδρία σας. Θα ήθελα εντάχει να τοποθετηθώ επί δύο σημείων που θεωρώ μίζωνα. Ήθελα να πω την αλήθεια, να σας ακούσω να μιλάτε πιο πολύ για τα βασικά θέματα της αναθεώρησης κοινή πολιτικής αλίας. Και μάλιστα στην αδελφή μου ακριβώς προσανατόλισαν την τοποθέτησή τους σε αυτό το ζήτημα, γιατί είναι αυτό το θέμα που μας απασχολεί περισσότερο. Δηλαδή, πέρα από όλα όσα υπόθεσαν ήδη για το θέμα της μεταρρύθμισης, και θα ήθελα την τοποθέτησή σας, ε, λίγο πιο εντελεχώ επί το θέματο, ποια θα είναι οι θέσει που θα υπερασπιστείτε στα πλαίσια τη μεταρρύθμιση, εγώ θα ήθελα να επισημάνω το θέμα τη περιφερειοποίηση. Διότι πράγματι η περιφερειοποίηση έρχεται να φέρει εις πέρας να υλοποιήσει μια μακρά προσδοκία του κλάδου και πιστεύω και προσωπικά ότι μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά ε, στην αλληλεία στο μέλλον μια τέτοια διαχείριση σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με την ανάληψη ευθύνη από του ίδιου ενδιαφερόμενου στη διαχείριση. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αποτρέψουμε την παράνομη αλληλεία καλύτερα, να προάγουμε καλύτερα τι καλέ πρακτικέ. Θα ήθελα λίγα λόγια παραπάνω από εσά για αυτό το ζήτημα δεν χρειάζεται να πω εγώ ποια είναι τα ωφέλη αυτής της ε, διαχείριση. Θα ήθελα επίσης να σα ρωτήσω κάτι άλλο. Λίγα λόγια για τη συμφωνία με το Μαρόκο. Το αναφέρατε εν παρόδο, είπατε ότι είναι ένα περίπλοκο ζήτημα το θέμα του Μαρόκου, αλλά για μας είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Θα ήθελα να σας ακούσω λίγο παραπάνω πώς πάνε οι διαπραγματεύσεις για αυτή τη συμφωνία και ποιες είναι οι προσδοκίες και το χρονοδιάγραμμα που μπορείτε να μας διαγραφήσετε. Τέλος, όχι μια ερώτηση, ένα σχόλιο μου επιτρέπετε. Όλοι εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε ό,τι αφορά την πρακτική της αφαίρεσης ε, των πτερυγίων ε, του Καρχαρία, ε, Έχουμε την διαθέση με εσά. Θεωρούμε ότι είναι μια υπονείδηστη πρακτική που ήδη από το 2003 έχει απαγορευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε όλοι να φανθούν κατά. Αναμφίβολα λοιπόν ότι αυτός ο, ο φάκελος πρέπει να προωθηθεί ε, τάχιστα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πατράου. κυρία Τέγια. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να καλωσορίσω ως Ευρωβουλευτής από την Ισπανία και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στον κύριο Υπουργό και στην ε, Κυπριακή Προεδρία εν Είμαι πεπισμένη ότι οι ιδέες και οι προτάσεις και το έργο που θα επιτελέσετε ε, νομίζω ότι θα κάνουν ιστορία, την ιστορία που κάνουν οι έξυπνοι λαοί. Ελπίζω λοιπόν να επιβεβαιωθώ και έχετε ήδη, ε, με έχετε ήδη πείσει γιατί έχετε πολύ καλές ιδέες, αλλά έχετε και προκλήσεις, πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσετε. Και σίγουρα ακούσατε εμάς εδώ που είμαστε από πολλά και ποικίλα διαφορετικά περιβάλλοντα και γεωγραφικά και πολιτικά. Έχετε αντιμετώπιστε πρόκληση λοιπόν γιατί ακούτε πάρα πολλά και διαφορετικά από όλους μας. Και εγώ θέλω να αναφερθώ στα περί της αληθικής συμφωνίας με το Μαρόκο. Ίσως είναι πρόωρο γιατί μόλις αναλάβατε καθήκοντα, αλλά για εμάς τους Ισπανούς ήδη είναι αργά. Ε, ήδη για την ε, μικρή κλίμακα Σαλία, διότι στην Ανταλουσία, Έχουμε, ε, ξέρουμε τι προτάσεις έγιναν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μεγάλου Βελινεκούς, ε, και ουσιαστικά έχουν οδηγήσει στην εγκατάλειψη της αλίας 600 τουλάχιστον σκαφών για την μικρή κλίμακα παράκτια αλία. Και εδώ και Επτά μήνες περίπου ε, δεν μπορούν ε, τα σκάφη να βγουν ε, να ψαρέψουν. Δεν υπάρχει πραγματικά καμία πρόοδος ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο. Συμφωνώ με αυτά που ε, λέτε και υπάρχουν κάποιες προθέσεις αλλά δεν ε, γίνονται τα ίδια σε σχέση με άλλες περιφέρειες, με άλλες περιοχές του κόσμου και με άλλες χώρες. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω εξ ονόματος ε, των ψαράδων αυτών της Ανδαλουσίας, μιας γης που πραγματικά μαστίζεται από την ανεργία. Σας παρακαλώ λοιπόν πραγματικά εκ μέσω αυτών των ψαράδων που χυμάζονται να κάνετε ό,τι μπορείτε για αυτή τη συμφωνία, για αυτή την κατάσταση με το Μαρόκο. Και επίσης, σε ό,τι αφορά την πολιτική των απορρίψεων, υπάρχει μια ημερομηνία ε, που συμφωνήθηκε στο Συμβούλιο ε, και για την μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Ποια είναι η άποψή σας επ' αυτής της ημερομηνίας, του χρονοδιαγράμματος και τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει, ε, παραδείγματος χάρη στη Μεσόγειο. Στη Μεσόγειο δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη Μεσόγειο όπως τη Βόρεια Θάλασσα ή όπως τον Ατλαντικό. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν κατά προτίμηση να δοθεί δηλαδή μια προνομιακή και ειδική προσοχή και στην περιοχή αυτή της Μεσογείου. Γιατί νομίζω ότι έτσι θα εμπλουτιστεί συνολικά η όλη πολιτική. Πρέπει να έχουμε ένα ευρύ όραμα ε, η Αλία είναι κάτι όπως και η Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι ένα ψηφιδωτό, ένα μοσαϊκό, είναι πολύπλευρη, πολυεπίπεδη. Το ίδιο είναι και η Αλία. Είναι πολιτισμός, είναι αστρονομία, είναι τοπίο, είναι περιβάλλον, είναι τρόπος ζωής και πρέπει να συνεχίσουμε να προασπίζουμε την οικονομική βιωσιμότητα, την κοινωνική βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Είμαι πεπισμένη ότι από αυτήν την έννοια θα είστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε αυτά τα θέματα ιδίω εσεί. Γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι μπορούμε να προασπίσουμε ε, και ιδίω οι αλληλεί και ιδίω επαναλαμβάνω η μικρή παράκτια αλληλεία μπορεί να προστατεύσει ε, την ε, βιωσιμότητα αυτή και να την εξασφαλίσει. Και βέβαια συμπίπτει η Προεδρία σας και με την έγκριση του πακέτου για την κοινελευτική πολιτική. Τι θα γίνει και με αυτό το θέμα. Ο Πρόεδρος. Να μην καθυστερήσουμε άλλο, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Προεδρεύοντα. Έχει να αντιμετωπίσει σωρία ερωτήσεων. Πράγματι κύριε Πρόεδρε, έχουν τεθεί αρκετά θέματα, αλλά ευχαρίστως θα προσπαθήσω να δώσω κάποιες απαντήσεις είχε τεθεί αρχικά το θέμα για τα χωρικά ύδατα. Είναι ένα θέμα που απασχολεί αρκετά κράτη-μέλη και ειδικά πράγματι τα μεσογειακά μέλη που αντιμετωπίζουν προβλήματα ιδιαίτερα με τις τρίτες χώρες. Γι' αυτό το λόγο υποστηρίζουμε εμείς την ενίσχυση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων των περιφερειακών οργανώσεων αλίες για το θέμα αυτό αλλά δεν είναι ένα εύκολο θέμα που μπορεί να επιληθεί τόσο σύντομα και τόσο εύκολα. Ε, αντιλαμβάνομαι ότι η Επιτροπή μελετά το θέμα της ε, αναθεώρησης της αλλαγής των κανονισμών για τη Μεσόγειο το οποίο είχατε αναφέρει. Ε, τέθηκε ερώτηση κύριε Πρόεδρε για τα MSY από, από πού αντλούμε τα δεδομένα. Ε, είναι πολύ καλά γνωστό ότι συλλέγονται αυτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το θέμα της ε, υπερχωρητικότητας, του overcapacity, είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε περαιτέρω στο Συμβούλιο και όταν έχουμε οποιαδήποτε εξέλιξη, κύριε Πρόεδρε, έντιμα μέλη της Επιτροπής, θα σας ενημερώσουμε ανάλογα Τώρα όσον αφορά τις απορρίψεις, έχουν δεσμευτεί τα κράτη-μέλη για κατάργηση των απορρίψεων στη βάση μιας στεριακής προσέγγισης. Αντιλαμβάνομαι ότι η Μεσόγειος είναι διαφορετική από τις άλλες χώρες, από τον Ατλαντικό. Εμείς στη Μεσόγειο, και λέω εμείς γιατί η Κύπρος είναι στη Μεσόγειο, έχουμε μειχτά αλλιεύματα Οπότε είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα σίγουρα στη Μεσόγειο. Για την μέγιστη βιώσιμη απόδοση θέλω να, να διευκρινίσω ότι η θέση του Συμβουλίου είναι ότι στηρίζει τη μέγιστη δυνατή απόδοση μέχρι το 2015 όπου είναι δυνατό, αλλά όχι αργότερα από το 2020. Ξέρετε, πολλοί θα θέλαμε να βλέπαμε τέτοιες ημερομηνίες να είναι δεσμευτικές και τελεσίδικες. Ε, θα πρέπει όμως να υπάρχει και ένας χρόνος, μια περίοδος ε, προσαρμογής για να βάλουμε κάτω ρεαλιστικά προγράμματα και να λαμβάνουμε και υπόψη τις κοινωνικο-οικονομικές επιτυχίες των αποφάσεών μας. Ε, έγινε αναφορά για τις ε, εμπορικές ε, κυρώσεις για το θέμα του σκουμπριού. Το Συμβούλιο έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει την θέλησή του για να προωθηθούν μέτρα εμπορικών κυρώσεων. Βελπιστούμε ότι με την έγκριση της πρότασης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εφαρμόσει και τις ανάλογες πρόνοιες του κανονισμού αυτού. Έγινε αναφορά από αρκετούς, ε, κύριε Πρόεδρε, έντιμα μέλη της Επιτροπής, τα πολυετή σχέδια διαχείρισης που τα θεωρούμε πραγματικά ένα βασικό και θα επαναλάβω επιτυχεμένο εργαλείο της υφιστάμενης κοινή αλληλευτικής πολιτικής και σίγουρα θα πρέπει να παραμείνουν στον πυρήνα της νέας ανεθεωρημένης κοινής αλλιευτικής πολιτικής. Ε, το Συμβούλιο μετά από αρκετή σκέψη για την προσέγγιση που θα ακολουθήσει για αυτά τα σχέδια έχει αποφασίσει για το πολιετές διαχρηστικό σχέδιο για το Σαφρίδι για το οποίο έκανα αναφορά και στην ομιλία μου. Το Συμβούλιο θέλει σίγουρα να αποφύγει μικροδιαχείριση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό θέλει να αφαιρεθεί η πρόνοια για τον κανόνα ελέγχου αλίευσης από το σχέδιο αυτό. Περιφερειοποίηση έγινε και γι' αυτό αναφορά κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει μια ευρεία συμφωνία ότι η ανάπτυξη της πολιτικής για βιώσιμη εκμετάλλευση και διατήρηση των πόρων απαιτεί περισσότερη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων, περισσότερες λύσεις που να είναι προσαρμοσμένες στην αλία και λιγότερες δευτικές λεπτομέρειες που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποστηρίζομαι θερμά πραγματικά την περιφερειακή εφαρμογή της κοινή αλληλευτικής πολιτικής, ιδιαίτερα του σχεδιασμού και της εφαρμογής περιφερειακών πολιετό σχεδίο καθώς και για να είναι αποτελεσματικά τα διαχειριστικά μέτρα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες του τύπου της αλίας της κάθε περιοχής, της κάθε περιφέρειας και να προνούν τη συνεργασία των, των ενδιαφερομένων κρατών και των σχετικών φορέων. Έγινε αναφορά για την αναδιάρθρωση του στόλου. Σαν Συμβούλιο δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη επί του θέματος. Έγινε μια ανταλλαγή απόψεων και θεωρώ ότι χρειάζεται περισσότερη συζήτηση. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας θα πρέπει να βρεθεί μια σωστή ισορροπία για να καταλήξουμε σε ένα μέσο που να στηρίζει τελικά την κοινή αλληλευτική πολιτική για να γίνει τέλος πάντων το επάγγελμα του Ευρωπαίου Αλλιέα αξιοπρεπές και βιώσιμο. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Αυτός είναι ο στόχος της αναθεώρησης. Έγινε αναφορά, κύριε Πρόεδρε, τη ε, στη, διαφορά που υπάρχει στις κατεξουσιοδότητες συμπράξεις. Είμαστε ενήμεροι ότι το πεδίο αυτό είναι καινούριο και ότι για το, για, οι θέσεις για το πώς θα επιτευχθούν οι ευθυγραμμίσεις υπόκεινται σε διστάμενες απόψεις. Είναι θέματα αυτά μιας πιο πλατιάς, οριζόντιας θα έλεγα συζήτησης που συνεχίζεται μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ε, και εμείς όπως είπα και στην ομιλία μου θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση για να λήξει το θέμα αυτό, για να μπορέσουμε να κάνουμε πρόοδο. Για την αλληλευτική συμφωνία σύμπραξης με το Μαρόκο, που τέθηκε το ερώτημα αυτό, το Συμβούλιο γνωρίζει τα νομικά ζητήματα και δεσμεύεται να σεβαστεί πλήρως τους κανόνες του διεθνούς δικαίου έχετε ενημερωθεί για το περιεχόμενο της εξουσιοδότησης για διαπραγμάτευση που υιοθετήθηκε το Φεβράρι του 2012. Έχουν γίνει κάποιες προκαταρκτικές ανεπίσημες συζητήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το Μαρόκο, αλλά δεν άρχισε ακόμη καμιά ουσιαστική διαπραγμάτευση. Ε, στο Συμβούλιο τα κράτη-μέλη με ειδική πλειοψηφία αποφάσισαν έγκριση και υπογραφή και προσωρινή εφαρμογή του προηγούμενου πρωτοκόλλου, αφού θεωρήθηκε ότι αυτό είναι συμβατό με το διεθνές ε, δίκαιο. Κύριε Πρόεδρε, στο τέλος θέλω να δηλώσω δύο πράγματα. Η αναθεώρηση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής καθώς και τα πολυετή διαχειριστικά σχέδια αποτελούν την πρώτη προτεραιότητα της δικής μας Προεδρίας. Παίρνουμε το θέμα πολύ σοβαρά και δεν θα αφήσουμε κόπο και χρόνο για να πετύχουμε στο θέμα αυτό. Στο τέλος θέλω να δηλώσω κύριε Πρόεδρε αυτό που είπα και σε άλλες περιπτώσεις, σε συναντήσεις που είχαμε. Ότι σέβομαι και αναγνωρίζω το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως αυτό προκύπτει από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει το Ευρωκοινοβούλιο. Δηλώνω το σεβασμό μου και είμαι έτοιμος για συνεργασία, διότι όπως είπα και χθε σε μια άλλη επιτροπή που παρουσιάστηκα, υπάρχει η λογική της φιλοσοφίας πίσω από την αλλαγή αυτή. Θέλει ο, Κύπρ, ο, ο πολίτης της Ευρώπης να νιώθει ότι οι αποφάσεις λαμβάνουν υπόψη τους εκλελεγμένους εκπροσώπους του. Και όχι μόνο μια ομάδα υπουργών και κάποιους γραφειοκράτες στα γραφεία του Βρυξελών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Προεδρεύοντα. Θέλω απλά να σας επαναλάβω ότι οι θύρες της Επιτροπής μας είναι ανοιχτέ και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε μια πολύ επικοδομητική συνεργασία κατά το εξάμεινο της Κυπριακής Προεδρίας. Σας ευχαριστώ και πάλι. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, συνεχίζουμε με το σημείο 11 της ημερήσιας διάταξης, που είναι η παρουσία της μελέτης «Ο ρόλος της Κίνας στην παγκόσμια λία». Όπως γνωρίζετε, είχε προταθεί η διενέργεια αυτής της μελέτης, ώστε να έχουμε στον δυνατόν μια ευρύτερη εικόνα για την αλία στην Κίνα, τις συναφείς δραστηριότητες για να δούμε ακριβώς ποιος είναι και ο ρόλος της Κίνας ε, στον τομέα της παγκοσμίας αλληλείας. Και βέβαια ε, είχαμε και προγραμματίσει και μια αντιπροσωπεία, επίσκεψη αντιπροσωπείας ε, στην Κίνα, αλλά έκτοτε ακυρώθηκε του λόγους που όλοι γνωρίζετε αυτή η επίσκεψη. Τέλο πάντων, όπως και να έχει, καλό είναι που έχουμε αυτή τη μελέτη. Ε, μπορούμε να την επεξεργαστούμε και μπορούμε να διαμορφώσουμε μια πάρα πολύ σαφή εικόνα για πολλά από τα θέματα που αφορούν μια μεγάλη δύναμη όπως είναι η Κίνα. Όλοι οι βουλευτές έχετε ήδη λάβει την έκθεση αυτή. Έχει διανεμηθεί νομίζω μόνο στα αγγλικά. Έχουμε εδώ έναν από τους ε, συντάκτες της μελέτης, τον Ντανιέλ Παουλή. Θα τον ακούσουμε καταρχάς και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν ενδεχομένως ερωτήσεις προς τους συντάκτες. Κύριε Πολύ, έχετε το λόγο. Και βέβαια να σας ευχαριστήσω που βρίσκεστε εδώ σήμερα. Thank you, Chair, for Ευχαριστώ Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την παρουσίαση. Δεν είμαι ο δόκτωρ πολύ, το πολύ είναι εδώ πίσω στην αίθουσα. Εγώ θα πω λίγα εισαγωγικά λόγια για αυτή τη μελέτη, η οποία εκπονήθηκε από μία ομάδα μεταξύ αυτών και ο δόκτωρ Πολύ από το British Columbia στο Βανκούβερ, μαζί με την Μέγκα Πέσκα, πορτογαλική εταιρεία και την Πλούμα Chance, τη δική μας ε, ε, εταιρεία που έκανε το συντονισμό. εντάχει. Πώς ε, οργανώσαμε να κάνουμε αυτή την παρουσίαση. Πρώτα πω όλα θα πω λίγα λόγια για τους στόχους και τη μέθοδο και μετά θα σας παρουσιάσουμε τα κύρια ευρήματα της μελέτης, καταλήγοντας σε συμπεράσματα και συστάσεις. Εντάχει να πω ότι οι στόχοι ποιοι είναι. Βασική μας πρόθεση είναι να δώσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή σας μια γενική εποπτεία της κατάστασης σχετικά με το ρόλο της Κίνας στην παγκόσμια ελεία. Ε, μια σειρά θεμάτων όπως η παράνομη, άναρχη και ελαθρέα ηλία, η ηλία υγιού. Θεωρούμε ότι χωρίς τη συμμετοχή της Κίνας σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, είναι δύσκολο τέτοιες πρωτοβουλίες να τελεσφορήσουν. Λαμβάνοντα υπόψη ε, το μέγεθος της Κίνας στην παγκόσμια ηλία. Έπειτα, είναι σημαντικό να δούμε ότι αυτή η μελέτη εστιάζει στα θαλάσσια λιεύματα, δηλαδή δεν μελετήσαμε τις ε, τα εσωτερικά ύδατα ή τις υδατοκαλλιέργειες. Ε, επίσης εστιάσαμε πιο πολύ στην υπηρετική Κίνα, Χονγκ Κόνγκ, Μακάο, δεν περιλαμβάνονται σε αυτή τη μελέτη. Κύριοι, ε, έξι κύριοι βασικοί τομείς, αλλιεύματα, στόλοι, εμπορικά ζητήματα, εισαγωγικές εξαγωγές αλλιευτικών προϊόντων, δραστηριότητες κινέζικου στόλου εκτός ε, κινέζικων υδάτων και τέλος η παράνομη αναρχή και ελαφρέα αλία. Τώρα θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο, στον δόκτορα Πολύ, ο οποίος θα σας μιλήσει για τα αλλιεύματα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ τα κύρια ευρήματα αυτής της μελέτης ε, τα έχετε ενώπιόν σας. Η α, Κίνα ενημερώνει ε, την ΦΑΟ για τα λιεύματά της. Βλέπετε τα αιτήσια λιεύματα όπως έρχονται από τα εγχώρια της ύδατα, από την άλλη όμως δεν μας δίνει εμπαρκή στοιχεία σχετικά με την αλίευση εκτός των κινέζικων χωρικών υδάτων. Εκτιμούμε λοιπόν 4 με 5 εκατομμύρια τόνους αλιευμάτων εκτός Κίνας από κινέζικα σκάφη. Και εξ αυτών το 10% μόνο καταγράφονται στη ΦΑΟ. Τα κινέζικα σκάφη καταγράφονται ως με κινέζικο πλήρωμα όχι να φέρουν τη σημαία της χή της χώρας, γιατί οι σημαίες ευκαιρίε αλλάζουν ε, εύκολα. Μιλούμε για κινέζικες εταιρείε με κινέζικο πλήρωμα, κατά κανόνα. Κατά κύριο όγκο τα αλλιεύματα προέρχονται από την Αφρική, πάνω από 3,1 εκατομμύρια τόνοι. Ασία, 1 εκατομμύρια τόνοι και λοιπές περιοχές. Αυτό το βουνό που βλέπετε σε αυτό το διάγραμμα είναι τα καταγεγραμμένα εγχώρια κινέζικα αλλιεύματα. Το 2001 δημοσιεύσαμε μία μελέτη ότι αυτά τα αλλιεύματα είναι παράλογα, είναι αδύνατο είναι πραγματικά. Και αν τα συγκρίνουμε με τα ιαπωνικά και ρωσικά αλλιεύματα στην ίδια περιοχή, βλέπετε ότι το 1980 φτάνουμε στο ανώτερα ποσοστά και μετά βλέπουμε μία μείωση. Θα τις χωρε μόνο στην Κίνα συνεχίζεται η αύξηση. Η αύξηση γίνεται μόνο για πολιτικου λογου γιατί ανταποκρίνεται σε ένα σχέδιο, δεν είναι μια πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα τα αλλιεύματα τη κινα είναι 5 με 6 εκατομμύρια τόνοι εντό Κίνας αναφέρουν τόσο υψηλά αλλιεύματα, ώστε να παρέμβει η κινέζικη κυβέρνηση και να πει δεν θα αυξηθούν. Έτσι λοιπόν η Κίνα όρισε αυτά τα ανώτατα ωραία στα 13 εκατομμύρια. Και έχουμε λοιπόν μια σταθερή κατάσταση α, από 1990 και μετά. Η ΦΑΟ κάλεσε την Κίνα να δώσει ρεαλιστικά στοιχεία. Και έτσι βλέπουμε και κάποιες μικροδιαφοροποίησεις, το 13%. Γι' αυτό βλέπετε μια μικρή διαφοροποίηση και όχι μια ευθεία γραμμή πλέον. Πέρα από αυτό, να πούμε ότι η Κίνα ενημερώνει για αλλιεύματα έξω από το δυτικό βόρειο ειρηνικό. Αυτά είναι τα αλλιεύματα που ενημερώνει για εκτός των χωρικών της και είναι πολύ χαμηλά. Γι' αυτό λοιπόν κάναμε αυτή τη μελέτη και αρχικά εκτιμ... κάναμε μια εκτίμηση του πού επιδίδεται η Κίνα. Μιλάμε για την ε, λαϊκή δημοκρατία της Κίνας και όχι την Ταϊβάν εδώ. Ε, βλέπετε λοιπόν με κόκκινο την αποκλειστική οικονομική ζώνη χωρών όπου επιδίδεται δραστηριότητα ε, ή καταγράφεται ότι επιδίδεται δραστηριότητα η Κίνα. Η κίτρινη γραμμή είναι η Ανταρκτική, όπου και εκεί ε, έχει δραστηριότητα η Κίνα. Εκτός εκει λοιπόν της Καραϊβικής. Η κινα εκτος λοιπον της καραιδικης η κινα βρίσκεται παντού στο τροπικό και τον υποτροπικό κύκλο και σε όλους τους ωκεανούς εκτός του Βόρειο Ατλαντικό. Αυτή η κίτρινη γραμμή είναι η ΑΟΣ που α, διεκδικεί η Κίνα. Τώρα για κάθε μία χώρα χωριστά κάναμε ενδελεχή έρευνα όλων των διαθέσιμων στοιχείων από άρθρα σε εφημερίδες, από επιστημονικές καταχωρήσεις, από το ίντερνετ και στην Κίνα, διότι είχαμε ε, στην ομάδα μας και Κινέζους επιστήμονες. Σε μια ομάδα 15 ε, μελετητών, 5 ήταν Κινέζοι. Κάναμε λοιπόν ενδελεχή λεπτομερή έλεγχο όλων των διαθέσιμων στοιχείων και επίσης προσπαθήσαμε να υπολογίσουμε τον πιθανό ρυθμό σκαφών, οι οποίοι βεβαίως έχουν και ένα περιθώριο λάθους για να καλύψουμε και αυτή την ε, αβεβαιότητα ε, που υπάρχει. Και μιλάμε για μια περίοδο 2000-2011, για την περίοδο έρευνας. Για κάθε σκάφος μετά για κάθε κατηγορία σκάφους, μάλλον, συσσωρεύσαμε από τη βιβλιογραφία για την αλληλεία τα τυπικά αλληλεύματα. Τα τυπικά λοιπόν για σκάφη με πολλαπλά αλληλεύματα. βλέπετε εδώ τα, ε, τους διάφορους ε, αν θέλετε, δείκτες και ε, ανακατηγορία ε, εργαλείων για την αλίευση του τόνου, για την αλίευση με γρηγρή, με παρασυρώμενα δίκτυα λοιπά Βλέπετε τις κατηγορίες. Και μετά με τον αριθμό των σκαφών ανακατηγορία εργαλείου από κάθε χώρα με αυτό που βλέπετε εδώ στην οθόνη. Και βλέπετε ότι δεν έχουμε κανένα μεμονωμένο ρυθμό για οτιδήποτε. Βλέπετε πάντα μια γκάμα, μια ψαλίδα. Αυτή είναι η μέθοδος Μοντεκάρλο. Δηλαδή, επαναλαμβάνεις 100.000 φορές. Ένα τυχαίο δείγμα ενό αριθμού από αυτή την κατανομή, κάνει όλου του υπολογισμού με αυτό το αριθμό και το επαναλαμβάνει. Και έτσι, αντί να επιλέξει έναν αριθμό, π.χ. τον αριθμό των σκαφών στη Μοζαμβίκη, παίρνει 10.000 αριθμούς, το πολλαπλασιάζεις επί 10.000 από εδώ πως βλέπετε. Και αυτό έγινε για τις 80 χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η Κίνα με όλες τις κατηγορίες σκαφών. Και να τα αποτελέσματα. Περίπου χίλια σκάφη εντοπίζονται να δραστηριοποιούνται σε αυτές τις 80 χώρες. Αυτό φαίνεται να είναι χαμηλότερο και από αυτό που παραδέχεται η Κίνα. Κίνα παραδέχεται 2.000 σκάφη. Δεν μπορούσαμε λοιπόν να λύσουμε αυτό το μυστήριο, γιατί η Κίνα έχει και σκάφη που δραστηριοποιούνται στην Κορέα και αυτά θεωρούνται εγχώρια δραστηριότητα, γιατί η Κορέα η είναι πολύ κοντά. Οπότε εδώ υπήρχε ένα πρόβλημα στη διάκριση. Μιλάμε για σκάφη που ανήκουν στα 2.000 σκάφη που δηλώνει η Κίνα ή τα ε, εν μέρη εγχώρια σκάφη, εγχώριες δραστηριότητε. Οπότε εμείς χρησιμοποιούμε μια εκτίμηση χιλίων σκαφών που δραστηριοποιούνται σε μακρινά ύδατα. Αυτά τα χίλια σκάφη σε συνδυασμό με την κατανομή των αλλιευμάτων ενός τυπικού σκάφους δίνει ένα μέσο αλλιεύμα 4,6 εκατομμυρίων τόνων συν πλην 600.000. Βλέπετε λοιπόν το 3,5 εκατομμύρια και πάνω ε, είναι στην Αφρική. Και αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία που εκτιμούμε. Με πολλέ συνέπειε όμως, διότι η Κίνα δεν δηλώνει πάνω από 400.000 τόνους. Άρα μιλάμε για ενιαπλάσιο, δεκαπλάσιο όγκο αλλιευμάτων σε σχέση με, τις, ε, με, τα δηλωμένα αλλιεύματα. Αυτό, επαναλαμβάνω, δεν μας επιτρέπει να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στα νόμιμα και παράνομα αλλιεύματα. Γιατί η Κίνα ίσως να έχει μια συμφωνία με κάποιες χώρες, αλλά τα ΜΜΕ, οι επιστήμονες σε αυτή τη χώρα δεν γνωρίζουν τη φύση αυτής της συμφωνίας. Άρα, τι θα πούν. Κίνα κάνει παράνομη αλληλεία στη χώρα Χ, σε μια χώρα με την οποία έχει συγκρούσει, ενώ αυτό δεν ισχύει. Μα εγώ δεν λέω ότι δεν κάνει παράνομη αλληλεία η Κίνα, αλλά λόγω των συμφωνιών, της φύσης των συμφωνιών που έχει συνάψει η Κίνα, συχνά είναι δυσδιόρατα, αν θέλετε, τα όρια ανάμεσα στο παράνομο και το νόμιμο. Και δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα θέσουμε αυτό το όριο. Δεν ξέρουμε δηλαδή αν μπορούμε να μιλήσουμε για παράνομα αλλιεύματα, υπό την έννοια της παράνομης, λαθρέας και άναρχης αλλίας. Με αυτή την έννοια της παράνομης αλλίας. Για την Αφρική και μόνο, 2,5 εκατομμύρια τόνοι είναι αυτά που δεν δηλώνονται. 5 έως χιλιάδες, 500 ε, τόνοι δηλώνονται ως συμπράξεις. Δηλαδή ένα πολύ μικρό κλάσμα αυτού του αλληλεύματος στην Αφρική μπορεί να δηλώνεται μεν, αλλά ως ε, σύμπραξη αλίευσης με Μοζαμβίκη ή με οποιαδήποτε άλλη αφρικανική χώρα. Επίσης, δεν κάναμε χωριστή αξιολόγηση των αλλιευμάτων στην ανοιχτή θάλασσα και στα, ε, κοντά, ε, στις παράκτιες περιοχές. Διότι μπορεί να υπάρχει νόμιμη αλληλεία στη ανοιχτή θάλασσα και παράνομη στην αποκλεισμή. Εκεί λοιπόν μπορεί να υπάρχει ε, μια δυσδιο, δυσδιάκριτη κατάσταση και δεν μπορεί κανείς να ορίσει τα όρια ανάμεσα στην παρανομία και την ομιμότητα στην αλληλευτική προσπάθεια. μπορεί κανείς να υπολογίσει τι θα πει ο Κινέζος πρέσβης, ότι είναι σφαλμένα αυτά τα συμπεράσματα. Αλλά στην Κίνα πουθενά δεν υπάρχει καμία δημοσίευση, ε, πουθενά ούτε στο ίντερνετ, πουθενά, καμία εκτίμηση για την ε, αλίευση, την ελευτική προσπάθεια ε, εκτός χώρας. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν, δεν γνωρίζουν στην Κίνα τέτοια στοιχεία. Έπειτα ένα άλλο μέρος αυτής της μελέτης εξετάσει το τι δηλώνει η ίδια η Κίνα. 300... 3.000 ε, περίπου ε, σκάφη στην εσωτερική εγχώρια δραστηριότητα και προσπαθεί να μειώσει τον στόλο και με, ο ένας τρόπος για τη μείωση αυτού του στόλου είναι να στέλνει ένα μέσο αυτού του στόλου για δραστηριότητα στο εξωτερικό. Δεν μιλάμε λοιπόν για σκάφη που ναυπηγούνται ειδικά για αλληλεία ε, στο εξωτερικό. Λοιπόν, συχνά είναι και στα πιο κάραβα. Δηλαδή είναι σκάφη που εργάζονται 24 στο 24 ώρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. Και για αυτόν τον λόγο ε, νικούν κατά κράτος τους ισπανικούς τόλους κτλ. Λοιπόν, στο έγγραφό μας έχουμε και μία σειρά στατιστικών στοιχείων για την Κίνα, ότι δηλαδή η Κίνα είναι μαζικός αγωγέας ε, ψαριών για επεξεργασία και μεταποίηση ε, και έπειτα κάνουν επανεξαγωγές. Οι επανεξαγωγές εν μέρη είναι νόμιμες, εν μέρη παράνομες είναι δύσκολο και εκεί να μπει η διαχωριστική γραμμή. Οι διάφορες τώρα ε, επαρχίες ε, της Κίνας που ουσιαστικά αντιστοιχούν ε, σε μια ευρωπαϊκή χώρα σε, βαθ... σε ό,τι αφορά τον όγκο των εισαγωγών εξαγωγών. Τουλάχιστον σε ό,τι δηλώνουν. Αλλά με βάση τα δικά μας στοιχεία Προσπαθούμε να κάνουμε εκτιμήσεις με βάση αυθεντικά στοιχεία, όχι με βάση ότι μας λένε οι Κινέζοι. Βέβαια στα κινέζικα στατιστικά στοιχεία πάντοτε πρέπει κανεί να τα βλέπει με επιφύλαξη. Γι' αυτό και προσπαθούμε να βρούμε αυθεντικά στοιχεία. Ξέρετε, η Κίνα έχει πολλέ δυσκολίε. Δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ούτε καν δεν θα βρει κανείς γυαλί μέσα ε, σε μια παιδική τροφή. Υπάρχουν τέτοια σοβαρά προβλήματα. Βλέπετε πόσα σκάνδαλα διατροφικά έχουν υπάρξει στην Κίνα. Η Κίνα πασχίζει να ελέγξει, να αντιμετωπίσει το φαινόμενο το κατά πόσον έχει επιτυχία ή όχι ε, στις προσπάθειές της, αυτό μπορείτε να το κρίνετε εσείς. Η Κίνα θέλει να ενταχθεί, να είναι μέλος της διεθνούς κοινότητας, αλλά οι πρακτικές της διέπονται από αδιαφάνεια. Γι' αυτό και υπάρχει και γνωστή έκφραση «εμένα αυτά μου φαίνονται κινέζικα», λόγω αδιαφάνειας. Ξέρετε, στο Βανκούπερο που ζω εγώ, ε, έχουμε πως πολλούς Κινέζους προσπαθούν να γεφυρώσουν αυτό το χάσμα και την ε, έλλειψη κατανόησης. Λοιπόν, ε, θα φτάσω και σε κάποιες συστάσεις προσπαθώντας να κρατήσω το χρόνο μου που μου δώσατε. Ουσιαστικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη θα πρέπει να πιέσουν μέσω ε, της ΦΑΟ να κάνει η Κίνα ε, δήλωση των πραγματικών αλλιευμάτων. Αυτό είναι σκάνδαλο. Δεν είναι κάτι απλά εσφαλμένο, είναι κάτι που ανήκει σε άλλο πλανήτη αυτό που συμβαίνει. Αν θέλουμε να γνωρίζουμε τι συμβαίνει στην Κίνα, πρέπει να δημιουργήσουμε μια ειδική μονάδα. Ίσως ε, σε ένα πανεπιστήμιο ή μια ερευνητική μονάδα που να ασχολείται αποκλειστικά με αυτό το θέμα. Και οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να μιλούν κινέζικα. Για να βρεις πληροφορίες πρέπει να σκάψεις πολύ βαθιά. έπειτα οι σχέσεις μας, οι σύνδεσμοι που έχουμε με άλλες χώρες, με τρίτες χώρες. Πρέπει να τους ενθαρρύνουμε να είναι ειλικρινείς και διαφανείς. Διότι αν δεν μας αποκαλύπτουν τους όρους της συμφωνίας που έχουν συνάψει με την Κίνα, τι να κάνουμε. Η Ευρώπη θέλει να είναι ε, ένας θεμητός, αν θέλετε, παίκτη. Θέλει να είναι το καλό παιδί, θέλει να παίζει τίμια το παιχνίδι. Αλλά να πώς έχει κατάσταση. Ξέρετε, αυτό που αντιμετωπίζει πολύ συχνά η Ευρώπη έναντι των ΗΠΑ είναι η ίδια κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουν οι αφρικανικές χώρες με την ε, Κίνα. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια. Τώρα, η ιδιοκτησία των στόλων. Κανείς δεν γνωρίζει σε ποιον ανήκει ένα ε, σκάφος. Αλλάζουν σημαία, ίσως όσο συχνά εγώ αλλάζω εσώρουχα. Εντάξει, μπορεί να υπερβάλλω. δεν ξέρουμε τίποτα ουσιαστικά. Σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποίησαμε εμείς τη μελέτη μας ε, ως κριτήριο κινέζικο σκάφος, κινέζικο πλήρωμα. Πολύ συχνά δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το, πλήρωμα, ε, αυτό το, κριτήριο, γιατί να διευκρίνησε τα στοιχεία. Επίσης, έχουμε μία σύσταση για την παράνομη αλλήλεια, Λέγοντα ότι η παράνομη αλληλεία θα πρέπει να μπει στο ποινικό δίκαιο. Δεν είναι θέμα έρευνας, δεν είναι θέμα διαχείρισης αλληλευτικών αποθεμάτων. Είναι θέμα, ε, θα πρέπει μάλλον να είναι θέμα διεθνούς ποινικού δικαίου. Αυτά ουσιαστικά. Σε ευχαριστώ πολύ. Thank you very much indeed. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο και εμάς μας έχει απασχολήσει εδώ και αρκετό καιρό στην ε, Επιτροπή Αλίας. Έπρεπε να μάλιστα να επισκεφθούμε ε, την ε, Κίνα με την αντιπροσωπεία μας στο τέλος του χρόνου, αλλά λόγω κάποιων ιστορικών διαμαχών από το Politburo του Πεκίνου ενημερωθήκαμε ότι δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε την επίσκεψη. Ελπίζουμε όμως να τα καταφέρουμε κάποτε και να επισκεφθούμε την Κίνα εξοπλισμένη με τις εκθέσεις. Μέχρι τώρα δύο συναδελφοί ζήτησαν τον λόγο. Κύριο κύριος Ρωμέβα και ο κύριος Παράλαβαν μετά. Uh, σας ευχαριστώ πρόεδρε. Προφανώς περιμένω με αδημονία να μελετήσω ολόκληρη την έκθεση. Είναι θέματα πολύ ενδιαφέροντα και μόλις βρω το χρόνο θα τη μελετήσω. Πάντως ε, θα ήθελα να κάνω μια γενική ερώτηση ξεκινώντας. Ξέρουμε τώρα που γίνεται η αλίευση αυτών των ηχθείων. Το θέμα είναι όμως ξέρουμε που πολλούνται τα ψάρια αυτά και πώς μπορεί να εξασφαλιστεί η χνηλασιμότητα των προϊόντων κάποια κινέζικη επιχείρηση που παραδείγματα τα διακινεί και οι Ευρωπαίοι πώ μπορούν να τα βλέπουν όλα αυτά, έρχονται σε ευρωπαϊκέ αγορέ. Απάντηση. Η μελέτη μα δεν επικεντρώθηκε στο θέμα αυτό. Ωστόσο, από τα όσα μελέτησα, και πρέπει να σα πω ότι έχω διαβάσει πολλά εντωμεταξύ, έχω την αίσθηση ότι ένα τρίτο των αλλιευμάτων της υπερπόντιας, του υπερπόντιου στόλου της Κίνας ε, τη χάνει επεξεργασία και πολίτε στο εσωτερικό τη χώρα. Το 1 τρίτο. Το άλλο τρίτο στην ε, ε, διεθνή αγορά, ιδιαίτερα τα ασπόνδυλα, καλαμάρια και ούτω καθεξής. Και άλλο ένα τρίτο εισάγεται στην Κίνα. Πάντως πρέπει να πούμε ότι αυτά τα σκάφη είναι όλα αληφτικά σκάφη τροφοδοτούν με το κεντρικό μητρικό σκάφος όπως ονομάζεται ε, στην μακρά περίοδο που μένουν στην ανοιχτή θάλασσα ε, τροφοδοτούν, αλληλοτροφοδοτούνται με το κεντρικό μητρικό σκάφος ε, και σε εξοπλισμό, εξαρτήματα αλλά και σε τροφή και τα υπόλοιπα αλλιεύματα πηγαίνουν στο, στις χώρες της περιοχής για το 1 τρίτο. Τώρα τι κάνει και πώς διοχετεύει σε άλλες χώρες εκείνα αυτά τα αλλιεύματα δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ τον Δόκτωρα Πόλη για την πολύ ενδιαφέρουσα ε, παρουσίασή του. Πολλά καινούρια στοιχεία εμφανίζονται και ακούγονται. Θα προσπαθήσω λοιπόν να τα βάλω σε μια τάξη για να αντιληφθώ καλύτερα την κατάσταση. Έχω αρκετέ ερωτήσει λοιπόν. Η πρώτη ερώτηση είναι. Γιατί φαντάζομαι ότι εσείς ε, παρουσιάσετε στους Κινέους τα, στοιχεία αυτά και του ζητήσατε μια απάντηση. Ποια ήταν η επίσημη απάντηση λοιπόν που έδωσε η Κίνα για τα στοιχεία αυτά. Δεύτερον, μας είπατε ότι υπάρχουν ε, και χίλια ακόμη ελευτικά σκάφη στα νερά, στα έξω από την Κίνα. Αυτοί όμως μας λένε ότι έχουν δύο χιλιάδες ελευτικά σκάφη. Δηλαδή είναι μάλλον μετριοπαθής η δική σας εκτιμήση και άρα ε, αλλιεύουν περισσότερες, μεγαλύτερες ποσότητες ακόμη ψαριών. Τρίτον, λέτε ότι α, κινέζικο είναι ένα πλοίο όταν έχει πλήρωμα Κινέζου, έστω και αν ε, πλέει υπό διαφορετική σημαία. Άρα ε, διαρωτώ με το αλλιεύμα αυτό ενδέχεται να δηλώνεται σε άλλη χώρα, τη χώρα της σημαία αν προκειμένου και ενδεχομένω να περνάει μη δηλω... μη δηλωμένο ή δηλωμένο σε άλλη σημαία. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Ναι, εάν ξεκινήσω από την τελευταία ερώτηση. Ε, από τις εφημερίδες και τις πληροφορίες, τις λοιπές πληροφορίες που συλλέγουμε, αποδεικνύεται, φαίνεται ότι εντοπίζεται χάρη στο προσωπικό του και, χαρακτηρίζεται ως κινέζικο ένα σκάφος και όχι από, το, ε, από τη σημαία ή λόγω της συμπεριφοράς του, του τρόπου δράσης δηλαδή του σκάφους. Υπάρχουν περιοχές στην Νότια Αμερική όπου μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι είναι ταϊβανέζικα τα σκάφη και δεν υπάρχει τρόπο να γίνει η διάκριση μεταξύ κινέζικου και ταϊβανέζικου. Στην Νότια Καραϊβική νομίζω μόνο υπήρξε κάποια επικάλυψη συγκεκριμένα που δεν ήταν σαφές αν πρόκειται για τα Ιβανέζικο και Κινέζικο σκάφος. Εγώ νομίζω πάντως ότι ο ορισμός μας είναι καλός. Οι δηλώσεις αυτών των ε, ε, κινέζικων εταιριών ε, που καταγράφουν, καταχωρίζουν εθνικό αλλιεύμα μόνο και μπορούμε να το πούμε μόνο για την Αφρική γιατί από εκεί έχουμε το 1 δέκατο των δηλώσεων των καταχωρήσεων ως εθνικών ε, αλλιευμάτων καταχωρίζεται. Άρα μπορεί το 1 τρίτο που σας λέω εγώ ότι πολίτες εθνικό, στην εθνική αγορά είναι σφαλμένο γιατί θα πρέπει να γίνει η εκφόρτωση. Αυτό κάπως, σε αυτό δεν μου βγαίνουν τα, τα νούμερα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το μεγαλύτερο ποσοστό, τα 9 δέκατα θα έλεγα αυτών των αλλιευμάτων, είναι αδήλωτη, παράνομη και λαθρέα ε, και άναρχη αλλία. Η Διεθνής Οργάνωση μας λέει ότι είναι μόνο το... είναι ένα λιγότερο από ένα δέκατο έξω από τη ζώνη της ε, ΕΦΕΙΟΥ. Άρα το υπόλοιπο είναι IUU. Παράνομη λαθρέα και αναρχελία δηλαδή. Αλλά ομολογώ εντωμεταξύ ότι ξέχασα την πρώτη σα ερώτηση. Μπορείτε να μου την υπερθυμίσετε. Ναι, ποια ήταν η επίσημη αντίδραση από πλευρά των Κινέζων και μια δεύτερη τώρα, αν μου επιτρέπετε, μια και μου φαίνεται ενδιαφέρον. Εξαγωγέ από την Κίνα, που είναι ο μεγαλύτερο εξαγωγέ ανά τον κόσμο. Τι μερίδιο των ψαριών που εξάγονται έχουν ψυχή στην εσωτερική αγορά και ξέρετε στη συνέχεια. Να σας απαντήσω, επειδή ολοκληρώθηκε πρόσφατα αυτή η μελέτη, εγώ δεν είχα την ευκαιρία να την ε, παρουσιάσω πάνω από μία φορά και έτσι... να έχω πολλές αντιδράσεις από Κινέζους, γιατί μόνο μία φορά την παρουσίασα ε, με παρουσία Κινέζων, όπου η αντίδραση ήταν απλούστατα δεν έχεις δίκιο, είναι λάθος. Δεν υπήρξε δηλαδή διάλογος αντιπαράθεση απόψεων και επιχειρημάτων. Την ίδια εμπειρία είχα πριν από 10 χρόνια, όταν για πρώτη φορά δημοσιεύσαμε τη μελέτη ε, που έλεγε ότι είναι αδύνατο να έχει τόσο υψηλό εγχώριο αλίευμα. Εν πάση περιπτώσει στην Κίνα μπορεί κάποιοι να γνωρίζουν τα πράγματα, αλλά δεν μιλάνε. Έχω ένα Κινέζο συνάδελφο που έχει ένα συνάδελφο ή συναδέλφου, που του λένε ότι δεν είναι τόσο υψηλό το εθνικό, το εσωτερικό, το εγχώριο συγγνώμη αλλά δεν φτάνει αυτό σε επίπεδο πολιτικό. Και θα συνεχίσουμε βέβαια τις προσπάθειές μας. Όσον αφορά δε αυτές τις ε, ε, πλεονάζουσες δηλώσεις ε, πέρασαν χρόνια για να μπορέσει η Διεθνής Οργάνωση να καταφέρει το ε, περιορισμό των αλλιευμάτων και αυτό μόνο κατά 10%. Άρα είναι ισχνές, ισχνά τα αποτελέσματα. Για την επανεξαγωγή των αλλιευμάτων πρέπει να σας πω ότι κάποια από αυτά ίσως επανεξάγονται αλλά κάποια άλλα από το, από το κύριο σκάφος, το πνητικό, φεύγουν κατευθείαν για τα ευρωπαϊκά κράτη. Κάποια άλλα γυρνάνε στην Κίνα και επανεξάγονται ίσως ως ε, κινέζικα ψάρια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν είναι λευκό ψάρι, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να αναμειχθεί με ψάρια από τη Ρωσία, από την Ινδονησία. Δεν υπάρχει τρόπος ανείχνευσης. Ο πρόεδρος. Η κυρία Καραμπάγιο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για το έργο σας, συγχαίρω μάλλον για το έργο σας αυτό. Πρόκειται για δύσκολο έργο, επειδή πρέπει να, είναι, να υπάρχει και δημοκρατία για να μπορεί κανείς να φέρει σε πέρα αυτή τη μελέτη υπό αυτές τις συνθήκες. Λοιπόν, για τον καθεσμό όλων αυτών των πρακτικών, εγώ Ξέρω ότι αποφασίσαμε εδώ και καιρό ότι για την Κίνα υπάρχουν κάποιοι εμπορικοί, οικονομικοί κανόνες διαφορετικοί. Ε, δεν με εκπλήσει λοιπόν αυτό που βλέπω. Είμαστε πολύ απαιτητικοί και καλά κάνουμε και με τις δικές μας χώρες και με άλλες τρίτες χώρες και συζητάμε τη διατήρηση των πόρων μας. Να όμως ε, από την άλλη πλευρά η αντίφαση και το μεγάλο παράδοξο. Πόσο δύσκολο δηλαδή μπορεί να είναι μέχρι και να έχει κανείς πρόσβαση στα στοιχεία για την Κίνα. Μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε εσείς, ότι πέραν του ότι τους ζητείτε να δώσουν στοιχεία για τα πραγματικά λεύματα. το πώς, πότε και πού. Α, πλήρη συχνηλασιμότητα. Γιατί έτσι θα έχει εγγύσεις και θα νιώθει ασφαλής και ο καταναλωτής ε, αλλά θα καταπολεμήσουμε αυτόν τον τρόπο αυτό και την πά. Επειδή μιλάμε όμως για μια τρίτη χώρα, αυτή η χώρα δεν δίνει πληροφορίες, αρνείται να δώσει πληροφορίες, εσείς προτείνετε κάποια μέτρα, όχι μόνο κυρώσεις, αλλά και ποινικού χαρακτήρα μέτρα. Εγώ συμφωνώ με την αρχή αυτή γιατί δυσκολευόμαστε μέχρι και στοιχεία να συλλέξουμε. Γι' αυτό σας ερωτώ, με ποιο μηχανισμό εσείς νομίζετε ότι μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Με δικαστικό τρόπο. Γιατί όλοι είναι όλο και πιο λίγο ευέλικτοι. Είπατε για τις επιχειρήσεις επίσης ότι δεν μπορεί να ελέγξει, ότι περνάνε, τέλο πάντων, με ένα περίεργο μου φαίνεται η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας να μην έχει μηχανισμούς ελέγχου για τις μεταφορές ε, μεταξύ επιχειρήσεων. Αυτό είπατε όμως. Και τελευταίο ερώτημα. Είπατε ότι θα είναι σημαντικό να υπάρχει ένα κέντρο ερευνητικό, ένα μέσο έρευνα ε, μόνιμο, για να μπορούμε τέλος πάντων να συγκεντρώνουμε αυτά τα δεδομένα. Αυτός ο ρόλος αυτό θα μπορούσε το ρόλο να διδαρματίσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ελέγχου Αλίας. Μας μίλησαν το πρωί για το ψηφιοποιημένο αυτό σύστημα που μπορεί να εντοπίζει που βρίσκονται σκάφη, που αλλιεύουν κτλ. Αυτό λοιπόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την ε, παράνομη αλία και δυστυχώς ε, για λόγους εξοικονόμησης διαγράφηκε ένα κονδυλί από τον περιπλωσμό του 12. Δεν ξέρουμε πώς γίνεται το και για το 13. Σε αυτό το πλανήτη όπου όλοι ε, κατοικούμε ε, δεν μπορούμε να ανεχόμαστε να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία ε, λέει μόνο μεγάλα και ωραία λόγια. Απάντηση. Ακούστε, η Κίνα αρχίζει τώρα να μπαίνει ουσιαστικά στο διεθνές προσκήνιο. Έχουν γίνει διάφορες ε, μελέτες από ανθρώπους που προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν. Και ίσως έτσι πιστεί η Κίνα να δεσμευτεί τέλο πάντων. Το θέμα είναι ότι αν δεν γνωρίζουμε αυτά που κάνουν, δεν γνωρίζουμε τίποτα για αυτά που κάνουν, δεν χρειάζεται και αυτοί να πούν τίποτα για όσα κάνουν. Αν λοιπόν όπως, προτείνω, όπως προτείνουμε τέλος πάντων, υπήρχε μια ομάδα Ευρωπαίων Επιστημών ακαδημαϊκών με βαθιά γνώση στα αλλιευτικά ζητήματα που θα μπορούσε να τους ε, στριμώξει κατά κάποιο τρόπο, τα ψέματα που, πάνω στα οποία βασίζονται σε κάποιες περιπτώσεις δεν θα μπορούν να τα συνεχίσουν. Αυτή τη στιγμή τα καταφέρνουν γιατί κανείς δεν μπορεί να προσβάλλει αυτά που λένε. Είναι όμως δυνατόν να γίνει αυτό. Για να σας δώσω ίσως το καλύτερο κατά παράδειγμα. Δηλαδή την ε, εκστρατεία για τα πτερίγια των καρχαριών. Πριν από πέντε χρόνια φαινόταν δεν θα άλλαζε ποτέ αυτό. Πριν από μια εβδομάδα, φαντάζομαι θα το ακούσατε, νομίζω ότι ήταν η Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος, ε, το πάντων υψηλό όργανο του κόμματος, αποφάσισε ότι η σούπα από πτερήγια καρχαρία πάβει πλέον να σερβίρεται επισήμω. Και αυτό είναι ένα τρομακτικό βήμα προς τα εμπρός, διότι όχι μόνο πρακτικά θα μειωθεί η ζήτηση, αλλά δέχτηκε η χώρα ότι είναι θεμητό το αίτημα αυτό που ζητούν να σταματήσει αυτή η πρακτική και είναι ένα τεράστιο βήμα αυτό. Νομίζω ότι αυτό που εμείς έχουμε ζητήσει, δηλαδή διαφάνεια, τήρηση των κανόνων, επισήμανση προέλευσης, διαφάνεια, παραλαμβάνω, είναι σημαντικά. Γιατί, ε, όπως είπατε όλοι μας από τον πλανήτη, πρέπει όμως ε, και εμείς να δίνουμε ένα καλό παράδειγμα και να τους ε, να συναλλασσόμαστε, αν θέλετε, μαζί τους με αποτελεσματικότητα. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε, να διαβάζουμε, να μαθαίνουμε τι κάνουν και έτσι να αποκρούουμε αυτά που κάνουν, έχοντας όμως πλήρη γνώση της κατάστασης. Αυτή λοιπόν η νίκη στο θέμα των πτερυγίων του Καρχαρία είναι σημαντικό γιατί πριν από πέντε χρόνια μας λέγανε είστε ρατσιστές. Αυτή είναι η δική μας κουλτούρα, αυτό είναι ο πολιτισμός. Όμως καταγάγαμε νίκη σε αυτό το θέμα. Πλέον δεν σερβίρεται σούπα με πτεριγιά Καρχαρία στην Κίνα. Και βλέπουμε ότι τελικά έχουν μία αντίσταση ε, και είναι θέμα αρχής μόνο σε, σε ό,τι λέμε. Ευχαριστώ πολύ κύριο Σκούν, έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ πολύ κύριε Παόλη για την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση σας. Αξιοσημείωτο βεβαίω είναι ότι έχετε και την απευθείας ε, συνεργασία με την ε, οργάνωση τροφίμων και γεωργίας στην FAO και δώσατε απευθεία στοιχεία και συγκρίνατε στοιχεία. Είναι χώρα αναβιώμενη η Κίνα με πάνω από ένα δισεκατομμύριο κατοίκους. Άρα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι και η εξασφάλιση των διατρεφικών αναγκών του ίδιου του πληθυσμού πρέπει να αποτελεί μια προτεραιότητα για τη χώρα αυτή. Επίσης, τα μικρά αλληλευτικά σκάφη ε, ίσως είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθούν συνδέτη στην ε, αποκλειστική οικονομική ζώνη. Δεν νομίζω ότι θα έχει τέτοια συστήματα όπως εμείς στην Ευρώπη, αλλά είναι μέλος της IMO, της Διεθνούς οργάνωσης ναυτιλίας. Επομένως, θα πρέπει σε αυτό το επίπεδο να εκτελεί, να επιτελεί τις υποχρεώσεις της. Και άρα πρέπει να υπάρχουν ε, τα στοιχεία για το μέγεθος, το φορτίο, την ε, χωρητικότητα και όλα αυτά μέσω του αυτόματου συστήματος των αντακλαστήρων που έχουν τα πλοία πάνω τους και μεταδίδουν τα στοιχεία. Άρα Πρέπει αυτό, αυτή η υποχρέωση να λειτουργεί. Πρέπει να υπάρχουν επίσης άλλε διεθνεί συμβάσεις ενδεχομένω που θα υποχρεούνται να τηρούν. Και φαντάζομαι ότι σε διεθνή ύδατα όπου πολλά σκάφη διαφορετικών κρατών τηρούν κάπως χαλαρά τις διεθνείς ε, προϋποθέσεις και συμβάσεις, ίσως είναι πιο δύσκολο να ελεγχθεί η, δράση αυτών των κινέζικων σκαφών. Από την άλλη η Ευρώπη έχει 500 εκατομμύρια κατοίκους και ανάγκη για 8 εκατομμύρια τόνους προϊόντων ηχθείων και ηχθείς. Με 3 εκατομμύρια είμαστε εμείς, ε, έχουμε τη δική μας παραγωγή, έχουμε και περίπου 800.000 τόνους 800.000 ε, ε, κιλά ηχθειοκαλλιέργειες, ε, αλλά αναγκαστικά θα εισαγάγουμε και από την Κίνα. Και εκεί πέρα είναι που θα δούμε τι είδου διαφοροποίηση θα γίνει, τι είδου διαφοροποίηση θα επιλέξει δική μα η αλία, ο αλληλευτικό στόλο, τι είδου νέο εξοπλισμό, τι ελέγχου ποιότητα, ε, βαρέων μετάλλων, ανείχνευση κ.ο.κ. Ε, αυτό μπορούμε στα εσωτερικά, στη δική μα παραγωγή να ελέγξουμε ή οφείλουμε να ελέγξουμε στα δε εισαγόμενα προϊόντα θα πρέπει ίσως να αναλάβουμε τον κίνδυνο ή να παραδεχθούμε ότι και εμείς δεν είμαστε τόσο αυστηροί στους ελέγχους στους δικούς μας. Απάντηση. Πρέπει να πω ότι η Ευρώπη ναι, ίσως να μην μπορεί να επηρεάσει τα όσα κάνουν ε, οι Κινέζοι στην αποκλειστική τους οικονομική ζώνη. Αλλά, μόνο να ενθαρρύνουμε μπορούμε δηλαδή, αλλά είπατε κι εσείς άλλωστε ότι η αλία στην ανοιχτή θάλασσα κάθε, με κάθε σκάφος έξω από την ε, αποκλειστική οικονομική ζώνη να ονομάζεται αλλοί ανοιχτή θαλάσσης, αλλά δεν αλλιεύουν σε ανοιχτή θάλασσα, αλλιεύουν στην ε, αποκλειστική οικονομική ζώνη άλλων κρατών. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε μια διαφορετική αντίληψη ε, και εσφαλμένη βέβαια αντίληψη και έτσι από ό,τι φαίνεται ο, ο, όρος που χρησιμοποιούν στα Κινέζικα είναι ε, αλλοί θαλάσσης ή υπερπόντια αλία, κάπω έτσι. Επομένω, ε, δεν διαφοροποιούν ω προς την, την αποκλειστική οικονομική ζώνη άλλου κράτου. Πάντως ε, αυτό που κάνουν οι Κινέζοι και σε αντίθεση με του Ταϊβανέζου είναι ότι αλλιεύουν μέσα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη άλλων κρατών. Και εσείς και η κυρία δίπλα σα νωρίτερα αναφέρθηκε ε, στην υποχρέωση των Κινέζων, στην ανάγκη για τους Κινέζους να σέβονται και να τηρούν κανόνους. Έχουν δεσμεύσει στη διεθνή κοινότητα, αλλά μόνο τα τελευταία 20 χρόνια. Θα μάθουν να το κάνουν, αναγκαστικά θα μάθουν να το κάνουν, να σέβονται δηλαδή τους κανόνες. Είναι σε διαδικασία εκμάθησης, μαθαίνουν σιγά σιγά. Ανάλογα βέβαια και με τις αντιστάσεις, ανάλογα και με τα καλά παραδείγματα που μπορούν να δουν και στο βαθμό που και άλλες χώρες διαπράττουν το ίδιο, δηλαδή αλλάζουν σημαίες, έχουν παρανομία, δηλωτή αλληλεία και το καθεξής, μπορούν να υποκρύπτονται οι Κινέζοι πίσω από αυτό, δηλαδή να λένε «Α, και εσείς το κάνατε έτσι». Επίσης, θα πρέπει εμείς στην Ευρώπη να έχουμε όσο το δυνατόν πιο τίμια και καθαρή συμπεριφορά, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να πιέσουμε τους άλλους να μας ακολουθήσουν. Και το άλλο είναι ότι όταν είπαμε ότι οι Κινέζοι με δυσκολία μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των ε, βρεφικών τροφών, να είναι καθαρά δηλαδή και όχι ε, μείγματα με επικίνδυνες ουσίες ή αντικείμενα. Ε, αυτό είναι δικό τους πρόβλημα, αν δεν τηρούν τις δικές τους προδιαγραφές ασφαλείας, αλλά αυτό το πρόβλημα το έχουμε και σε σχέση με άλλες χώρες. Θα σας υπενθυμίσω κάτι ψάρια από την Τανζανία που είχαν τύχει Επεξεργασία με εντομοκτόνο και άλλα αντίστοιχα. Και βέβαια περιπτώσει, χωρί να θέλω εγώ να κάνω διδάγματα σε κανέναν, θα πρότεινα η Κίνα να αντιμετωπιστεί όπω κάθε άλλη χώρα. Αυτοί μπορεί να θεωρούν ότι του αξίζει μια διαφορετική μεταχείριση γιατί είναι διαφορετική. Ε, όχι, δεν είναι διαφορετική. Έχουν ενταχθεί, μόλι πριν από 20 χρόνια εντάχθηκαν στην διεθνή κοινότητα και έτσι πρέπει οι ίδιες προδιαγραφές να ισχύουν και για αυτούς όπως για οπουδήποτε άλλο. Αυτό μακροπρόθεσμα θα είναι και το επιχείρημα το οποίο θα φέρει τα αποτελέσματα του. Γιατί αυτό είναι και το σωστό. Είναι το σωστό να κάνει ο καθένας τη δουλειά ε, και να, επιτελεί, να εκπληρεί τις υποχρεώσεις του όπως απαιτείται για τον κάθε άλλον. Η κυρία Ρόντου, ευχαριστώ πολύ σύντομα. Πρέπει να πω ότι με εντυπωσίασαν πολύ αυτά που είπατε. Είχα πολλά διαβάσει ήδη, αλλά με εντυπωσιάζουν, εντυπωσιάζονται συγκεκριμένα αυτά που ακόμα απτά. Θα ήθελα να αναφερθώ λοιπόν στην ε, παράνομη αλία και τη δήλωση, ε, τη τελευταία σας φράση συγκεκριμένα, ότι θα πρέπει να μετατραπεί σε ποινικό αδίκημα επιτέλους η λαθρέα αλία. Πώς θα το ορίσουμε αυτό, εάν έχουμε ένα σκάφος αλληλευτικό ε, κινέζικο στο, παράνομη αλία στην ίδια την Κίνα, τι είδους κυρώσεις προβλέπονται. Είπα και κάποιο συνάδελφο σήμερα το πρωί ότι έχουμε την ε, υπηρεσία ελέγχου που θα μας δώσει κάποιες ε, προτάσεις για την αντιμετώπιση των ε, αρκετών μάλλον πλήστων ίσως περιπτώσεων λαθρέας ε, αλίας, έτσι ώστε να δώσουμε πια ένα τέλος σε αυτή την ε, παρανομία. Είπατε ότι έχουν ενταχθεί οι Κινέζοι εδώ και 20 χρόνια στην κοινωνία των εθνών, στη διεθνή κοινότητα και ακόμα δεν έχουν μάθει και χρειάζεται να σου δοθεί περισσότερο χρόνος για να μάθουν. Εντάξει, αλλά ε, πόσο καιρό ακόμα θα χρειαστούν, Στη τελευταία ανάλυση, πόσο περιθώριο έχουμε ακόμα πριν να δέσουν θάλασσές μας. Απάντηση. Αν σας γυρίσω πίσω στο χάρτη και σας δείξω τη Βόρεια Χαβάη, εδώ έχουμε τις Ηνωμένε Πολιτείες, έτσι, πώς μπορούν να πάνε οι Κινέζοι να αλλιεύουν στις ε, Ηνωμένε Πολιτείε. παράνομα μόνο. Τι κάνουν λοιπόν, πάνε τα σκάφη τους, μιλούσα γερμανικά τόση ώρα, α, με συγχωρείτε. Ας γυρίσω στα αγγλικά. Λοιπόν, κατάσχονται τα σκάφη. Κατάσχεται το σκάφος από τις Αμερικανικές Αρχές, συνήθως αυτό συμβαίνει. Πλην όμως Και αυτό δεν αφορά μόνο τα κινέζικα σκάφη. Είναι τόσο εποφελής η αλληλεία, επί παραδείγματι στην Ανταρκτική, που κάποιοι αλληλευτικοί στόχοι και ευρωπαϊκών κρατών έχουν πέντε σκάφη και όταν ε, λαθραλιεύουν και έρχεται ένα ε, σκάφος ε, της αυτοφυλακής, λιμενικό κτλ θυσιάζεται ένα σκάφο. θυσιάζεται μέχρι όχι μόνο κατάσταση, μέχρι και βήθηση. για να μπορέσουν τα υπόλοιπα 4-5 να συνεχίσουν να αλλιεύουν. Ε, έτσι λοιπόν ε, είναι τόσο υποφελή αυτή η αλλία που είναι διαδεδομένη πρακτική. Χωρί να θέλω να σα κάνω ε, προπαγάνδα υπέρ των Κινέζων, είναι έτσι τα πράγματα. Είναι κάτι το οποίο πράττουν, διαπράττουν και σκάφη άλλων κρατών. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να κάνει η Κίνα η Ευρώπη συγγνώμη, είναι να είναι εκείνη άμεμπτη στη συμπεριφορά της, ώστε να μπορεί από θέση ηθικής υπεροχής να πει κοιτάξτε εμείς το κάνουμε, πρέπει και εσείς, οφείλετε και εσείς να τηρείτε τους κανόνες. Όταν είναι κανείς ε, βουτυγμένος με στη λάσπη, μόνο μαζί με τους άλλους που βουτάνε στη λάσπη μπορεί να διαπραγματεύεται. Και αυτό πιστεύω σε ένα βαθμό είναι αυτό που συμβαίνει. Υπάρχουν πολλοί στόλοι στην Αρκτική και πολλοί από αυτούς ή όλοι από αυτούς ε, προβαίνουν σε λαθραλίευση. Οι Κινέζοι έχουν μεγάλο μερίδιο στη λαθραλία εκεί και στην Αφρική, αλλά δεν ήταν αυτοί που ξεκίνησαν την ε, λαθραλία. Άρα λοιπόν η μεταρρύθμιση που θα πρέπει να υλοποιηθεί θα πρέπει να συμπεριλάβει και τις άλλες χώρες. Εάν μπορούν δηλαδή καλύτερα να οργανωθούν οι χώρες ε, στον οποίο την αποκλειστική οικονομική ζώνη αλλιεύουν ε, οι Κινέζοι αλλά και οι άλλοι και να μπορούν έτσι να αμυνθούν καλύτερα, να αμυνθούν κατά των ευρωπαϊκών αλλά και κατά των κινέζικων σκαφών, τότε νομίζω θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Και είναι μεγάλη χώρα. Ό,τι και να κάνουν, μεγάλη κλίμακα θα έχει. Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε ότι αφήνουν ένα τόσο μεγάλο αποτύπωμα από μια τέτοια δραστηριότητα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο το πράττουν, ε, νομίζω ότι θα θυμηθείτε την ε, Ιαπωνία ή την Ταϊβάν πριν από 20 χρόνια ή ε, και την Ισπανία ακόμη θα έλεγα πριν από μερικά χρόνια. Ίσως, ίσως, ίσως. Πριν από μερικά χρόνια. Ευχαριστώ κύριο Σάντσες Πρισέδο. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ένα από τα συμπεράσματα της έκθεσης είναι ότι μάλλον έχει φτάσει στα όρια κατανάλωσης η Κίνα, στα όρια κατακεφαλήν κατανάλωσης. Σας έλεγα λοιπόν ότι ένα από τα συμπεράσματα της έκθεσης είναι ότι η Κίνα έχει φτάσει στο όριο της ε, κατακεφαλήν κατανάλωσης, υπερβαίνει δηλαδή ε, την κατακεφαλήν κατανάλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι είδους κατανάλωσης καλύπτεται από την αλία από τον Κινέζικο στόλο και τι ε, ποσοστό αντιστοιχεί στις εισαγωγές και τι δυνατότητα. Κάτι είπατε για τα δύο τρίτα και κάτι άλλο. Στην Αφρική. Η Αφρική είναι το 70% των αλευμάτων εκτός κινέζικων χωρικών υδάτων. Στο παράδειγμα 2 όμως η σχέση των διεθνών συμφωνιών της ΦΑΟ δεν αναφέρει, μάλλον εκεί στον κατάλογο αυτό δεν αναφέρει καμία αφρικανική χώρα. Εκτός από τη Μαυρτώνια, μια δημόσια ε, κρατική επιχείρηση. Τι γίνεται ακριβώς. Απάντηση. Οι κινέζικες στατιστικές για την ε, κατανάλωση ψαριών και θαλασσινών επηρεάζονται πάρα πολύ από το γεγονός ότι η Κίνα παράγει τα δύο τρίτα των προϊόντων εχθοκαλλιέργειας στον κόσμο. Δεν μπορείς λοιπόν να υπονοήσεις ότι εξαρτώνται από ψάρια ξένων χωρών, άλλων χωρών. Περισσότερο, τα περισσότερα θαλασσινά που καταναλώνται στην Κίνα προέρχονται από την ε, υδατοκαλλιέργεια είναι αυτά τα δίθυρα μαλάκια, τα μύδια και όχι δεν είναι τόσο ψάρια δηλαδή. Και όλα αυτά παράγονται από τη χθεοκαλλιέργεια, υδατοκαλλιέργεια. Είναι λάθος λοιπόν που λέγεται ότι κάθε δεύτερο ψάρι που τρώμε προέρχεται από την χθεοκαλλιέργεια. Είναι λάθος, είναι ανοησία αυτό. Τα περισσότερα είναι δίθυρα και τα περισσότερα στην Κίνα καταναλώνονται. Αυτός ο στόλος αλληλευτικός ε, μακρών αποστάσεων, περπόντιος της Κίνας, ουσιαστικά δεν θρέφει, αν θέλετε, την Κίνα. Είναι εμπορική επιχείρηση ουσιαστικά. Είπα ότι ίσως το 1 τρίτο ε, των ελληνικών εκφορτώνονται τοπικά, το 1 τρίτο σε άλλες αγορές και τα οι είδη του βυθού που αρέσουν στους ε, Κινέζους πολλούνται και καταναλώνονται στην Κίνα. Τα υψηλά λοιπόν επίπεδα κατανάλωσης δεν, ε, στην Κίνα δεν προέρχονται από ε, ψάρια τα οποία εισάγουν από άλλες χώρες. Δεν το πιστεύω αυτό. Το δεύτερο, σε ό,τι αφορά συμφωνίες πρόσβασης, τις διάφορες συνθήκες και συμφωνίες. Το ανέφερα. Οι συμφωνίες πρόσβασης, με αυτές τις συμφωνίες λειτουργεί η Κίνα, είναι απόλυτα αδιαφανής. Δεν ξέρουμε τι λένε. Ίσως υπάρχουν, μάλλον υπάρχουν, αλλά θα μπορούσε να πρόκειται για μια ανταλλαγή επιστολών μεταξύ της ε, Προεδρίας και της Πρεσβείας μιας χώρας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αυτό επαρκεί για να θεωρείται νόμιμη παρουσία της Κίνας. Αλλά δεν είναι γνωστό τίποτα, ούτε καν και στην ίδια τη χώρα για αυτές τις συμφωνίες. Πολύ επειδή έχω ζήσει στην Νοτιοανατολική Ασία ε, πολύ καιρό, 20 χρόνια περίπου, πολλές δραστηριότητες γίνονται από κινέζικες οικογένειες που ε, μάλλον πολλοί ακτιβιστές ε, διευκολύνουν κατά κάποιο τρόπο τις συμφωνίες αυτές. Είναι ιδιωτικέ. Είναι ακτιβιστές που ζουν εκεί, σε αυτές τις χώρες. Είναι ιδιωτικά συμφωνητικά λοιπόν. Και μετά έχουν ως αντιστάθμιζα κάποιον άμεσων επενδύσεων, κάποιων έργων, ε, δομη, κατασκευαστικό κτλ. Είναι κάτι που αρέσει στις ε, τρίτες χώρες αυτό, παραδείγματος χάρη ε, στην Αφρική. Άρα νόμιμη είναι η παρουσία του σε πολλές περιπτώσεις, αλλά χωρίς να το κοινοποιούν και ούτε και στην ίδια την χώρα. Όταν λοιπόν μία τράτα, ένα γρηγρή κινέζικο καταστρέφει τα παραγάδια που έχουν ρίξει, παραδείγματο χάρη, οι μικροί αλεί λένε παράνομοι, ε, λαθραλεί το κάνουν αυτό κτλ. Μα όχι, δεν είναι έτσι. Μπορεί να μην πρέπει να είναι στα 10 ή στα 5 μίλια, αλλά νομίμω ε, επιχειρούν σε αυτή, δραστηριοποιούνται οικονομικά σε αυτή τη χώρα. Τώρα βγάλτε εσείς στην άκρη. Σίγουρα είναι ένα πρόβλημα το ότι είναι τελείως αδιαφανείς σκοτεινές αυτές οι συμφωνίες. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο ε, ως τελευταίο μήτρα, αλλά για πρώτη φορά στην κυρία Τόμας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και καταρχάς ευχαριστώ πολύ για, το πολύ, για την πολύ δεξοδική αυτή παρουσία του τρόπο με τον οποίο οργανώνεται σε διεθνέ επίπεδο η ΕΛΙΕ, e τουλάχιστον θα οργανωνόταν εάν δεν είχαμε όλα αυτά τα προβλήματα. Είπατε ότι μπορεί να μην έχουν ε, απαραίτητα ε, κινέζικη σημαία, τα κινέζικα πλοία, αλλά τότε ρωτώ, Μήπως αυτό έχει στόχο όταν παίρνει παραδείγματι η σημαία Αφρικανικού κράτους. Μήπως έχει στόχο να εμφανίζονται ως Αφρικανικά κράτη και να μπαίνουν σε συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι πιο υποφελής ε, και έτσι καταφέρνουν κάτι που θα κατάφεραν εάν είχαν την Κινέζικη σημαία ή υπάρχει άλλος λόγος ενδεχομένω. Δεύτερη ερώτηση. Γιατί να μην έχουν δηλαδή σημαία Κίνας. Στο χάρτη σας που είναι πολύ ενδιαφέρον αλλά και πάρα πολύ ανησυχητικό σας προς την εικόνα που μας δείχνει. Βλέπουμε ότι ο Βόρειος Ατλαντικός είναι η μόνη ζώνη η οποία φαίνεται να μην έχει εκτεθεί σε αυτές τις πρακτικές, είναι απαλλαγμένη από τέτοιου πρακτικές. Πώς το εξηγείτε αυτό. Ευχαριστώ πολύ σύντομα κύριε Πόλη. Απάντηση. Δεν ε, γνωρίζω τόσο το δημόσιο διεθνές δίκαιο στο να σας απαντήσω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το θέμα της σημαίας ευκαιρίας. Και δεν νομίζω τι αποτέλεσμα θα είχε. Τι συνέπεια θα είχε το να υψώσει σημαία κάποιου άλλου κράτους ε, ένα πλοίο. Δεν γνωρίζω. Α, αν αυτό μπορούσε να οδηγήσει περισσότερη διαφάνεια, τι να σας πω. Αλλά δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω, πρέπει να μου λες ότι δεν το γνωρίζω. Τι ήταν η άλλη σας ερώτηση τώρα. Βόρειος Ατλαντικός. Ναι, γιατί ο Βόρειος Ατλαντικός. Τι να σας πω, εάν εμφανιζόταν κανείς για να πει χαίρετε, ήρθαμε να ψηφίσουμε στην Καντάμπρια ή στην Σκοτία. Ε, φαντάζομαι ότι θα υπήρξαν αυτά, υπήρχαν αντιδράσεις. Υποθέτω ότι η Κίνα όταν ξεκινάει να αναπτύσσει δραστηριότητε κοντά σε μια χώρα, κάτι τη προσφέρει. Ε, στου Ισλανδού λοιπόν φαίνεται ότι δεν έκαναν προσφορά. Δεν το αποκλείω όμω, μπορεί και να συμβεί. Είπατε δεν θεωρείτε ότι αυτός είναι ο λόγος. Ε, δεν ξέρω. Εγώ δεν, δεν περίμενα ότι θα πήγαιναν να ψαρέψουν στην ε, Βόρεια Θάλασσα. Ξέρετε ότι όταν ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρχαν χώρες οι οποίες δεν δικαιούνται να ψαρέψουν, να αλλιεύουν στη Βόρεια Θάλασσα. Και η Νορβηγία σε μεγάλο βαθμό γι' αυτό απέρριψε την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ήθελε να αλλιεύουν ε, ευρωπαϊκά σκάφη στα δικά της ύδατα. Επομένως κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει τις αντιδράσεις φαντάζομαι που θα παθαίνατε πανικό όλοι, συλλήβδιν. Υπήρξε περίπτωση όπου ένα κινέζικο σκάφος πήγε στο Σουέζ και εμφανίστηκε με σημαία Γαλλία και υπήρξε τέτοια αντίδραση από τον τύπο και γενικά την κοινή γνώμη που αναγκάστηκε να κινητοποιηθεί πολεμικό σκάφο τη Γαλλία. Ε, με τη Μαυριτανία φαντάζομαι ότι κάποιες κάποια ανταλλάγματα θα έχουν δώσει. Αλλά καθώ περνάνε πιο πολύ στο Ιναλία τόνου, γιατί προ το παρόν δεν αλλιεύουν τόσο πολύ τόνο, οι Ταϊβανοί είναι αυτοί οι οποίοι ψαρεύουν τόνο, ε, φαντάζομαι ότι θα μετακινηθούν προ την Καραϊβική. Ευχαριστώ πολύ ε, τον κύριο Παουλή και όλους τους συντάκτες αυτής της ε, μελέτης. Να σας αποχαιρετήσουμε αυτή τη στιγμή. Ας περάσουμε τώρα στην έκθεση του κυρίου Ριβελίνη, Γενικός Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Οικονομία του 2013, τροπολογίες ως τις 16 Ιουλίου το μεσημέρι. Τώρα θα ε, κάνουμε μία παρουσίαση. Ο κύριος Ριβελίνη έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα σας παρουσιάσω σήμερα μία ε, έκθεση, ένα έγγραφο εργασία μάλλον, που ε, αναπτύσσεται σε τρία σκέλη. Πρώτα απ' όλα θα μιλήσω για τον ε, σκοπό αυτή τη πρόταση. Στο δεύτερο σκέλο θα μιλήσω για την πρόταση προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι τροποποιήσει που θα πρέπει να γίνουν σε κάποιες συγκεκριμένε γραμμές προπολογισμού, στο κεφάλαιο Αλίας. Τέλος, θα κάνουμε μια ανάλυση των πιλωτικών project που παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή μας και μια πρώτη αξιολόγηση του. Σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό 2013, ω εισηγητή, τοποθετούμε προτείνοντα ε, συγκεκριμένε προτάσεις που αφορούν ε, τις ε, πιστώσεις για το κεφάλαιο αλληλεία, θεωρώντα ότι οι γενικέ γραμμές Συμφωνώ με την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά πιο συγκεκριμένα επιθυμώ την αύξηση των ε, πιστώσεων για κάποιες γραμμές, τουλάχιστον στο ύψος του προπολογισμού του 2012. Αν μάλιστα είναι αληθέ ότι η πρόταση Επιτροπή ε, συνδέεται και εντάσσεται στα πλαίσια τη ε, γενικότερη οικονομική κρίση, ταυτόχρονα είναι αληθέ ότι εντάσσεται και σε ένα πλαίσιο τέλος ε, δημοσιονομικών οπτικών και παρότι από τη μία είναι λογικό να έχουν μειωθεί ε, κάποιοι πόροι ε, για τους οποίους υπάρχει ανάληψη υποχρεώσεων για το κεφάλαιο 11, αλλήλεια δηλαδή, σε άλλες γραμμές όμως του προπολογισμού που αφορούν την διατήρηση των πόρων Θεωρούμε ότι οι μειώσει είναι απαράδεκτε γιατί ουσιαστικά επιβάλλουν κυρώσει στον τομέα τη ελληνία και αλληλευτικέ θαλάσσιε υποθέσει. Διότι πρόκειται για μια πολιτική πολύ σημαντική για την ισορροπία στι επιμέρου περιοχέ, για την διασφάλιση των οικοσυστημάτων και την οικονομική κατάσταση όπω ορίζονται στου στόχου τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Επίσης, ε, το σχέδιο προπολογισμού, όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν λαμβάνει υπόψη την προσχώρηση μιας άλλης παράκτιας χώρας, της Κροατίας. Άρα, είναι οπωσδήποτε αναγκαίο να διορθωθεί ο προπολογισμό εν το χρόνο, ώστε να προβλεφθούν οι απαραίτητες, ε, απαραίτητοι πόροι για ε, μια χώρα νεοεισερχόμενη, αλλά και να εγγυηθούμε και τους ε, ήδη πόρους για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Προτείνουμε λοιπόν κάποιε αυξήσει σε σχέση με τα επικαιροποιημένα στοιχεία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα θα πω σε κάποιε λεπτομέρειε. Στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώ χρονοσκόπιμο, να αυξηθούν και οι πιστώσει ανάληψη υποχρεώσεων και πληρωμέ στι εξή γραμμέ. Διακυβέρνηση τη κοινή πολιτική αλεία, γραμμή προπολογισμού 11, 0401. Ε, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει 5.390 εκατομμύρια για την ανάληψη υποχρεώσεων και άρα μία μείωση κατά 15,8% σε σχέση με τον προπολογισμό του 2012. Ενώ για τις πληρωμές προτείνει 4.868.000 δηλαδή μία μείωση κατά 13% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Λαμβάνοντα υπόψη τη σημασία των δραστηριοτήτων που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη γραμμή του προπολογισμού, προτείνουμε οι πιστώσει ανάπτυξη προχρεώσεων να φτάσουν τουλάχιστον το επίπεδο του 2012 και σε ό,τι αφορά τις πληρωμές, επαναλαμβάνω για τι πληρωμές, μιλώ, είναι σκόπιμη μία αύξηση κατά 16% σε σχέση με την πρώτη της Ευρωπαϊκής ώστε ε, πληρωμές, μιλώ για πληρωμές για άρα δεσμές που έχουν ήδη αναλυφθεί, ε, που να φτάνουν ε, στο ύψος της προηγούμενης χρονιάς. Σε ό,τι αφορά τώρα την ε, προστασία των θαλάσσιων πόρων, γραμμή προπολογισμού 11.0701, η Κομισιόν προτείνει μία μείωση κατά 3,2% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά σε ό,τι αφορά τις πιστώσεις ανάπτυξης προσώσεων περνώντας από τα 46,5 εκατομμύρια ευρώ στα 46 εκατομμύρια. 7,3% λιγότερο σε ό,τι αφορά τις πληρωμές που περνούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 38 εκατομμύρια, περίπου εκατομμύρια σε 35 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Και για αυτή τη γραμμή και λόγω της σημασίας που έχει είναι πολύ σημαντικό αντί για μείωση να προβλέψουμε μια αύξηση τουλάχιστον κατά 4% το ύψος αυτών των πληρωμών σε σχέση με το 2012 ώστε να καταλήξουμε σε ανάληψη υποχρεώσεων που να φτάνουν τα 48 εκατομμύρια ευρώ και πληρωμές που να φτάνουν τα 37 εκατομμύρια ευρώ. Σε ό,τι αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ελέγχου της Αλίας, η γραμμή του προπολογισμού 11.08.05.01 και για τη γραμμή του προπολογισμού 11.08.05.02 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μία μείωση κατά 0,4% σε σχέση με το 2012 σε ό,τι αφορά ε, τις πιστώσεις ανάπτυξης υποχρεώσεων και πληρωμών και σε ό,τι αφορά τη γραμμή 11.08.05.01 που αντιστοιχεί στις διοικητικές δαπάνες του οργανισμού ορίζει μία χρηματοδότηση 7.311.395 ευρώ ενώ σε ό,τι αφορά τις πληρωμές που ανέρχονταν πέρυσι στα 7 εκατομμύρια 370 ε, περίπου χιλιάδες ευρώ, η Επιτροπή προτείνει μία μείωση κατά 0,4%. Επίσης, σε ό,τι αφορά την άλλη γραμμή, την 11.08.05.02, που αντιστοιχεί στις δράσεις που αναλαμβάνει ο οργανισμός, η Κομισιόν μειώνει τα ποσά κατά 4,2% σε σχέση με πέρυσι, σε ό,τι αφορά την ανάληψη υποχρεώσεων και μειώνει τις πληρωμές από 39,8 κατά μάλλον 39,8% ώστε να φτάσουν από 2.600.000 σε 1.600 μόλις. Η σημασία αυτού του οργανισμού είναι πραγματικά μεγάλη και το έργο της, ε, οργανισμού αυτού είναι απαραίτητος για τον αλληλευτικό κλάδο. λοιπόν απαράδεκτες αυτές τις προτάσεις και εντελώς δυσανάλογες και γι' αυτό προτείνω να ε, φτάσουν οι ε, ανάληψεις υποχρέωσης στα 7,5 εκατομμύρια και οι πληρωμές για την πρώτη γραμμή του προπλογισμού και στα 1,7 ε, εκατομμύρια σε ό,τι αφορά τη δεύτερη γραμμή για τον οργανισμό σχετικά με τις πληρωμές η εξοικονόμηση και η λιτότητα σε εποχή κρίσης είναι κάτι κατανοητό, αλλά όχι με τόσο υπερβολικό τρόπο ε, σε τέτοια κεφάλαια. Αυτά τα τεχνικά στοιχεία είναι δυσνόητα, είναι ακατανόητα μάλλον και η γραμματεία θα σας δώσει, αν όχι σήμερα, αύριο τους ακριβείς πίνακες για να μπορέσετε να τους μελετήσετε. Πίνακες που μόλις και εγώ έλαβα. Να τελειώσω με τα πιλωτικά project για την Αλία και να περάσω στην ανάλυση των πιλωτικών project που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια πρώτη ε, αποτίμηση σκοπιμότητας. Δυστυχώς μόλις ένα πιλωτικό project έλαβε μία κατάλληλη χρηματοδότηση, άρα να εφαρμοστεί άμεσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. το project αυτό έχει ως ε, τίτλο θεματοφύλακε τη θάλασσα. οποιοδήποτε λοιπόν θέλει να εφαρμόσει αυτό το project θα μπορέσει να έρθει σε επαφή με το γραφείο μου. Τα άλλα πυροδικά project που παρουσίασαν ε, οι λοιποί συνάδελφοι της Επιτροπής αξιολογήθηκαν αρνητικά από την Κομισιόν εκτός από ένα, αυτό του ε, κυρίου Φεραίρα με τίτλο για τη δημιουργία μιας ε, δημόσιας ασφάλειας για τις ε, απρόβλεπτες συνθήκες στην Αλία που αξιολογήθηκε με βαθμό Β και άρα λοιπόν μπορεί να τύχει επανεξέταση. Η γραμματή της Επιτροπής μας, αμέσως μετά από αυτή τη συνάντηση, θα σας αποστείλει ένα email με το έντυπο που πρέπει να συμπληρώσετε ώστε επίσημος να παρουσιάσετε τα πιλωτικά project που επευλήθησαν στην Επιτροπή με τη μορφή τροπολογιών επί του προπολογισμού. Όπω είπα, Πρόεδρε, η καταλητική προθεσμία για την υποβολή αυτών των πιλωτικών project, όπω και για την παρουσίαση τροπολογιών ε, στο δικό μου κείμενο, είναι η Δευτέρα 16 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Φράγα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Ριβελίνη Έχω να κάνω κάποιες ερωτήσεις προς τον εισηγητή, κυρίως όμως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που φαντάζομαι ότι βρίσκεται εδώ και μπορεί να απαντήσει. Καταρχάς, το 11.01.01.03 για το παρατηρητήριο τιμώνα. Βλέπω ότι έχει μεγάλη μείωση, 68, κάτι της 100 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Είναι προπαρασκευαστική ενέργεια, δεν κατάλαβα, λίγη, ολοκληρώνεται, διότι εκπλήσω με το παρατηρητήριο. Είναι κάτι που πάντοτε το στήριζε το Κοινοβούλιο, έχει λειτουργήσει σχετικά καλά, γιατί έχει τόσο μεγάλες περικοπές. Σε ό,τι αφορά το 11.03, για τι προπαρασκευαστικέ ενέργειες των νέων αλληλευτικών, διεθνών αλληλευτικών οργανώσεων και άλλες μη υποχρεωτικέ ε, ε, μάλλον υποχρεώσεις σε διεθνείς κτλ. Επίσης εδώ βλέπουμε μεγάλη ε, περικοπή 23,3% ενώ το κονδύλιο αυτό έχει να κάνει με προπαρασκευαστικέ ενέργειες ε, των γνωστών περιφερειακών οργανώσεων αλλά και διεθνών ελευτικών οργανισμών που εκεί είναι παρατηρητής, ε, έχει ρόλο παρατηρητή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δεν καταλαβαίνω γιατί 23,3% λιγότερο. Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μου εξηγήσει το γιατί και το πώς. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο εισηγητής, με το 1104 για τη διακυβέρνηση Πραγματικά και αυτό είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβουμε. Η εκτέλεση ήταν καλή στη συγκεκριμένη γραμμή. Πάλι μεγάλες περικοπές. Γιατί? Τουλάχιστον να σπάσει τον προπολογισμό ε, της προηγούμενης χρονιάς. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Και συμφωνώ, γιατί και το πρωί ο διευθυντής της υπηρεσίας ελέγχου είπε ότι πρέπει να αυξηθεί κατά τουλάχιστον 500 ευρώ. Το κονδύλι που αφορά την υπηρεσία για τον του της Αλία. Μία ερώτηση προ την, τον εισηγητή. Δεν έχουμε τα τελικά στοιχεία για την πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου. Ναι, το ξέρω, το λέω. Αλλά υπάρχουν κάποια νούμερα που ακούγονται και τα οποία λίγο πολύ έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο κορεπέρ και γνωρίζουμε ότι πολλές από τις ε, γραμμές, πολλά από τα κονδύλια που αφορούν την ΑΕΑ θα μειωθούν σημαντικά και ιδίως ε, ό,τι έχει να κάνει με το ΦΕΠ. Το να έχουμε, πώς θα έχουμε τις τροπολογίες έτοιμες τη Δευτέρα όταν πρέπει να απαντήσει το προσία του προπολογισμού, ο εισηγητής ε, και για προηγούμενες περικοπές στην πρόταση του Συμβουλίου. να μην κάνουμε τσάμπα δουλειά. Φαντάζομαι ότι οι συγκεκριτές πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ασχοληθεί με το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Ας ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Τζόνσο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα έρθω στα μεμονωμένα σχόλια και θα προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματα, αλλά θα ήθελα καταρχάς να κάνω κάποια σχέδια, σχέδια για το σχέδιο γνωμοδότησης που συζητείτε αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή σας και να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, στο σχέδιο γνωμοδότησης, ε, αυτό το οποίο λέει ο εισηγητής για την Κροατία, τα στοιχεία, ε, παράγραφος 2, τα στοιχεία για την Κροατία, μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι πράγματι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προβεί σε τροπολογία για τον προπολογισμό του 2013 σε έφτατο χρόνο. Η προσχώρηση της Κροατίας ε, θα πραγματοποιηθεί μάλλον στα μέσα του 2013. Είναι πρόωρο λοιπόν τώρα να σας κάνουμε συγκεκριμένη πρόταση. Σε αυτό το πλαίσιο, να σας υπενθυμίσω ότι την προηγούμενη εβδομάδα μόλις εγκρίναμε πρόταση τροποποίησης της πρότασής μας για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο του 2014-2020 ώστε να ληφθούν υπόψη τα περί εντάξεις της κρατίας. Στην τρίτη παράγραφο της μαμοδότησης αναφέρεται ότι υπάρχει μείωση της τάξης του 2,7% του υπερπολισμού για θαλάσσια ζητήματα και για την αλία. Ουσιαστικά, αν αποκλείσουμε τις ε, διοικητικές δαπάνες, η διαφορά μεταξύ 12 και 13 είναι 1,5%. Τα στοιχεία είναι 996 εκατομμύρια ευρώ το 2012 ε, και 980 εκατομμύρια που προτείνουμε για το 2013. Εάν λάβουμε υπόψη μας ε, τον τρόπο με τον οποίο ε, έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση της αλληλευτικής πολιτικής, έχουμε γράψει όλο το ποσό στους προϋπολογισμούς του 2011 και του 2012, αν εξαιρέσουμε το ποσό για τη θαλάσσια πολιτική από τον προπολογισμό του 2012, οι προπολογισμοί μεταξύ του 2012 και του 2013 ουσιαστικά είναι ταυτόσιμη. Σε ό,τι αφορά τώρα τις πιστώσεις πληρωμών, να πω το εξής. Για τις επιχειρησιακές δαπάνες και πάλι έχουμε μια αύξηση 3,7%, όχι 3,1%. Έρχομαι τώρα στις δυο συγκεκριμένες ερωτήσεις που ετέθησαν. Φυσικά έχουμε προτείνει έναν προπολογισμό ο οποίος καταρτίστηκε σε δύσκολες ε, συνθήκες. Υπάρχει όμως νομίζω κάποια παρανόηση σε σχέση με περικοπές σε κάποιες γραμμές του προπολογισμού. Ας δούμε την περίπτωση της υπηρεσίας ελέγχου της αλίας. Οι πόροι που θα διατεθούν σύμφωνα με τη δική μας πρόταση στον οργανισμό Ελέγχου της αλίας για το 2013 θα είναι ακριβώς οι ίδιοι με αυτούς που είχαν διατεθεί στην υπηρεσία ελέγχου το 2012. Αυτό μπορεί να μην είναι προφανέ αν δει κανεί ε, τα νούμερα, να μην ε, χτυπάει στο μάτι άμεσα, γιατί όπω και όλοι οι οργανισμοί και ο Οργανισμό Ελέγχου τη Αλίας μπορεί να χρησιμοποιεί τι μη εκμεταλλευτήσει ε, πιστό των προηγουμένων ετών. Assigned revenue το λέμε στα αγγλικά αυτό. Και έτσι έχουμε κάποιε κάποιες που δεν χρησιμοποιήθηκαν από το 2011 και εγγράφονται εσ νέο, εγγράφονται στον προεπισμό του 2013 στην περίπτωση και Ξέρουμε ότι ε, λειτουργούν ε, με ταχύτητα κρουαζιέρα, αν θέλετε, όλες, όλοι οι οργανισμοί, το ίδιο και ο οργανισμός αλληλείας. Άρα, επαναλαμβάνω, πιστεύουμε το 2013 θα κάνουν το ίδιο με το 2012, άρα θα διατεθεί όλο το ποσό το οποίο προβλέπουμε. 9.216.000 ευρώ. Επαναλαμβάνω ακριβώς το ίδιο ποσό με αυτό που είχαμε διαθέσει φέτος για τον οργανισμό. Σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις που προτείνονται και τα ερωτήματα που ετέθησαν σε σχέση με το κεφάλαιο για τη διακυβέρνηση, πληροφορία και επικοινωνία. Πράγματι, να σας τονίσω σε αυτό το σημείο ότι το 2012 δεν θα εκτελεστούν όλες οι πιστώσεις, όλες τις αναλήψεις υποχρεώσεων. Για πολλούς και διαφορούς λόγους. Ο βασικός έχει να κάνει με την διαφημιστική ενημερωτική εκστρατεία για την κοινή αλληλευτική πολιτική. Ήταν πολύ μεγάλη η εκστρατεία πέρυσι. Φέτο είναι πιο ε, μικρή ε, εμβέλεια σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση δηλαδή τη κοινή αλληλευτική πολιτική. Θεωρούμε ότι αυτό είναι πιο σκόπιμο, αν ληφθεί υπόψη και το που βρισκόμαστε στην νομοθετική διαδικασία. Το 2013 λοιπόν θα έχουμε ένα παρόμοιο επίπεδο ενημερωτικών δραστηριοτήτων. Φυσικά και προσβλέπουμε στη μεταρρύθμιση την περιμένουμε με ενυπομονησία και ίσως ε, κάποιες από τις δράσεις που χρηματοδοτούνται με αυτό το κονδύλιο του προπολισμού θα πάψουν να χρηματοδοτούνται μετά τη μεταρρύθμιση. Εξαρτάται από τις ε, ενώσεις ε, που συμμετέχουν στην ΑΚΦΑ. Εκεί σκεφτόμαστε να υιοθετήσουμε έναν διαφορετικό μηχανισμό διαπραγμάτευσης, άρα δεν θα χρηματοδοτούνται. Έτσι εξηγείται η κατάσταση ό,τι αφορά τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, ό,τι αφορά τις πιστώσεις πληρωμών. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και επιφυλακτικοί. Οι πληρωμές είναι αυτό που μετράει ε, για τις χώρες, αυτό που πληρώνουν με τον προπολογισμό. Δεν πληρώνουν σαν αλήψη υποχρεώσεων. Επομένως, τι κάναμε στην προκειμένη περίπτωση. Αναλύσαμε όλες τις νομικές δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει και που θα αναλάβουμε κατά πάσα πιθανότητα εντός του 2013 και προτείναμε ένα κατάλληλο θεωρούμε ποσό ε, πιστώσεων πλήρωμων σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο διατήρηση και την πρόταση για αύξηση των ανλήψεων υποχρεώσεων. Η κατάσταση ως εξή. Κατά το παρελθόν δεν είχαμε ε, πλήρη ε, εκτέλεση του κονδυλίου. Το ποσό που προτείνουμε για το 2013 βασίζεται σε αυτό το οποίο θεωρούμε ότι ήταν ένα εύλογο ποσό με βάση τα παλαιότερα ποσοστά. Οπότε και δεν είχε αποφροφηθεί, επαναλαμβάνω. Βασιστήκαμε λοιπόν σε ανάλυση των ανλήψεων υποχρεώσεων που είναι ανοιχτέ και που θα ε, προκύψουν. Σε ό,τι αφορά τώρα το, κεφάλαιο, το διεθνές κεφάλαιο για τις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλίας. Τα ποσά για τα οποία μιλάμε εδώ στόχο έχουν να καλύψουν και το προπαρασκευαστικό έργο για τη σπόδα, αλλά και τις ε, εθελοντικές ε, συμμετοχές. Αυτό τι σημαίνει, αν θέλουμε να κάνουμε μια πληρωμή ε, σε ένα πρόγραμμα που υπερβαίνει αυτά τα οποία συνήθως καλύπτουμε με την εισφορά, τη συμμετοχή του μέλους, το βάζουμε σε αυτή τη γραμμή του προπολογισμού. Άρα το ποσό που προτείνουμε και το οποίο πράγματι είναι μειωμένο υπολογίστηκε με βάση το ότι γνωρίζουμε τι χρειαζόμαστε για το προπαρασκευαστικό έργο και έχουμε και τον σχεδιασμό μας για το είδος των ενεργειών που θέλουμε να προωθήσουμε και των δράσεων. Σε ό,τι αφορά τα πιλωτικά προγράμματα, Πολύ σωστά ο εισηγητής σας περιέγραψε την κατάσταση. Η υλοφόρη της θάλασσας είναι κάτι το οποίο δεν καλύπτεται από κάποια νομική βάση και είναι μια δραστηριότητα που θα πρέπει να την προωθήσουμε. Η θεματοφύλακε, συγγνώμη, της θάλασσας, ε, όχι χιλοφόρη. Και ε, πράγματι βαθμολογία ήταν Β. Αυτό τι σημαίνει. Ότι το πλωτικό πρόγραμμα έχει στοιχεία που θεωρούμε ότι ναι, μπορούμε να τα συνεχίσουμε, αλλά θα πρέπει να προβληματιστούμε λίγο και να τα επεξεργαστούμε καλύτερα. Ολοκληρώνοντα, ε, θα μιλήσω λίγο. Α, ναι, υπάρχει και κάτι άλλο για το παρατηρητήριο. Κυρία Φράγκα έθεσε αυτό το ερώτημα. Είπε ότι μιλάμε για μείωση ε, στην προκειμένη περίπτωση. Δεν ισχύει αυτό. Το παρατηρητήριο στον προβληματισμό του 2012 έχει ένα ποσό της τάξης των 500.000 ευρώ. Στον προϋπολογισμό του 2013 προτείνουμε 750.000 ευρώ. Εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε τα αποτελέσματα του έργου που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του πολιτικού προγράμματος. Ετοιμαζόμαστε πια να μπούμε στην παραγωγική φάση ε, της υπηρεσίας αυτής, στα πλαίσια και του Ταμείου Διαθάλασσα και την Αλία. Καλύπτεται λοιπόν από το, Ευρωπαϊκό, από το δημοσιομικό πλαίσιο. Τέλος, να σας πω πού βρισκόμαστε με το Συμβουλίο. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, είπε η κυρία Φράγκα ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία, κάποια νούμερα ε, που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο κορέπερ. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μάλλον απίθανο να αλλάξουν ε, από τώρα μέχρι τις 26 Ιουλίου, οπότε και θα εγκρίνει την ανάγνωση του προβολισμού του Συμβούλιο. Να επισημάνω όμως κάποια από αυτά τα στοιχεία που εμάς μας ανησυχούν και που θα έπρεπε νομίζω να ανησυχούν και την Επιτροπή σας. Έχουμε λοιπόν μειώσεις στις πιστώσεις πληρωμών που προβλέπονται, σημαντικές μειώσεις σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας, 30 εκατομμύρια ευρώ, όταν μιλάμε το στόχο της μετατροπής, και 5 εκατομμύρια ευρώ για το στόχο μη, μη Ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί στις εκτιμήσεις των πιστώσεων πληρωμών για άλλα κονδύλια του προπολογισμού. Το ίδιο πράξαμε και στις εκτιμήσεις των πιστώσεων πληρωμών για τις συγκεκριμένες θέσεις του προπολογισμού. Μπορώ να σας πω ότι μάλλον μπορούμε να θεωρήσουμε σίγουρο ότι αν, έχουμε, ε, αν είχαμε περικοπή ε, των 5 εκατομμύρια σε αυτό το κεφάλαιο θα μας δυσκολέψει πάρα πολύ αυτό. Δεν θα μπορούμε να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας απέναντι στα κράτη-μέλη. Το τελευταίο όμως που θέλω να αναφέρω είναι η προτινόμενη περικοπή για την υπηρεσία ελέγχου τη αλίας, που είναι μια πραγματική περικοπή. Το Συμβούλιο λοιπόν έχει ακολουθήσει μια οριζόντια πολιτική, προτείνει μείωση της άξιος του 1% για όλους τους παραδοσιακούς οργανισμούς που λειτουργούν πλήρω. 73.000 ευρώ λιγότερα λοιπόν στον προπολογισμό αυτής της υπηρεσίας. Νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι θα συμπεριληφθούν ε, στον, ε, στη θέση που θα εγκρίνει το Συμβούλιο για τον προπολογισμό στις 26 Ιουλίου. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Φράγκα νομίζω ότι θέλει να κάνει κάποια ακόμη συγκεκριμένη ερώτηση. Ναι, να κάνω μια ακόμη παρατήρηση. Σε ό,τι αφορά τον οργανισμό ελέγχου τη Αγγλία, εντάξει δεν με απασχολεί 3,3% αλλά ένας οργανισμός με νέα καθήκοντα που πρέπει να φέρει πέρα. Λογικό δεν είναι να έχει επιπλέον χρηματοδότηση. Αυτά τα νέα project που είναι μείζονος ενδιαφέροντος πρακτικά δεν θα εφαρμοστούν. Διότι αν δεν δοθεί αυτό το επιπλέον μισό εκατομμύριο ευρώ, Πώς θα γίνουν. Εντάξει, κατάλαβα ότι γενικά πρέπει να γίνουν περικοπές 1%, αλλά πρακτικά αυτό τι σημαίνει, ότι δεν θα χρηματοδοτηθούν κάποια project. Δεύτερον, γιατί στο 11.03.03 για το προπαρασκευαστικό έργο για τους διεθνείς οργανισμούς αλίας, βλέπουμε μία μείωση. Πρέπει να μας πει η Κομισιόν γιατί. πρέπει να μας το πει. Έτσι το ε, Αναλαμβάνω αυτή τη διεθνή διάσταση. Ωραία, εξηγήστε μου, με, με, με ποια εκτίμηση καταλήξετε σε αυτό το ποσό που διαφέρει τόσο πολύ από τα περσινά αντίστοιχα ποσά. Οι διεθνεί οργανισμοί, όπου έχει ρόλο παρατηρητή η Κομισιόν, δεν έχουν αλλάξει κάτι. Ρωτώ λοιπόν γιατί αυτή η μείωση και το ίδιο. Να πω ότι δεν καταλαβαίνω τι γίνεται με τη διακυβέρνηση. Ειλικρινά. Δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται. Μπορούσα σε μια τέτοια μεταρρύθμιση κοινή συλλεκτική πολιτική. Η Κομισιόν μας λέει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται από τη βάση ε, προς την κορυφή, ότι θα λαμβάνουν πιο πολύ υπόψη του περιφερειακούς οργανισμούς και όλα αυτά. Μας τα λέτε και μετά κόβετε τα κονδύλια. Ε, δεν μπορώ να το καταπιώ αυτό το πράγμα. Πρέπει να μου δώσει μια εξήγηση. Ως τώρα δεν έχω λάβει απάντηση. Και ζητώ από τον εισηγητή αυτή η γραμμή να επιμείνει να φτάσει τουλάχιστον το ύψος περσινής χρονιάς. Και τέλος, να πω ότι όσο αφορά τον ελεκτικό οργανισμό, εκεί είναι περίτρανο το, το παράδειγμα ότι η Κομισιόν δεν μπορεί να κάνει αυτές τις προτάσεις. Αν δεν έχουμε μια αύξηση τουλάχιστον μισού εκατομμυρίου για τον οργανισμό, ε, τα νέα τόσο σημαντικά project που συζητούσαμε το πρωί δεν πρόκειται να υλοποιηθούν. Ευχαριστώ τρει ακόμη αγορητέ και μετά στον κύριο Ριμπελίνδο. Στον λόγο, παρακαλώ λοιπόν να είστε σύντομοι, γιατί έχουμε ακόμη άλλα δύο σημεία και πρέπει να σταματήσουμε Στι Τόμας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή για την έκθεσή του, στην οποία απογραμμίζει πράγματι ε, την έλλειψη φιλοδοξίας τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Ε, εξού και πρώτη μου παρατήρηση για την ε, υποστήριξη της αδέλφου Φράγκα για το θέμα των ελέγχων ποτέ δεν πρόκειται να εφαρμοστεί ένα σωστό μέτρο, μάλλον να εφαρμοστεί σωστά ένα μέτρο, αν δεν υπάρχει ο κατάλληλος έλεγχος. Και ακούσαμε ότι δεν αρκούν οι πόροι, ούτε οι πολιτικές εκτελούνται, άρα η μείωση των πόρων είναι καταστροφική. Το ίδιο ισχύει και για το θέμα της διακυβέρνησης. Άλλωστε το είπε και ο εκπρόσωπος της Κυπρικής Προεδρίας προηγουμένως, ότι η προτεραιότητα είναι τα σχέδια διαχείρισης. Άρα η διακυβέρνηση που είναι κάτι σημαντικό για την ε, υλοποίηση αυτών των σχεδίων πρέπει να είναι εξίσου προτεραιότητα. Τώρα, για τους ε, ρυθμούς εκτέλεσης, ε, τα ποσοστά εκτέλεσης προηγούμενης χρονιάς. Πολλές φορές βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη ε, αποστασιοποιούνται και σταματούν κάποιες δεσμεύσεις. Και εδώ πλέον αντίθεται θέμα με την εκτέλεση, γιατί έχουν και την υποχρέωση της συγχρηματοδότησης τα κράτη-μέλη. Βλέπουμε λοιπόν ε, να μην υπάρχει αντιστοιχεία μεταξύ των επιλέξιμων και των αναγκαίων για τους φορείς και για τους κλάδους. Και τέλος, ευχαριστώ την προσοχή σας ε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αν είναι μικρός ο προβλησμός του 2013 και για το επόμενο πολιτές νομικό πλαίσιο βασιστούμε από εκεί και πέρα στο 2013, ποιες είναι οι φιλοδοξίες πλέον που έχουμε για τον πολιτικό υπολογισμό. Αν βασιστεί δηλαδή στον ίδιο αποδυναμωμένο προπολογισμό του 2013 η επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Ευχαριστώ κύριε, κυρία Ρόντου, τώρα έχει τον λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Βεβαίω, σημειώνω τόσο είπε η κυρία Φράγκα. Είναι κατάσταση σοβαρά. Πρέπει να συζητήσουμε για μια νέα μεταρρύθμιση της αλληλεία και πρέπει να το κάνουμε γιατί υπάρχει το υπεραλίευμα, γιατί υπάρχει ε, το πλεόνασμα αλληλευτική ικανότητας. Άρα, εάν θέλουμε να συζητήσουμε ε, τα προβλήματα χωρί όμω να είμαστε διατεθειμένοι να ε, περικόψουμε τους ε, προϋπολογισμούς. Πείτε μου πώς μπορούμε να ε, δείξουμε στους άλλοις ε, ότι θέλουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση στην αλληλεία αλλά δεν θα υπάρχουν αρκετά κονδύλια για να τους στηρίξουμε. Όλοι θέλουμε εξοικονομήσεις και τελικά δεν θα μπορέσουμε ποτέ να εξασφαλίσουμε καμία ε, ουσιαστική μεταρρύθμιση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καντέκ έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ πολύ στομα να πω ότι συμμερίζομαι απολύτως τόσο είπε η Κάρμεν Φράγα. Ε, δηλαδή ότι για το μελλοντικό ταμείο, αλληλευτικό ταμείο, θα πρέπει να διατεθούν προς τώρα χρήματα για τον έλεγχο, για την υπηρεσία ελέγχου. Σύντομα δεν ήτανε. Πολύ ωραία. Τέλεια, τέλεια. Μακάρι να ήταν πάντοτε έτσι. Η Επιτροπή θέλει και πάλι το λόγο. Όχι, ο κύριος Ριμπελίνη τότε. Η Κομισιόν. Ήθελα απλώς να πω ότι βεβαίως είμαστε μέσα στην ε, εξελίξη ε, δημοσιονομική διαδικασία. Η αρχή αρμόδια ε, για τον προϋπολογισμό έχει αναλάβει από την Επιτροπή την πρόταση όταν παραμένει στατικό κάτι, πρέπει να σας πω ότι και αυτό συμβαίνει τώρα με την ελευτική πολιτική, ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς δεν ε, αισθάνονται ιδιαίτερα χαρούμενοι. Αλλά πρέπει να σας πω ότι έχουμε να κάνουμε ένα εκατομμύριο ε, ευρώ προϋπολογισμό. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ προπολογισμό για να υποστηριχθεί η κοινή πολιτική. Έστω και αν μένει στάσιμο λοιπόν και δεν αρέσει αυτό ο αλλή, ε, υπάρχουν αρκετά ποσά, δεν έχει περικοπεί και πρέπει να δούμε και την εκτέλεση μέχρι τώρα στο παρελθόν Πρέπει εμείς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβουμε υπόψη την προηγούμε, τις προηγούμενες εκτελέσεις, τα προηγούμενα έτη δηλαδή, ε, για να κάνουμε τις προτάσεις μας αν πρόκειται να είναι διαφορετικές. Ο κύριος Στρεπίλαν θέλει να προσθέσει κάτι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. να θέλω να προσθέσω κάτι εντάχει. Πρώτον, ευχαριστώ τους συναδέλφους γιατί υποστήριξαν την πρότασή μου και δεν μπορώ παρά να συνεχίσω επί της ίδιας γραμμής. Συμφωνώ και εγώ με αυτά που ακούστηκαν. Πρέπει να καταγγείλουμε πραγματικά ε, και να αρνηθούμε αυτές τις προτάσεις της Κομισιόν. Ήταν πάντω χρήσιμα αυτά που μα είπε η Κομισιόν, γιατί είδαμε ότι η Κομισιόν ασπάζει τι γενικέ γραμμέ, το δικό μα προσανατολισμό και κρίνει τροποντινά ότι είναι χρήσιμο να συνεχίσουμε να έχουμε ένα τροποντινά σε επίπεδο χρηματοδότηση του προπολογισμό. Όμω προσπάθησε λιγάκι να παίξει με τους αριθμούς. Βεβαίως με τους αριθμούς δύσκολα παίζεις. Δεν μπορεί. Δύο συν δύο κάνουν τέσσερα. Δεν μπορεί να κάνουν ούτε πέντε ούτε τρία. Άρα θα πρέπει λοιπόν η Κομισιόν να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε σήμερα. Κάποιες γραμμές λοιπόν είναι πολύ σημαντικές, ιδίως για τους νέους ορίζοντες που ανοίγουν το 2013 για την Ελία θα δω με μεγάλη προσοχή ε, τις τροπολογίες και φυσικά δέχομαι ευχαρίστως την ε, συμβουλή της κυρίας Φράγκα να έχω τα μάτια μου ανοιχτά και να καιροφυλαχτώ βεβαίως επειδή πάντως υπάρχει ενιαία θέση των συναδέλφων επί του θέματος, θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε τι καλύτερε τροπολογίε τροπολογίες μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ριμπελίνη. Άρα λοιπόν η προθεσμία για τροπολογίες είναι 16 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα και να υπενθυμίσουμε επίση ότι και η η Επιτροπή μας και 40 ευρωβουλευτές μπορούν να υποβάλουν τροπολογίες επί των ε, αριθμητικών στοιχείων προπολογισμού στις 7 Σεπτεμβρίου και οι πολιτικές ομάδες έχουν μια άλλη προθεσμία 13 Σεπτεμβρίου. Άρα υπάρχει ακόμα δυνατότητα για την υποβολή τροπολογιών ώστε να σπηρεστούμε καλύτερον τον τρόπο τις θέσεις μας. Πάμε στο σημείο 13. Θέσπιση του προγράμματος πλαίσιο για την έρευνα και την κοινοτομία ορίζον 2020. Εισηγητής ο κύριος Τσουκαλάς Δυστυχώς δεν είναι πάρον ο κύριος Τσουκαλάς, αλλά θα τον υπερασπιστεί, αν θέλετε, θα παρουσιάσει ουσιαστικά την ε, γνωμοδότηση του κ. Καντέκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι ο συνάδελφός μας ε, Τσουκαλάς ε, είναι ασθενή και μου ζήτησε να τον αντικαταστήσω. Έμεινε στην Ελλάδα. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν το σχέδιο γνωμοδότησής του και θα συλλέξω και τα δικά σας σχόλια. Πρόκειται λοιπόν για το ε, πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία 2020-2014-2020. γνωμοδότηση της Επιτροπής μας στην καθήλυνα αρμόδια Επιτροπή Ήτρε. Μου έδωσε και το κείμενο, θα σας το διαβάσω με αιτήσια κατανάλωση γύρω στα 12 εκατομμύρια τόν σε λευτικά προϊόντα αξία σε περίπου 55 εκατομμύρια ευρώ. Επενθυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μία από τι πρωτοδοκτισμένε αγορέ που δεν μπορεί όμω να αποκριθεί επαρκώ στην εσωτερική κατανάλωση τη Ευρώπη, διότι γνωρίζετε ότι το 70% όσων καταναλώνουμε τα εισάγουμε. Η αλληλεξάρτηση μεταξύ θαλάσσιου περιβάλλοντο και Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί υψηλό επίπεδο έρευνα στον τομέα τη θάλασσα και τη ναυτιλία για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα και να να προστατεύσουμε καλύτερα τα θαλάσσια οικοσυστήματα και να αναπτύξουμε βιώσιμη ελεία που θα σέβεται το περιβάλλον, λαμβάνοντα υπόψη κοινωνικο-οικονομικέ ανάγκε των παράκτιων και νησιωτικών κοινοτήτων. Πάνω από το 90% τη θαλάσσια βιοπικιλότητας δεν έχει εξεταστεί. Και αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της θαλάσσιας και ε, ναυτικής έρευνας. Δεν υπάρχουν ε, επιστημονικά στοιχεία αξιόπιστα, άρα πολύ δύσκολα να υπάρξει υπεύθυνη διαχείριση των λευτικών αποθεμάτων. Και γι' αυτό με την γνωμοδότηση αυτή έχουμε στόχο να βελτιώσουμε την κατανόηση των αναγκών τη θαλάσσια και ναυτική έρευνα, λαμβάνοντα υπόψη ε, τι περιβαλλοντικέ, κοινωνικέ και οικονομικέ ανάγκε, στο βαθμό βέβαια του δυνατού, όπω το ίδιο κάνουμε και στη μεταρρύθμιση τη κοινή αλληλευτική πολιτική. Ε, πιο στενή συνεργασία μεταξύ των ρευτικών προγραμμάτων και των διαθροτικών ταμείων θα μπορέσουμε να επηρεάσουμε θετικά του τομεί τη αλληλεία ε, και έτσι θα μειωθεί η γραφειοκρατία με στοχευμένε δράσει σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Πιο στενέ σχέσει με την πολιτική συνοχή, περιφερειακή πολιτική και διαρθρωτικά ταμεία είναι κάτι που θα διευκολύνει και τη συμμετοχή των περιφερειών στη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και την προσπάθεια τη Ευρώπη να αντιμετωπίσει τι προκλήσει του σύγχρονου κόσμου. Ο αποτελεσματικός συντονισμός, η συμπληρωματικότητα των δράσεων στο πλαίσιο του οριζόντα 2020 μαζί με χρηματοοικονομικές, μάλλον με δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο για την Αλία και τη Θάλασσα, είναι σημαντικά στοιχεία για να μην έχουμε ε, αλληλεπικαλύψεις. Η στήριξη της θαλάσσιας επιστήμης, ε, δυνατότητες κινητικότητας για τους ερευνητές, Ευχαριστώ πολύ. Η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η παρακίνηση συμμετοχή στι τελευταίε δραστηριότητε μπορούν να κάνουν τι ευρωπαϊκέ περιφέρειε που εξαρτώνται από την αλληλεία πολύ ανταγωνιστικά σε ευρωπαϊκό και διεθνέ επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό, στόχο τη θαλάσσια έρευνα θα πρέπει να είναι παραγωγικέ θάλασσε και ωκεανοί για τη βιώσιμη ανάπτυξη, για την αλληλεία, για την δατοκαλλιέργεια και να υπάρξει κατάλληλη χρηματοδότηση. Γιατί αν δεν επαρκεί χρηματοδότηση, αφενό το μεγάλο δυναμικό του, της τεχνολογίας και στις θαλάσσιες θα παραμείνει ανεκμετάλλευτο και η, ε, θα υπάρχει υπερακμετάλλευση στις θαλάσσιες έρευνα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε να δημιουργήσουμε ειδική γραμμή στον προπολογισμό για εγκάρσιες δράσεις για να αναπτύξουμε συνέργειες μεταξύ θαλάσσιων ναυτικών θεμάτων για να έχουμε την καλύτερη αναγνώριση των μακροχρόνιων προκλήσεων και τον κατάλληλο προπολογισμό για να τα αντιμετωπίζω. Σας ευχαριστώ για την σχετική σας προσοχή. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Καντέκ ε, Τσουκαλά, λέει ο πρόεδρος. Θέλει το λόγο κάποιος από τους συναδέλφους, όχι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, θέλετε. Έχετε το λόγο λοιπόν. Thank you very much, Ευχαριστώ πρόεδρε. Να πω απλά ότι Εκτιμούμε ιδιαίτερα τη δυνατότητα να κάνουμε κάποια σχόλια για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης και τις σχετικές τροπολογίες που προτείνεται. Πρώτα απ' όλα να πω κάτι εν είδη υπενθύμησης. Είναι ένα θέμα που έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν. Πρέπει να σε υπενθυμίσω ότι το νέο πρόγραμμα Horizon 2020 έχει σχεδιαστεί ώστε να αυξήσει τη γνώση σχετικά με τη διάδραση ανάμεσα στην αλληλεία και το θαλάσσιο περιβάλλον, και θα λάβουμε υπόψη τις κοινωνικο-οικονομικές πτυχές σε ό,τι αφορά τις νησιωτικές και παράκτιες κοινότητες. Ε, πιστεύουμε ότι θα έχουμε πιο αξιόπιστα στοιχεία για να στηρίξουμε τη βιώσιμη διαχείριση της αλληλείας και πέρα από αυτά προτείνουμε και μια αύξηση του προπολογισμού σε σχέση με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, συνολικό ποσό για αυτή την πρόκληση είναι το υπερδιπλάσιο σε σχέση με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Και βεβαίως είμαστε σε θέση να δούμε και εγκάρσια ζητήματα με πολυτομιακή έρευνα και αυτό πιο αποτελεσματικά από ό,τι στο παρελθόν, χρησιμοποιώντας βεβαίως και την κτηθή σε εμπειρία. Έχουμε μια πολύ ισχυρή εντολή ώστε η καινοτομία να είναι συνιστόσα όλων αυτών των πρωτοβουλειών και να συμμετάσχει η βιομηχανία και ιδίω μικρομεσαίε επιχειρήσει και να θέσουμε περισσότερο ε, στην ενίσχυση της εφαρμοσμένης έρευνας και άλλες μορφές καινοτομίας όπως προαγωγή των αποτελεσμάτων, διάδοσή τους κτλ. Ε, σε ό,τι αφορά κείμενα και μελλοντικά ερευνητικά προγράμματα και ελπίζουμε να υπάρχουν μεγαλύτερες συνέργειες με τα θεωρητικά ταμεία και ιδίως με το νέο ταμείο για την αλληλεία και τη θάλασσα και επίσης με τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΜΑΡΕ και τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ έρευνα και ανάπτυξη θα υπάρξει κατάλληλη αλληλοκάλυψη, αλληλοσυμπλήρωση για να έχουμε αυτές τις απαραίτητες συνέργειες και βεβαίως τα ερευνητικά προγράμματα, ξέρετε γενικά. Έχουμε ένα καλό ιστορικό καθώς προσελκύουμε, μάλλον ενθαρρύνουμε με αυτόν τον τρόπο την κινητικότητα των ερευνητών και έχουμε καλύτερη ε, εκπαίδευση για τον ολοκλάδο. Και λίγα σύντομα σχόλια σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες, σε γενικές γραμμές. Ε, είμαστε σε θέση να χαιρετήσουμε την έμφαση που δίνεται στην βιοτεχνολογία σε θέματα ε, θαλάσσιου περιβάλλοντος, ετοκαλλιέργειας και αλίας. Το χαιρετίζουμε αυτό, αλλά να πω ότι έχουμε και κάποιες ε, ενδυνάμει επιφυλάξεις για αυτές τις τροπολογίες. Δεν ξέρω αν θέλετε να διατρέξω τώρα αυτές τις επιφυλάξεις. Αλλά κάποιες αφορούν π.χ. τον τίτλο. Η αλλαγή του τίτλου μπορεί να είναι πολύ περιοριστική, γιατί εμείς θέλουμε να καλύψουμε και την ε, θαλάσσια βιοτεχνολογία. Όταν περιορίζεται λοιπόν τον τίτλο στην αλία και την για να μην με περιορίζει το πεδίο εφαρμογή. Επίση, σε ό,τι αφορά τα επίπεδα χρηματοδότησης και να είναι αναλογικά με το δυναμικό των διαφόρων ε, πηγών τροφίμων. Ξέρετε, δεν καλύπτουμε εδώ μόνο τα τρόφιμα, αλλά και ε, πολλά άλλα. Και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να το συνδέσουμε λοιπόν και με του άλλου τομεί που καλύπτουμε. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει ναι, να προβούμε σε αυξήσει χρηματοδότηση σε πραγματικού ε, όρου. Συλλογή δεδομένων. Αυτό δεν είναι κομμάτι των ερευνητικών δραστηριοτήτων. Αυτό είναι καλύτερο να χρηματοδοτηθεί μέσω του Ταμείου Ελεία. Και όπω είπαμε και νωρίτερα, προτιθέμεθα να διερευνήσουμε τρόπου ενίσχυση των εγκάρσεων πτυχών όχι δηλαδή μόνο στα πλαίσια των επιστημών, των θετικών επιστημών, των επιστημών της ζωής, αλλά και να δούμε και το πώς συνδέονται και με τα περιβαλλοντικά ζητήματα, με τις μεταφορές κτλ. Έχουμε και μακρά εμπειρία ε, και με το project «Η ωκεανή του αύριο» και να σας πω ότι χθες δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 55 εκατομμύρια συνολικά για τα εγκάρσια ζητήματα. Έχουμε λοιπόν μια κάποια εμπειρία πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε και η γενική εντύπωση είναι ότι θα επιτύχουμε πολύ περισσότερο στο μέλλον, στα επόμενα βήματα. Γνωρίζετε επίσης ότι η πρόταση της Προεδρίας δεν καλύπτει στο βασικό κείμενο, στη βασική πρόταση και αυτές τις εγκάρσεις πτυχές, αλλά πλέον καλύπτονται αυτές τις προκλήσεις με τις τροποποιήσεις που έγιναν. Πιστεύω λοιπόν ότι έχουμε πλέον τον κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να είμαστε σίγουροι ότι αυτά θα γίνουν πράξη στο μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Λόβεν, ζήτησε το λόγο, παρακαλώ. Ναι, μόνο πολύ σύντομα. Ήθελα να πω ότι θα είχα κάποια σχόλια ή ερώτηση, ίσως προς τον κύριο Τσουκαλά μάλλον, για τις ε, τροπολογίες του. Εκεί που αλλάζει τους όρους στα θαλάσσια έρευνα. Το βλέπω στα σουηδικά, σας το διαβάζω λοιπόν στα σουηδικά. οι ωκεανοί θα πρέπει να ε, ξεδαστούν μέσα από τις, ε, ιδέα της βιώσιμης εκμετάλλευσης κτλ. Εδώ βλέπω ότι σαν να περιορίζεστε. Ζητώ συγγνώμη γιατί δεν λαμβάνω την μετάφραση στα ισπανικά. Ska jag eh, Τώρα είμαστε εντάξει, μπορώ να ξαναμιλήσω. Καλώς, λοιπόν, στην υπαριθμόν 4 τροπολογία. Ο κύριος Τσουκαλάς βλέπω να έχει αλλάξει τον όρο θαλάσσιοι πόροι με τον όρο ε, παραγωγική αλληλεία, που σημαίνει κάτι τελείως διαφορετικό. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τι είχε υπόψη του, τι πρόθεση είχε με την αλληλεγγύη αυτή του όρου. Ευχαριστώ. Καλώς, η κυρία Φράγαφη, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στην Κομισιόν. Δεν είμαι σίγουρη ότι κατάλαβα πολύ καλά. Ή έχω κουραστεί. Τι ήθελε να μας πει η Κομισιόν με την ομιλία αυτή που έκανε ο κύριος αυτός για την εφαρμοσμένη έρευνα στην Αλία ότι δεν εμπίπτει στο έγγραφο το καταπληκτικό αυτό ή εγώ υποσύγχυση ή δεν κατάλαβα. Γιατί αν έτσι έχουν τα πράγματα τότε δεν χρησιμεύει τίποτε αυτό το πρόγραμμα πλαίσιο. Κρατήστε το εκεί που το έχετε. Δεν συμφέρει την αλία σε τίποτε. Δεν, τη χρέω, δεν το χρειαζόμαστε. Κυρία Ρόντου, έχει τώρα το λόγο. Ναι, το ίδιο θα έλεγα κι εγώ. Γιατί πρέπει η έρευνα να περάσει μέσα από το πολιτισμο δημοσιονομικό πλαίσιο. Έχουμε το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα για να μην μπει εκεί η έρευνα για την αλία. Τόσε πολλά είναι τα κενά που έχουμε ω προς τις γνώσεις, τις λεγόμενες γνώσεις. Νομίζω ότι θα βοηθούσε πάρα πολύ να τι βελτιώσουμε. Ευχαριστώ η επιτροπή παρακαλώ. Σα ευχαριστώ για την ευκαιρία να δώσω μια διόρθωση προ μια παρεξήγηση εφαρμοσμένη αέρια, είπα ότι είναι ένας από τους τομείς που μπορεί να καλυφθεί και είπα ότι θα καλύψουμε περισσότερο ακόμα στο επερχόμενο χρηματοδοτικό μέσο ε, σύνολο προτάσεων για το 2020. Υπάρχει μάλιστα μια συζήτηση να συμπεριληφθεί ολόκληρο το φάσμα από την βασική έρευνα μέσα στην εφαρμοσμένη ε, αλλά και την εμπορία με πολύ, πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα Όπω φαίνεται. Άρα μπορούμε στον ορίζοντα 2020 να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση για την έρευνα αυτή. Ο συσχετισμό με το πολιετέ μεσονομικό πλαίσιο έχει να κάνει με την ανάγκη για συμβατότητα. Και βέβαια τη λήψη υπόψη των αποτελεσμάτων τη έρευνα όπου χρειάζεται. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Καντέκ για να κλείσουμε. Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Θα απαντήσω στην Ιζαμπέλα. Θα ήθελα μάλλον να της πω ότι δεν μπορώ να τη απαντήσω δεν έχω απάντηση για την ερώτησή σα, Θα διαβιβάσω στον κύριο Τσουκαλά την ερώτηση για την ε, τροπολογία παριθμό 4. Πάντω συμφωνώ και με του άλλου συναδέλφου ότι αυτή η γνωμοδότηση που τροποποίησε ο εισηγητή είναι πολύ αξιόλογη εν γέννη. Θα προσδοριστεί φαντάζομαι η ημερομηνία για κατάθεση τροπολογιών. Πάντω, σα διαβεβαιώνω ότι θα ενημερώσουμε τον άλλου κύριο Τσουκαλά. Πράγματι, ο πρόεδρο σα ανακοινώσει την προθεσμία κατάσταση απολογιών 12 το μεσημέρι στι 16 Ιουλίου. Τότε λίγη προθεσμία. Γιορτάζουν οι Κάρμεν Στην Ισπανία. Μα δεν μπορείτε, λέει κυρία Φράγκα. Ε, σκοτώμαστε στη δουλειά κάθε μέρα. Δεν, δεν προλαβαίνουμε. Πρόεδρος, ναι, και όλα... Ε, έχεις και τη γιορτή σου γίνεται. Ναι, ε, υπάρχει ανάγκη, είναι κατεπήγον. Αλλιώ δεν το καταλαβαίνω. Μας μένουν δύο μέρε δουλειά ε, πριν τι διακοπέ και πρέπει να τα κάνουμε όλα μέσα σε αυτέ τι δύο μέρε. Να το πάμε τέλειου Ιουλίου. Προβλέπετε να ψηφιστεί στην Επιτροπή μας το Σεπτέμβρη και στην Ήτρε 9 ε, Οκτωβρίου. Τι να κάνω, το βάλω 18. Ακούστε, τι μπορούμε να κάνουμε. Καταρχήν, αν συμφωνείτε, όσο μπορούμε θα καθυστερήσουμε την προθεσμία μέσα στον Ιούλιο Επισήμω θα σα ανακοινώσουμε το πότε θα λύγει η προθεσμία. Θα ενημερώσουμε φυσικά και τον εισηγητή. Συμφωνείτε? Ωραία. Και περνάμε στο επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξη, τελευταίο για σήμερα, το σημείο 14. Αλληλευτικέ δυνατότητε και γραμματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη Συμφωνία Αλληλευτική Σύμπραξη μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Κοινότητα αφενό και τη κυβέρνηση τη Δανία και τη τοπική κυβέρνηση τη Γρυλανδία. Αφετέρου. Προβλέπετε να στείλει επίσημη αίτηση έγκριση ε, εντό του Ιουλίου το Συμβούλιο, ενώ από πλευράς Επιτροπής τώρα θα ακούσουμε την παρουσίαση που όπως θυμάστε δεν έγινε την προηγούμενη φορά που συνεδριάσαμε. Δίνω λοιπόν ευθύς αμέσως το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, το είναι αυτό πρωτόκολλο που μονογράφηκε το προηγούμενο Φεβρουάριο θα το περιγράψω ως προς τα αδρά του σημεία υπογραμμίζοντας τις βασικές διαφορές ε, ταυτόχρονα μεταξύ αυτού του πρωτοκόλλου και του πρωτοκόλλου με τη Γρυλανδία και των λοιπόν αλλιευτικών συμφωνιών πρωτοκόλλων που έχουμε ε, συνάψει με χώρες ΑΚΕ. Η πρώτη διαφορά είναι Ε, διαπραγματευόμαστε κάθε χρόνο το επίπεδο της αλληλευτικής δυνατότητας με βάση επιστημονική, ετήσια επιστημονική έκθεση που παρουσιάζει η CIOM, e τα e στα αγγλικά, για την αλληλευτική ε, προσπάθεια και τις δυνατότητες της αλληλευτικές σε κάθε είδος. Αυτή είναι η πρώτη διαφορά. Δεύτερη διαφορά, ιδιαίτερη, η διότι ένα μέρος των αλληλευτικών δυνατοτήτων που προβλέπει αυτή, αυτό το πρωτόκολλο καλύπτεται από τη διμερή συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, Βασιλείου της Νορβηγίας και αφορά μια ανταλλαγή πληροφοριών αμοιβαία έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα της ε, ε, την αλληλευτική δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτά τα αυτές τις περιόδους. Και άλλη μια τρίτη ιδιαιτερότητα είναι το πρωτόκολλο με τη Γερλανδία εντάσσεται μέσα σε ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο που καλύπτει την, ε, το συνολικό πλαίσιο εταιρική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Γερμανία. Πρόκειται για ένα πρωτόκολλο δηλαδή το οποίο αποτελεί έναν από τους δύο άξονες αυτής της ε, διμεριούς αλληλευτικής ε, συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιρλανδίας. Αυτό είναι το πρώτο πρωτόκολλο. Τώρα το νέο πρωτόκολλο που μονογράφηκε το Φεβρουάριο έχει περίοδο τριών ετών, έχει διάρκεια τριών ετών. Τα κράτη που κυρίως έχουν ε, αλληλευτικές δυνατότητες είναι η Δανία, η Εστονία, η Λετωνία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία. Έχουμε δηλαδή ένα αρκετά ευρύ φάσμα μεγάλο αριθμό κρατών που μπορούν να υποφεληθούν από αυτές τις ε, αλληλευτικές δυνατότητες, πράγμα το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την γενική και θετική αξιολόγηση πρέπει να γίνει για το πρωτοκόλλο. Όσον αφορά την αλληλευτική δυνατότητα, έχουμε πρόσβαση από τις διαπραγματεύσει μας σε διάφορα είδη ανάλογα και βασιζόμενη στην πτυχή της διάρκειας. Τα της διάρκειας εκμετάλλευσης, δηλαδή τα είδη στα οποία υπήρξε υπεραλίευση, υπερεκμετάλλευση, ε, βγήκαν από τη συμφωνία προκειμένου να διασφαλιστεί αυτή η βιωσιμότητα η διάρκεια στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης όπως γνωρίζετε, την οποία, στην οποία, έγκριση προχωρούμε, αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία από την υπηρεσία μας αλλά και από, τον Επίτροπο, από την Επίτροπο στην ιδέα αυτή της διάρκειας. Άρα η, τα αποθέματα είναι ο γάδος με 200.000 τόνους στο 2.000 ε, τόνους, ο Σεβαστός 3.000 τόνους, Μερσάλ 2.000 τόνους, ο το φλετάν του Ατλαντικού, η Βόρεια Γαρίδα με 1.900 τόνους, ο... το Καλκάνι του Ατλαντικού με 450.000 τόνους και ο Γραναδιάρος με 200 τόνους. Ε, θα ήθελα λοιπόν να προσθέσω μια ε, διευκρίνηση ότι οι ποσοστώσεις αυτές είναι ενδεικτικές και κάθε χρόνο αφορούν, ε, ε, υπάγονται μάλλον σε μια επανεξέταση από τη Μεκτή Επιτροπή και πάλι σε βάση, με βάση την επιστημονική έκθεση της ΕΜ για να μην υπάρξει υπεραλίευση, υπερεκμετάλλευση, πράγμα το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία πρέπει να υπογραμμίσω για το μέλλον των αποθεμάτων. Όσον αφορά τα οικονομικά ζητήματα, πολύ σημαντικό επίσης το ετήσιο κόστος αυτής της συμφωνίας ανέρχεται σε 17,8 εκατομμύρια με την εξής κατανομή 15,1 για την πρόσβαση και 2,7 εκατομμύρια το χρόνο για την στήριξη στον τομέα. Μέσα στα 15,1 εκατομμύρια υπάρχει ένα αποθεματικό της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για να καλυφθούν ενδεχόμενες νέες αλληλευτικές δυνατότητες πέραν των ποσοστώσεων που προσδιορίστηκαν και εφόσον η κατάσταση των πόρων το επιτρέπει. Για την τομεακή στήριξη, όπως εξήγησα, έχουμε προβλέψει μια ετήσια πρικοδότηση τάξης των 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε, όπως ήθιστε τα τελευταία δύο χρόνια, συμπεριλάβει νέα ρήτρα στο πρωτοκόλλο αυτό, μια ρήτρα δηλαδή η οποία αναφέρεται στο σεβασμό των ανθρωπινών δικαιωμάτων και σε περίπτωση παραβία των ανθρωπινών δικαιωμάτων, άρσης του πρωτοκόλλου και επίση έχουμε και την ρήτρα ερεσιμότητα όσον αφορά το, το, τη στήριξη στον τομέα. Εάν δεν λειτουργεί δηλαδή καλά, εάν δεν λειτουργεί η στήριξη, τότε πάλι ε, επέρχεται άρση του πρωτοκόλου ε, ε, μια νέα διάταξη, μια νέα ρήτρα την οποία έχουμε μπορέσει να εισαγάγουμε στο πρωτόκολλο με τους εταίρους ε, ΑΚΕ τα τελευταία δύο χρόνια, μια καινοτομία η οποία προβλέπεται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης και της ανακοινώσή μας άλλωστε. Ε, πρέπει επίσης να σας πω ότι το νέο πρωτόκολλο είναι αρκετά εξισορροπημένο για τις δύο πλευρές εγγράφεται μέσα στην παράδοση συνεργασίας, στη θετική παράδοση συνεργασίας που έχουμε με τις αρχές της Βιλανδίας, οι οποίες άλλωστε διατύπωσαν και τη βούλησή τους για, ένα νέο πρωτόκολλο, για συνεργασία περαιτέρω μαζί μας, για τη βελτίωση και την εξασφάλιση των αποθεμάτων και την σωστή αλληλεία. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, με στη σας. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε τον λόγο στον κύριο Κρίστερσεν τώρα, τον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την Κομισιόν για αυτή την παρουσίαση. Ήδη απαντήσετε σε κάποια από τα ερωτήματά μου, οπότε θα είμαι και εγώ σύντομος με δύο επιπλέον ερωτήματα. Σε γενικές γραμμές ε, είσαστε θετικοί στα θέματα έρευνας ε, παρακολούθησης και τα προγράμματα εκπαίδευσης. Αυτό πιστεύω ε, αφορά την Αγριλανδία και είναι κοινή θέση όλων. Όμως αυτό δεν έχει αντίστοιχα θετικό αντίκτυπο στην ε, δημιουργία θέσεων εργασίας τοπικά. Τι γίνεται λοιπόν στα πλαίσια του νέου πρωτοκόλλου για να υπάρξει βελτίωση από αυτού σε ό,τι αφορά τώρα την χρηματοδότηση. Εξηγήστε μας γιατί το ετήσιο ποσό που καταβάλλεται για την πρόσβαση στην ΑΟΣ στη Γρυλανδία σε ό,τι αφορά ευρωπαϊκούς στόλους αυξήθηκε κατά 1 εκατομμύριο ευρώ όταν οι λευτικές ευκαιρίες έχουν μειωθεί. Ευχαριστώ πολύ. Okay. Ich kann mich ganz kurz fassen. Μπορώ να Είμαι πολύ σύντομο. Βλέπω με ικανοποίηση ότι έχουμε μια, αιτιολο... λεπτομερή αξιολόγηση του πρωτοκόλλου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νέο στοιχείο λοιπόν που βελτιώνει την ασφάλεια. Όπω επισημαίνει και ο εισηγητή κ. Κρίστινσεν έχουμε σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα για την πρόσβαση στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Γρυλανδίας με 6.000 τόνους συνολικά λιγότερο ψάρι Άρα πιστεύω θα πρέπει να δώσουμε έμφαση ακριβώς στο θέμα των υποδομών. Και δεν θέλω να ρωτήσω τι υπάρχει από πλευράς Φιλανδίας, ε, τι είδους ε, υποδομές υπάρχουν για την ε, κατεργασία αλλά και την εκφόρτωση στους χώρους εκφόρτωσης. Επίσης, ερώτηση έχω για το Βασίλειο της Νορβηγίας. Είπατε ότι έχετε εντατικέ διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις για την κοινή αλίευση στα ύδατα αυτά. Όλοι, όλοι όμως γνωρίζουμε ότι και η ρωσική ε, ομοσπονδία ενδιαφέρεται και έχει πολύ μεγάλη δραστηριότητα στην περιοχή αυτή με χίλιους τόνους γάδου. που εν τέλει συνεπάγονται πολύ σημαντικό ανταγωνισμό για τους αλληλείς μας και αποτέλεσμα να έχουν πέσει σημαντικά τα, αποτελ... τα... αποθέματα του γάδου στα ύδατα αυτά. Ερωτώ λοιπόν τι μπορείτε να κάνετε γι' αυτό. Κύρια Φράγα παρακαλώ έχετε το λόγο. Ναι, να κάνω και εγώ μερικές ερωτήσεις στην Κομισιόν. σε ό,τι αφορά τον, ε, ε, το καβούρι. Ναι, ναι. δεν βλέπω να υπάρχει κάποια τροποποίηση στην πρότασή σας. Ε. Βλέπω το ίδιο όπως παλαιότερα. Και υπάρχει πρόβλημα όμως με αυτό το αλίευμα. Και όσοι κάνουν αλίευση αυτού του καβουριού δεν έχουν ποτέ πρόσβαση στην Γρυλανδία. Να δούμε πώς μπορούμε να το συντονίσουμε αυτό εσωτερικά. Δεύτερο, Ξέρετε, το σύστημα αδειών, επιμερισμού των αδειών, έχει τύχει πολλών επικρίσεων, γιατί είναι πάρα πολύ άκαμπτο. Διότι αν τελικά καταλήγει σε μια μεγαλύτερη ποσότητα, να λαμβάνει μεγαλύτερη ποσόστοση ακόμη και δεν τη χρειάζεται, ουσιαστικά πρέπει να την πληρώσει. Πρέπει να γίνουν κάποιες διορθώσεις. Και επίση πείτε μας κάτι άλλο. Στο προηγούμενο πρωτόκολλο, το ποσοστό χρηματοδότησης τη Ένωση ήταν 85% σε σχέση με το 15% των ε, πλειοκτητών. Ε, μένουμε σε αυτό το ποσοστό ή όχι. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές για τις ερωτήσεις που μου υπέβαλαν. Τι σημείωσα νομίζω λίγο πολύ και θα προσπαθήσω να απαντήσω συνολικά. Ναι, υπάρχει διαφάνεια και έγινε εξωτερική αξιολόγηση όπου και μας ε, επικρίνουν κατά κάποιο τρόπο για το ότι δεν δημιουργήθηκαν θέσεις εργασίας με την πτώμακη προσέγγιση. Κάτι που μπορεί να ισχύει, αλλά ξέρετε ότι ουσιαστικά πρόκειται ε, για μια συνεννόηση μεταξύ της Γρυλανδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Γρυλανδία είναι αυτή η οποία πρέπει να καθορίσει τους άξονες προτεραιότητας για να υπάρξει σε αυτούς η τομεακή στήριξη. Δική τους ήταν η απόφαση να ενθαρρύνουν το θέμα της διακυβέρνησης αλίας, που είναι πολύ σημαντικό και επίκαιρο πρόβλημα, όπως επίσης και τον έλεγχο και την εφαρμογή, αλλά και τον τομέα Τη έρευνα και των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων. Τρει είναι οι βασικοί λοιπόν αυτοί οι άξονες που σα προανέφερα που χρησιμοποιήθηκαν για την διοχέτευση του ε, προπολογισμού μέσω τη τομεακή στήριξη. Δυστυχώ δεν υπήρχε τίποτα για τη δημιουργία θέσεων ε, απασχόληση, αλλά νομίζω ότι αυτά τα τρία κέντρα, αν θέλετε, ενδιαφέροντος αξίζουν θετική αξιολόγηση ό,τι έφερε τη χρήση του. Ω προ την. Ε, μάλλον ως προς το κόστος πρόσβασης ε, υπήρξαν ε, στην αλληλευτική δυνατότητα μειώσεις. 6.000 τόν ήταν η μείωση συνολικά πράγματι. Αλλά βάσει αναφοράς είναι η τιμή της αγοράς από τότε. Για κάποια ε, αλλιεύματα αυξήθηκε το κόστος, το αγοραίο κόστος. Και γι' αυτό χρειάστηκε να έλθουμε σε διαπραγματεύσεις με τους Γρυλανδούς. Και δεν σας κρύβω ότι οι οικονομικές απαιτήσει ήταν τεράστιες σε σχέση με τα νούμερα. Τα τελικά, τα οποία καταφέραμε να διαπραγματευτούμε. Κάναμε λοιπόν ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Εγώ ηγήθηκα των διαπραγματεύσεων, θέλω να σας πω. Και το οικονομικό αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό. Γιατί μειώθηκαν οι λιευτικές ε, ε, προσπάθειες. Δεν το επέτρεπε το μέγεθος του αλλιεύματος, ε, των αποθεωμάτων. μάλλον. Είδαμε, κάποιοι δυσαρεστήθηκαν όταν είδαν θα μειώσουμε την αλληλευτική προσπάθεια, αλλά το κάναμε βασιζόμενοι σε επιστημονικά στοιχεία και γιατί δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε να έχουμε ποσοστά οι ποσοστώσεις αλίευσης τόσο υψηλά, ενώ επιστημονικά αυτό δεν ήταν επιτρεπτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κάβουρα της Ακτικής, ε, πράγματι δεν το είχαμε χρησιμοποιήσει, αλλά υπήρξε έντονο αίτημα από την Ισπανία για να διατηρηθεί το αλίευμα, η αλίευση αυτού του είδους και διατηρήθηκε πράγματι και ελπίζουμε να είναι τέτοιοι όροι για την χωρίς αυτής της άδεια και άσκηση αυτής της αληφτής δραστηριότητας που θα ικανοποιεί τους στόλους που έθεσαν αυτό το αίτημα. Σε ό,τι αφορά τώρα τον γάδο και τις σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία, εδώ συζητούμε τη Γρυλανδία, δεν συζητούμε τη Ρωσία. Βέβαια, γνωρίζουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ έντονος ανταγωνισμός με την αλληλευτική προσπάθεια των ρωσικών πλοίων. Ανταγωνισμός που δυστυχώς μεταφράζεται σε μείωση της τιμής αγοράς του γάδου. Αλλά επαναλαμβάνω και το είπα και στην εισαγωγή μου. Αυτή η συμφωνία με την Ιρλανδία είναι πολύ σημαντική γιατί μέρος αυτών των λεφτικών δυνατοτήτων είναι σαν αντιστάθμισμα, σαν αντιπαροχή ε, για να έχουμε και στα νορβηγικά ύδατα ε, αλληλευτικέ δυνατότητε. Αυτή η συμφωνία συνάπτεται σε τέτοια βάση με την Ιρλανδία είναι απαραίτητη. Και επαναλαμβάνω, είναι και μία από τις σπάνιες συμφωνίες που με τη δυνατότητα σε πολλές χώρες να μπορούν να αλλιεύουν στα ύδατα της Ιρλανδίας πολλές φορές ε, εδώ στο Κοινοβούλιο κατηγορήθηκε η Κομισιόν, κατηγορηθήκαμε ότι συνάπτουμε συμφωνίε περιορίζονταν σε 2, 3, 4 δικαιούχε χώρου. Εδώ βλέπετε πάνω από 10 είναι οι χώρε δικαιούχοι. Άρα έχει διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογή και εκμετάλλευση αυτών των συμφωνιών. Δεν ξέρω αν μου διέφυγε κάποια ερώτηση. Θα, θα μου το επιθυμήσετε φαντάζομαι. Πρόεδρο, θέλει να προσθέσει κάτι ο κ. Κρίστενσεν. Ουδέν. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω όλους, διότι με αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε τη σημερινή μερίσια διάταξη και μάλιστα ακριβώς την ώρα μας. Να ευχαριστήσω όλα τα μέλη και τους διερμηνείς. Αύριο θα ξεκινήσουμε στις 9 και μάλιστα σε 9 ακριβώς. Έχουμε συνεδρία των συντονιστών για μισή μόνο ώρα. Και πριν ολοκληρώσουμε, σε σχέση με το προηγούμενο σημείο που είπα κάτι για την ε, προθεσμία. Λοιπόν, λίγη προθεσμία 23 Ιουλίου. Σας δίνουμε άλλη μια εβδομάδα δηλαδή, κυρία Φράγκα. Ναι, κύριε Πρόεδρε, επειδή αύριο θα έχετε τη συνεδρίαση των συντονιστών που θα είναι τελευταία πριν τις ε, θερινές διακοπές και επειδή στην τελευταία ολομέλεια, όπως θα θυμάστε και εσείς, μετά την ερώτηση για την κατάσταση με τη σήμαση Σάιτες, οπότε είχε και ζητηθεί παρουσία της Επιτρόπου Δαμανάκη και του Επιτρόπου Περιβάλλοντος που δεν ξέρω το όνομά του. Και επειδή τελικά, προς μεγάλη μας χαρά, ε, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος όταν άρχισε να μιλήσει η πρώτη, όταν άρχισε να μιλήσει η πρώτη που ήμουν εγώ από την ε, πλειοψηφική ομάδα, ε, σηκώθηκε και έφυγε από την αίθουσα. Πείτε το αύριο στου συντονιστέ και κλεισμένο των θερών δεν ξέρω εγώ πώ θα αποφασίσω ότι είναι το πλέον σκόπιμο και οι δύο επιτρόποι να έρθουν στην Επιτροπή μας και να μας εξηγήσουν τι γίνεται με αυτό το θέμα. Και οι δύο όμως, έτσι, ώστε να είναι ο ένας απέναντι από τον άλλο και να μας πούν τις απόψει τους και οι δύο. Είναι σοβαρότατο, δεν πηγαίνει καλά η κατάσταση, το είπα και τι προάλλε, οι ε, εθνικές αλληλευτικές διοικήσει ε, δεν ε, είχαν ενημερωθεί, το γνωρίζω γιατί στη χώρα μου δεν είχαν ενημερωθεί τους το έκρατσαν μυστικό και είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα. Και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα. Ζητώ λοιπόν να παρευρεθούν ε, οι δύο αυτοί οι επίτροποι που για πολλούς και διαφόρους λόγους που δεν με ενδιαφέρουν διόλου δεν ήταν το εστόλος παρόντες στην Ολομέλη σε αυτή τη συζήτηση. Είναι σοβαρό αυτό γιατί το θέμα είναι επίσης σοβαρό. Πρόεδρος, ναι πράγματι θα στείλαμε την επιστολή και τους είχαμε προσκαλέσει. Αλλά επειδή δεν ε, ανταποκρίθηκαν, θα κάνουμε ένα βήμα παραπάνω και θα τους ζητήσουμε πλέον να είναι, θα τους το απαιτήσουμε. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε τα υπόλοιπα αύριο.